Good morning. I ask everybody if you can sit in order that we... Παρακαλώ καθίστε για να μπορέσουμε να αρχίσουμε με την ακρόασή μας. Good morning, everybody. My name. Καλή σας μέρα. Ονομάζομαι Ινές Ζούμπερ και είμαι αντιπρόεδρος της Επιτροπής Απασχόλησης εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα μιλήσω όμως πορτογαλικά που είναι η μητρική μου γλώσσα. Καλημέρα σε όλους σας λοιπόν. Καλώς ήρθατε σε αυτό το κοινό σεμινάριο στην Ακρόαση που διοργανώνεται από την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Θέλουμε <clears throat> τις, ε, τα, τέσσερα, τις τα τέσσερα όργανα που εργάζονται σε αυτόν τον τομέα να συνεργαστούμε μαζί τους για να συζητήσουμε το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Πρότυπο ως θεμελιώδες στοιχείο για την ανταγωνιστικότητα στην, της Ευρώπης. Με μεγάλη χαρά λοιπόν σήμερα υποδεχόμαστε σε αυτό το σεμινάριο έχουμε ήδη διοργανώσει σεμινάρια <clears throat> με διαφορετική βέβαια μορφή και σύνθεση και είχαμε και τη διοργάνωση ε, εδώ και κάποιο χρόνο προηγούμενα του τελευταίου τον Ιούνιο 2011. Με αυτή την αφορμή κυρίως συζητήσαμε τα θέματα τα οποία συσχετίζονται με την απασχόληση των νέων, την εργασία και απασχόληση των νέων. Και αντιμετωπίζουμε τα θέματα της εκπαίδευσης και σε σύνδεση με τη θέση απασχόλησης πάντα για τους νέους και για να συζητηθούν επίσης και τα θέματα τα οποία συσχετίζονται με την ανάγκη, την αναγκαιότητα να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης για τους νέους. Κυρίως στο πλαίσιο <clears throat> της αντιμετώπισης του φαινομένου ΝΕΠ, δηλαδή των νέων που δεν βρίσκονται ούτε σε εκπαίδευση, ούτε σε κατάρτιση, ούτε έχουν και θέση εργασίας, θέση απασχόλησης. Και μέσα σε αυτή τη συζήτηση αυτό το οποίο τονίστηκε ήταν η συμπληρωματική εργασία που μπορούν να αναπτύξουν τα διάφορα όργανα όσον αφορά την κοινωνική πολιτική και την απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η συζήτηση θέλει να αναζωογονήσει και να αναδημιουργήσει το προηγούμενο πνεύμα των προηγούμενων συζητήσεων και σεμινάριων συμπληρώνοντας έτσι το έργο και με τις συνέργειες που μπορούν να δημιουργηθούν μεταξύ των τεσσάρων αυτών οργάνων ΣΕΝΤΕΦΟΠ, ETF, OSA και Eurofound και σήμερα συζητάμε ακριβώς το θέμα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Πρότυπου. Θέλω ευθύ εξ αρχής να καλωσορίσω λοιπόν <clears throat> ε, Υπουργέ Βαλερή Ατάρ τον Πρωθυπουργό και Υπουργό Οικονομικών στην ε, Δημοκρατία της ε, Μολδαβίας που θα είναι και ένας από τους συμμετέχοντες ε, στο πάνελ που θα αναπτύξουν τα θέματα αυτής της συζήτησης. Επίσης, να καλωσορίσω τους επικεφαλείς των τεσσάρων αυτών οργάνων. Κρίστιαν Λέτμαϊερ από το ΣΕΝΤΕΦΟΠ, Χουάν Μενέντες Βαντές από το Eurofound, Κρίστα Σέντλατσεκ από την και Madlen Serban από το ETF, European Training Foundation. Θα ήθελα επίσης να απευθύνω έκκληση σε όσους συμμετέχουν σε αυτό το σεμινάριο να τους πω ότι μπορούν να συμπληρώσουν ένα δελτίο αξιολόγησης το οποίο έχει διανεμηθεί. Αξιολόγησης αυτού του σεμιναρίου με τέτοιο τρόπο ώστε μετά να μπορέσουν να παραδοθούν αυτά τα δελτία στη γραμματεία στο τέλος. Και ευθύ εξ αρχής και εξ ονόματος των διευθυντών των τεσσάρων αυτών οργάνων δίνω τον λόγο στον Κρίστιαν Λέτμαϊερ που είναι διευθυντής επικεφαλής του ΣΕΝΤΕΦΟΠ. Παρακαλώ. Έχετε τον λόγο. Αγαπητά μέλη του Ευρωκοινοβουλίου, αγαπητοί Ευρωβουλευτέ, κυρίε και κύριοι, εξ ονόματο τη δική μου υπηρεσία και των υπηρεσιών, είναι δική μου χαρά να σα καλωσορίσω και θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Μπερές και την κυρία Τσούμπερ και όλα τα μέλη τη Επιτροπή Απασχόληση που διοργάνωσαν αυτό το σεμινάριο σήμερα για μα και μαζί μα. Επίσης, σε σχέση με τον κύριο Πράτσεφανέη, θα ήθελα να ευχαριστήσω, καθώς επίσης και τον κύριο Πρωθυπουργό Λαζάρ, Πρωθυπουργό της Μολδαβίας, τα μέλη Μπέκερ, Γκέντς, Μακιντάιρ, τον κύριο Κόμπιχεν, που είναι ο επικεφαλής της ΣΕΜΕΤ, Φίσμπαχ Πίτερ από πλευράς των συνδικάτων των κρατικών υπηρεσιών και τέλος τον κύριο Ρεγκού από το, το Διευθυντήριο των European Policy Advisors. Παρότι είναι δύσκολο να πει κανείς ακριβώς τι είναι το ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο, είναι ακριβώς η ιδιαίτερη αυτή πτυχή για την flexicurity, security και την πολιτική απασχόληση. σε Αυτό το κοινωνικό πρότυπο που διαφοροποιεί την Ευρώπη από τη ΣΥΠΑ και άλλες χώρες. Πέρα από διαφορετικά ιδεολογικά θέματα, αυτό συναποτελεί ένα τμήμα της ευρωπαϊκής ταυτότητας. Ο πρόεδρος Μπαρόζο το 2012 κάλεσε για ένα εξυγχρονισμένο σύστημα κοινωνικής προστασίας και υπογράμμισε ότι ο κοινωνικός διάλογος είναι κέριο στοιχείο του ευρωπαϊκού κοινωνικού Πρωτέπου δεν το παρατηρούν πάντα οι πολίτες, όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει και ιδιαίτερα σήμερα έχει μια ιδιαίτερη κοινωνική συνιστόσα. Όπως τα παραδείγματα των σκανδιναβικών χωρών της Γερμανίας και της Αυστρίας καταδεικνύουν, αυτό δεν είναι κάποιο εμπόδιο ή πρόσκομα, αλλά μάλλον ένας λόγος που ευνοεί την ανταγωνιστικότητα κιόλας. Και όσον αφορά την αηφορία στην ανταγωνιστικότητα, αυτή εξαρτάται σε κάποιο βαθμό και συνδέεται με τις κοινωνικές επενδύσεις και τα συστήματα προστασίας για τους πολίτες. Εξού και ο τίτλος για το σημερινό σεμινάριο. Δεν προσπαθεί να τετραγωνίσει τον κύκλο καθόλου. Αντανακλά αυτό το οποίο θα έπρεπε να είναι πρόδειλο και προφανές. Οι τέσσερις υπηρεσίες, SEDEFOP, ε, ETF, OSA και Eurofound, αντανακλούν από την απλή ύπαρξή τους ότι ανησυχούν και ενδιαφέρονται για αυτά τα θέματα τα ευρωπαϊκά όργανα. Η Eurofound και η SEDEFOP το 1975 είχαν ιδρυθεί ως ε, οι πρώτες υπηρεσίες. Έχουμε τριμερείς, ε, τριμερή διοικητικά συμβούλια σε, αυτές, ε, σε αυτά τα όργανα. Συμμετέχουν οι κοινωνικοί εταίροι που η συμμετοχή τους είναι τόσο σημαντική όπως γράμισε ακριβώς ο κύριος Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μπαρόζο. Το σημερινό σεμινάριο είναι πραγματικά μια μεγάλη ευκαιρία για να δείξουμε και καταδείξουμε πώς συνεισφέρουν οι υπηρεσίες μας και να συνεισφέρουμε και προσθέσουμε σε μια συζήτηση που βρίσκεται υπό εξέλιξη για τις κοινωνικές πολιτικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα προσεγγίσει την Ευρωπαϊκή Ένωση στους πολίτες. Θα αυξήσει την ε, ταυτότητα και τον ευδιάκριτο χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. <clears throat> Σε πολλές χώρες υπήρξε σκεπτικισμός εναντί της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν πραγματικά μπορούμε δηλαδή εμείς να βελτιώσουμε τις ζωές των πολιτών μας Επίσης θέλω να καλωσορίσω και να ευχαριστήσω και τους δύο συναδέλφους ε, από την Επιτροπή <clears throat> Απασχόλησης και των οργάνων που διοργάνωσαν αυτό το σεμινάριο. Ευχαριστώ λοιπόν πολύ ε, όλους σας. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Λεπμάιρ Και τώρα θα δώσω τον λόγο Πρώτα απ' όλα θέλω να καλωσορίσω τον Σαβιέ Πράτσα Μονέ που είναι ο Γενικός Διευθυντής ε, <clears throat> για την εκπαίδευση και τον πολιτισμό στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και θέλω να του δώσω τον λόγο για να μας παρουσιάσει το keynote speech, τον κύριο λόγο που ε, έχει να παρουσιάσει σε αυτό το σεμινάριο. Καλημέρα σας κυρία Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με ευχαριστίες. Ευχαριστώ την Επιτροπή Απασχόλησης, ίσως και γιατί πριν από δυόμιση χρόνια πολύ συχνά είχα να κάνω με την Επιτροπή Απασχόλησης και ειλικρινά θυμάμαι ότι πάντα οι συζητήσεις που είχα μαζί σας ήταν ιδιαίτερα επικοδομητικές και ιδιαίτερα με την κυρία Μπερές. Κάτι άλλο, όχι τόσο προσωπικό, αλλά να υπάρχει ένα μάθημα για το μέλλον που έχουμε να πάρουμε όσον αφορά το μέλλον του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου είναι ότι η απασχόληση και τα επαγγελματικά προσόντα πάνε μαζί. Και όσοι φορείς ασχολούνται με το ένα και με το άλλο θέμα στα κράτη-μέλη θα πρέπει να συνεργάζονται, ενώ αντίθετα δεν μιλάνε αρκετά συχνά μεταξύ τους. Γι' αυτό πολύ χαίρομαι που βρισκόμαστε εδώ σήμερα. Ευχαριστώ επίσης και τις διάφορες, τους διάφορους οργανισμούς. Νομίζω ότι οι πολίτες δεν καταλαβαίνουν πώς είναι δυνατόν να υπάρχουν αυτές οι τέσσερις υπηρεσίες που ασχολούνται στην Ευρώπη και στις γείτονες χώρες, πώς λοιπόν αυτές οι τέσσερις υπηρεσίες δεν καταφέρουν να συνεργαστούν αρκετά μεταξύ τους. Και έπειτα γιατί βρισκόμαστε εδώ εμείς οι τέσσερις. Υπάρχει ένας βασικός λόγος και αυτός είναι ότι οι υπηρεσίες μας θα βοηθήσουν να έχουμε πολιτικές και να εκπονούμε πολιτικές οι οποίες βασίζονται πολύ περισσότερο σε γεγονότα, σε δεδομένα. Ε, πρέπει να μάθουμε περισσότερα για το τι συμβαίνει, τι ισχύει στις διάφορες χώρες, να χρησιμοποιήσουμε την εμπειρία μας. Νομίζω επίσης ότι είναι πάρα πολύ καλό που το σεμινάριο αυτό ονομάζεται Κοινωνική Ευρώπη και Ανταγωνισμός. Γιατί, γιατί Πραγματικά η ουσία του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου δεν είναι μόνο το ότι η αλληλεγγύη είναι κάτι θετικό, ο κοινωνικός διάλογος είναι κάτι θετικό, είναι και το ότι είναι ουσιαστικά και θεμελιώδη στοιχεία για την ανταγωνιστικότητα. Αν θέλουμε να κερδίσουμε και να έχουμε ένα πραγματικά ισχυρό ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο, αυτό θα το πετύχουμε όχι μόνο ενισχύοντας την αλληλεγγύη, αλλά εάν φροντίσουμε για τα οικονομικά ωφέλη από την αλληλεγγύη. Αυτό ακριβώς λοιπόν θα προσπαθήσουμε σήμερα να κάνουμε. Επιτρέψτε μου λοιπόν πολύ σύντομα να σας πω τρία πράγματα. Πού βρισκόμαστε όσον αφορά το κοινωνικό μοντέλο, ποιες είναι οι προοπτικές για το μέλλον και μετά θα αναφερθώ σε έναν τομέα ο οποίος κατά τη γνώμη μου μπορεί να μην σας εκπλήσει. Εξακολουθούμε να αγνοούμε και είναι το μέλλον του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου. Εδώ μιλάω εκ μέρου και αυτού μου, έτσι. Καταλαβαίνετε ότι για το κοινωνικό μοντέλο δεν μπορώ να μιλήσω εκ μέρου ολόκληρη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής, οπότε τα σχόλια που θα σας κάνω είναι προσωπικά. Λοιπόν, πώ έχει σήμερα το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο. Είναι προφανές ότι όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή τη εδώ και τόσα χρόνια φτιάχνει και έχει στη διάθεσή της με τη διεύρυνση που έκανε. Όλα αυτά αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε δοκιμασία, ακριβώς επειδή βρισκόμαστε σε κρίση. Και μάλιστα όταν οι οικονομικοί αυτοί περιορισμοί πιέζουν υπερβολικά τις δημόσιες δαπάνες, άρα και τις ε, δαπάνες των χωρών μελών, πάνω στις ε, παροχές και το κοινωνικό μοντέλο. Τώρα η Ευρώπη τι ρόλο έχει μέσα σε όλα αυτά. Νομίζω ότι είναι καλό να αποφύγουμε να λέμε μεγάλα λόγια για την Ευρώπη. Ας κοιτάξουμε πρώτα απ' όλα τους περιορισμούς που έχει η Ευρώπη. Και ο πρώτος περιορισμός που αντιμετωπίζει είναι καθαρά συνταγματικό για την εκπαίδευση, την κοινωνική προστασία. Τα κράτη-μέλη, οι βουλευτές, ο κόσμος θέλουν η Ευρώπη να παίζει ένα καλό ρόλο, αλλά περιορισμένο ρόλο. Το ίδιο το συνταγματικό δικαστήριο στη Γερμανία είπε ναι κοινωνικές πολιτικές, αλλά όχι παραπάνω. Οπότε μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για έναν πραγματικό περιορισμό. Αλλά εάν πολιτικές ε, αυτές δεν κάνουν τη διαφορά, πώς θα γίνει. Γι' αυτό και πρέπει να φροντίσουμε να δείξουμε στους πολίτες ότι μπορεί η Ευρώπη να συνεισφέρει θετικά για την επιβίωση και την ευημερία του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να μην το ξεχνάμε. Τώρα υπάρχουν τρία εμπόδια όσον αφορά την πολιτική για το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο. Το πρώτο είναι η πραγματική φύση των πολιτικών που προσφέρουν αυτή την κοινωνική ευημερία ενέργεια για παράδειγμα. Αν θέλετε να εκπονήσετε μια πολιτική για την ενεργειακή ασφάλεια, τότε πρέπει να αναλύσετε τις οικονομικές πραγματικότητες, τα τεχνικά ζητήματα, να συζητήσετε κοινού στόχους και να καταλήξετε σε ένα σεβασμό μεταξύ εθνικών συμφερόντων. Αυτή είναι η καθημερινή ζωή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν όμως έρθετε στο κοινωνικό τομέα και στο ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο, πρέπει να τα κάνετε όλα αυτά που ήδη είναι πολύ περίπλοκα και επιπλέον όμως πρέπει να λάβετε υπόψη σας τις τόσο ισχυρές συνήθειες, νοτροπίες, ιδεολογίες που ισχύουν στις διάφορες, χρώτες, στις διάφορες χώρες μέλη. Αυτοί οι περιορισμοί μπορεί να μην σας φαίνονται τόσο απτοί, είναι όμως πραγματικοί και δυσκολεύουν τη ζωή μας προκειμένου να φέρουμε την προστιθέμενη αξία που θέλουμε. Γιατί Θέλουμε να είμαστε αντικειμενικοί και αυτό δεν πρέπει να το υποτιμάμε. Αυτό ήταν το πρώτο εμπόδιο. Το δεύτερο εμπόδιο είναι ένα παράδοξο. Είναι ότι από τη μια μεριά οι κοινωνικέ αλλαγέ, δηλαδή όλα αυτά που περιορίζουν το κοινωνικό μοντέλο, προέρχονται από εσωτερικού παράγοντες τη κοινωνία μα και ακολουθούν τα μοντέλα των διάφορων κοινωνικών μοντέλων, είτε είναι ακλοσαξονικό, είτε είναι σκανδιναβικό, είτε οτιδήποτε άλλο. Από την άλλη όμως η κρίση και η παγκοσμιοποίηση απαιτούν περισσότερη και πιο ουσιαστική δράση για την κοινωνική προστασία και τις κοινωνικές πολιτικές. Η παγκοσμιοποίηση, για παράδειγμα. Το πιο σημαντικό, κατά τη γνώμη μου, από την παγκοσμιοποίηση, στην Ευρώπη κυρίως, και για το κακό κοινωνικό μοντέλο, είναι κάτι πολύ απλό. Όταν η Τέο Σοβιετική Ένωση, η Ινδία, η Κίνα αποφάσισαν να μπουν στο παγκόσμιο εμπόριο, τότε το εργατικό δυναμικό διπλασιάστηκε. Και αυτό εξηγεί σε ένα μεγάλο μέρος γιατί αμφισβητείται το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο. Γιατί υπάρχει πίεση στους μισθούς και στην ανταγωνιστικότητα από αυτές τις δυνάμεις. Έπειτα οι διαρθρωτικές ε, δομές αλλάζουν εξαιτίας της γύρανσης του πληθυσμού, ε, εξαιτίας ε, των προδιαγραφών που υπάρχουν ένας διεθνής οργανισμός για την προστασία των κοινωνικών ε, κεκτημένων ε, στηρίζεται γύρω από τις οικογενειακές παραδόσεις, τη μετανάστευση, την ισότητα αντρών και γυναικών, την διαβίου κατάρτιση κλπ. Οπότε υπάρχει μια δυσκολία εδώ η οποία απορρέει από τις τάσεις που υπάρχουν από τις εσωτερικές πιέσεις στα διάφορα κοινωνικά μοντέλα και τον δημογραφικό παράγοντα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο λοιπόν να βρούμε το ρόλο που πρέπει να παίξουν οι εθνικές ή οι ευρωπαϊκές αρχές σε αυτό το πλαίσιο. Και το τελευταίο μου τρίτο εμπόδιο που δεν ε, λαμβάνουμε πολύ υπόψη γιατί δεν τον γνωρίζουμε, είναι ο εξή. Και αυτό είναι η ποικιλομορφία που επικρατεί μεταξύ 28 διαφορετικών χωρών. Δείτε την κρίση, δείτε τι κοινωνίε μα, δείτε ε, την ανεργία των νέων, των γυναικών. Οποιοδήποτε δείκτη, ο οποίο είναι σημαντικό για το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο, θα δείτε ότι διαφέρει δραστικά από χώρα σε χώρα. Είναι ψευδέστηση λοιπόν να νομίζουμε ότι μπορούμε να έχουμε ουσιαστικέ πολιτικέ και απαντήσει για το μελλοντικό ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο που θα είναι οι ίδιε για όλου. Άρα αυτή την κυκλομορφία πρέπει να τη διαχειριστούμε και πρέπει να αποφύγουμε τον κίνδυνο τα λόγια μα και οι πολιτικέ μα για το κοινωνικό μοντέλο να είναι ίδιε παντού. Αυτό είναι ο κίνδυνος επειδή θέλουμε να προστατεύσουμε τους ε, πάντες. Δεν μπορούμε λοιπόν να χρησιμοποιούμε γενικόλογα ε, τις ε, απόψεις μας χωρίς να μπαίνουμε σε κάτι πιο συγκεκριμένο. Σας είπα λοιπόν, η εσωτερική εξέλιξη των συστημάτων κοινωνικής προστασίας, η ποικιλομορφία, η γύρανση του πληθυσμού, είναι πράγματα τα οποία μειώνουν τη σύγκληση και δημιουργούν μεγαλύτερη ένταση ακόμα στην κρίση. Πρέπει λοιπόν αυτά τα τρία στοιχεία να τα λάβουμε υπόψη μας αν θέλουμε καλές προοπτικές για το μέλλον του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου. Τώρα έρχομαι ακριβώς στο μέλλον. Είπαμε τους περιορισμούς, τα εμπόδια, τα προβλήματα. Δεδομένως, ο δεδομένο ότι υπάρχουν όλα αυτά, είναι πολύ εύκολο κανείς να προσπαθήσει να καλυφθεί και να προστατευτεί από το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο. Όμως πόσο μπορούμε να βοηθήσουμε την Ευρώπη εμείς να μιλάει με μία φωνή όταν βλέπουμε την τεράστια ποικιλομορφία που υπάρχει στην αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης και στις επιπτώσεις της κρίσης αυτής της χώρας μας. Και ενώ προσπαθούμε να βρούμε μια έξοδο από την κρίση, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να βρει ποιο είναι ο δικό τη ρόλο, να έχει έναν πιο ισχυρό ρόλο σήμερα από ό,τι κατά το παρελθόν. Για έναν πολύ απλό λόγο, και αυτό είναι το κόστος της μη επένδυσης ή της λάθος επένδυσης, όταν δεν επενδύουμε στα προσόντα, στις δεξιοτεχνίες, στους ανθρώπους. Οι άνθρωποι και η γνώση παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στο μέλλον της Ευρώπης και της οικονομίας της, ε, της κοινωνίας της γνώσης. Το καλό νέο πάντως είναι ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες παρά το σκεπτικισμό που έχουν για την Ευρώπη γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο ενώνει τους Ευρωπαίους. Ρωτάτε από τη Ρήγα στην Αθήνα, τους Ευρωπαίους πολίτες, τι περιμένουν από τις ευρωπαϊκές αρχές τώρα στην περίοδο της κρίσης, ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι κοινωνίες μας και τι σας απαντάνε το ίδιο. Δουλειά, απασχόληση, μείωση της φτώχειας, κοινωνικές υπηρεσίες, αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος εκπαίδευση και προσόντα κατάλληλα για τον 21ο αιώνα. Άρα η Ευρώπη δεν μπορεί παρά να έχει ένα σημαντικό ρόλο. Ποιο όμως ακριβώς. Η διάγνωση είναι εύκολη. Οι λύσεις όμως είναι πιο δύσκολες. Η ολοκλήρωση της Ευρώπης ανθίζει όσον αφορά την ανάπτυξη κατά τη διάρκεια των κρίσεων. Τώρα λοιπόν Ακριβώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε μήνε, μήνες, οχτώ μήνες θα έχουν μια εντολή. Το νέο Κοινοβούλιο και η νέα Επιτροπή δηλαδή σε λίγους μήνες θα ξεκινήσουν τη νέα τους θητεία και θα φροντίσουν να καταλήξουν σε μια στρατηγική εξόδο από την κρίση που θα δίνει απαντήσεις στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο. Είναι δύσκολο, ναι, αλλά δεν είναι αδύνατο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρώτα απ' όλα μπορούν να βοηθήσουν να εντοπιστούν οι επιπτώσεις της κρίσης τις πολιτικές μας, να φροντίσουν για κοινωνική δικαιοσύνη, για τις κατάλληλες μεταρρυθμίσεις και να φροντίσουν για βιώσιμη ανάπτυξη. Ε, οι τέσσερις οργανισμοί ακριβώς αυτό θα προσπαθήσουν να κάνουν από σήμερα. Τέλος. Έξι λεπτά νομίζω έχω ακόμα, ε, αν ε, κατάλαβα καλά το χρόνο που έχω στη διάθεσή μου. Γιατί μπορούμε να κάνουμε περισσότερα υπάρχουν ήδη στην ημερήσια διάταξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά πρέπει να είμαστε περισσότερο παρόντες, πιο ισχυροί. Και αυτό θα κάνω και εγώ εδώ στο Κοινοβούλιο, προκειμένου να στηρίξουμε την εκπαίδευση και τις δεξιοτεχνίες. Γιατί είναι στοιχείο κλειδί για να αναβαθμίσουμε τη μελλοντική ημερήσια διάταξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα επόμενα πέντε χρόνια. Εκπαίδευση και δεξιοτεχνίες είναι ισοτική σημασία για την ευρωπαϊκή ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα, για την απασχόληση και για την ε, δυνατότητα προσαρμογής σε αλλαγές και για τη δικαιοσύνη βέβαια, την κοινωνική. Θέλουμε μια στρατηγική εξόδου από την κρίση που να βασίζεται σε αυτά τα στοιχεία, στη γνώση, γιατί μόνο μέσα από τη γνώση μπορούμε να καθορίσουμε τις δυνατότητες που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση να στηρίξει το κοινωνικό της μοντέλο. Και κάτι πιο σημαντικό είναι ότι έρχεται ένα τσουνάμι στον τομέα της εκπαίδευσης. Τώρα έχουμε τη δυνατότητα να το μεταλλάξουμε και να το κάνουμε μια ευκαιρία για την Ευρώπη και όχι μια πρόκληση. Πάνω από έναν αιώνα οι άνθρωποι διδάσκονται με τον ίδιο τρόπο. Το 1913 ένας χειρούργος και σήμερα ένας χειρούργος δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο έξω από τον χώρο χειρουργίας. Το ίδιο και ένας καθηγητής. Τώρα γίνονται οι αλλαγές, τώρα αρχίζουν οι αλλαγές με την τεχνολογία και την παγκοσμιοποίηση. Συνδυασμένες έχουν τεράστιε επιπτώσει σε κάθε πτυχή της κοινωνίας μας. Μουσική, τράπεζες, μέσα ενημέρωση, Ε, ήρθε η ώρα για αλλαγές στην εκπαίδευση. Να χρησιμοποιήσουμε μείγμα τεχνολογίας και κατάρτισης. Η δυνατότητα οι άνθρωποι να μπορούν να μάθουν όπου και όποτε θέλουν. Είμαι Ισπανό. Θα έχετε ακούσει για τον Δοκιχώτη βέβαια. Λοιπόν, ο, Δοκιχώτη, ο γράφτηκε πριν από 400 χρόνια. Μέχρι πριν από 10 χρόνια μπορούσαμε να διαβάσουμε τον Δον Κιχώτη ναι. μόνο εάν υπήρχαν αντίγραφα του Δον Κιχώτη. Σήμερα όμως οποιουσδήποτε, οπουδήποτε, οποτεδήποτε και δωρεάν μπορεί να διαβάσει τον Δοκιχώτη. Ε, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν εκτιμάμε αρκετά για τις δυνατότητες που μας δίνει, για τα πόσα μας υπόσχεται για το μέλλον των παιδιών μας και των κοινωνιών μας. Αυτό ακριβώ λοιπόν θέλω να σα πω λοιπόν, ότι πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα επικεντρώσουμε τι προσπάθειέ μα στο μέλλον, σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο, ώστε η εκπαίδευση να αποτελέσει μέρο όχι μόνο της ημερήσιας διάταξης ε, της εκπαίδευσης της χώρας μας, αλλά ολόκληρης της Ευρώπης. Και θα σας δώσω εδώ τέσσερις προκλήσεις, οι οποίες θα βρεθούν μπροστά στην Ευρώπη πολύ σύντομα. Πρώτον, τα νέα δεδομένα. Και ποια είναι αυτά, μαζί με το CD έχουμε συζητήσει στον ΩΣΑ, ότι η Ευρώπη δεν έχει αρκετά προσόντα. Δηλαδή οι πιο μεγάλοι στην ηλικία δεν έχουν αρκετά προσόντα. Μόνο τρεις χώρες στην Ευρώπη ε, διαπιστώνουν ότι οι ενήλικες τους διαθέτουν τις δεξιοτεχνίες και τα προσόντα που χρειάζονται. Αντίθετα στις μεγάλες χώρες διαπιστώνουμε ότι οι δεξιοτεχνίες αυτές είναι πάρα πολύ λίγες στις ηλικίε αυτές. Άρα πλήττεται η ανταγωνιστικότητά τους και η Ευρώπη. Τι είναι? Ανταγωνιστικότητα. Ένα στους πέντε στην Ευρώπη ενήλικας μάλιστα έχει τόσο περιορισμένα προσόντα που κινδυνεύει να μην μπορεί να βρει δουλειά καθόλου. Το εργατικό δυναμικό στην Ευρώπη έχει μειωθεί βέβαια τα τελευταία χρόνια, το ξέρουμε. Άρα αυτή είναι η πρώτη πρόκληση. Συνεπώς πρέπει να βελτιώσουμε τα προσόντα των ελίκων στην Ευρώπη. Δεύτερον, επενδύσεις. Υπάρχει ένας πολύ απλός ε, τρόπος, όπως είπε κάποιος από το Harvard, ένας πρίτανης. Hm. Είπε αν πιστεύετε ότι είναι ακριβή. Αν είναι ακριβή, προσπαθήστε να την κάνετε πιο φθηνή. Όσον αφορά τώρα την ε, ανάπτυξη στην Ευρώπη, πρέπει να έχουμε επενδύσεις οι οποίες να είναι υποφελείς για την εκπαίδευση από τις έρευνές μας 10 χώρες έχουν μειώσει τις δαπάνες τους σε αυτό το τομέα σε απόλυτους αριθμούς. Έρχομαι στην τρίτη πρόκληση, είναι αναγνώριση των, προσεν, των προσόντων. Έχουμε τα ευρωπαϊκά πλαίσια, αναγνώριση προσόντων, πολλών, ιστίες κτλ. Πολλέ διαδικασίε. Ποια είναι όμω η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι ότι ακόμα δεν έχουμε έναν χώρο μέσα στον οποίο να μπορούν ελεύθερα να κυκλοφορούν οι, οι ιδέες και οι ό,τι περνάει το κεφάλι των ανθρώπων. Τέλος, δεν εκμεταλλευόμαστε τις δυνατότητες που δίνει η εκπαίδευση και η τεχνολογία για την κοινωνία μας ολόκληρη. Πρέπει όλοι να μπορούν να επωφεληθούν και να επικρατεί και η αριστεία. Άρα λοιπόν πρέπει να αλλάξουμε τα μοντέλα της εκπαίδευσής μας. Έχουμε τη δυνατότητα σήμερα τις προκλήσεις αυτές, τις τέσσερις, να τις αντιμετωπίσουμε, αλλά οι χώρες από μόνες τους δεν μπορούν να τις αντιμετωπίσουν. Αυτό είναι το πιο ισχυρό επιχείρημα. Επικουρικότητα, έτσι ώστε να μπορούμε να παίξουμε έναν μεγαλύτερο ρόλο στην εκπαίδευση στις χώρες μέλη αλλά και στην Ευρώπη ολόκληρη. Τέλος, κάνω μια έκκληση. Όταν συζητάμε το μέλλον του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου, σκεφτόμαστε πώς οι δεξιοτεχνίες και τα προσόντα μπορούν να συνεισφέρουν στην ευημερία και την ανταγωνιστικότητα. Και δεν είμαστε μόνοι μας στον κόσμο. Το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο και μια πιο ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση για να γίνουν πραγματικότητα στο μέλλον θα πρέπει να θυμόμαστε ότι η πρόκληση της Ευρώπης είναι να βελτιώσει τις ηλικές συνθήκες ζωής των Ευρωπαίων να μην παραμείνει μια ψευδέστηση, να υπάρχουν αποτελεσματικές αγορές και αρκετή φυσική πόρη. Αυτό θα έλυνε το πρόβλημα. Δεν πρέπει όμως να κοιτάμε και πέρα από τα σύνορά μας. Μερικές φορές η Ευρώπη κάνει κηρύγματα στους άλλους. Στην απασχόληση μάλιστα θα λέγαμε ότι αυτό ισχύει περισσότερο. Ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα αποτελεί παράδειγμα σε έναν χώρο που βασίζεται στο δίκαιο. Μην δίνουμε λοιπόν εμείς μαθήματα στους άλλους, ας φροντίσουμε πρώτα να αποτελέσουμε ένα καλό παράδειγμα με το δικό μας κοινωνικό μοντέλο, ώστε οι άλλες χώρες να μπορούν να κοιτούν προς την Ευρώπη όπως κοιτούσαν πριν από μερικά χρόνια και να τη θεωρούν πηγή έμπνευσης. Αυτό θα καθορίσει το μέλλον μας και την αξιοπιστία μας. Και βέβαια δεν τελειώνει η ιστορία εκεί. Πρέπει να σκεφτούμε ποιο είναι ο ρόλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση για να διατηρήσει το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο. Δεν είναι δικιά μου δουλειά, σίγουρα όμω είναι δουλειά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των τεσσάρων οργανισμών που βρίσκονται εδώ, ώστε η συζήτηση αυτή να παραμείνει ζωντανή και στο μέλλον. Σα ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτά που μας είπατε, που ήταν πολύ ενδιαφέροντα. Κυρίως στη σημερινή εποχή στην οποία ζούμε και τις ανάγκες που έχουμε και πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Δυστυχώς η πραγματικότητα και τα ιδανικά δεν συμπίπτουν και δεν συγκλίνουν. Και αυτό είναι ένα από τα προβλήματα που σήμερα πρέπει να αντιμετωπίσουμε ως προκλήσεις. Περνάμε στη θεματολογική μας ε, ανάλυση τώρα και για τις παρουσιάσεις ε, των ε, διευθυντών των τεσσάρων αυτών οργάνων που υπροσωπούνται σήμερα εδώ και συμμετέχουν. Παρακαλώ κάθε παρέμβαση να έχει το πολύ 10 λεπτά διάρκεια <clears throat> πάνω κάτω. Και δίνω και πάλι τον λόγο στον κύριο Κρίστιαν, Κρίστιαν Λετμάιερ, διευθυντή της ΣΕΝΤΕΦΟΠ θα έχουμε αυτή την παρέμβαση εξ ονόματος της ε, ΣΕΝΤΕΦΟΠ για την προπαρασκευή ακριβώς των πολιτών για την αγορά εργασίας ε, που βρίσκεται υπό μετεξέλιξη και να υπάρξει έτσι εκπαίδευση και κατάρτιση κατάλληλη. Ευχαριστώ. Ladies and gentlemen. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ευρωβουλευτές, ε, το ΣΕΝΤΕΦΟΠ είναι το η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Επαγγελματική Κατάρτιση υποστηρίζει νέε πολιτικέ, ετοιμάζει στοιχεία και βοηθάει στη διαμόρφωση αυτών των πολιτικών. Αυτό δεν σημαίνει μόνο στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με τι κυβερνήσει των κρατών μελών και του κοινωνικού εταίρου, αλλά σημαίνει ε, επαφή με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, ε, συζητήσεις, ε, με οργανώσεις, ε, συζητήσεις με οργανώσεις των stakeholders κτλ. Επίσης, ε, προσπαθούμε να πιέσουμε την Κομισιόν να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στις ε, πολιτικές για την αγορά εργασίας. Θέλουμε να βελτιώσουμε την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη διαβημάθηση. Φυσικά, ε, ένας από τους σημαντικότερους δείκτες της ποιότητας του συστήματός μας είναι η προσπάθεια που κάνουμε για μάθηση ε, και η διαβίου προσπάθεια για να αναβαθμίσουμε τα, τις δεξιότητές μας, ε, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και τις εξελίξεις της. Ε, εστιακό σημείο είναι οι εξελίξεις αγοράς εργασίας, οι μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες τάσεις που θα επηρεάσουν την επαγγελματική κατάρτιση, την εκπαίδευση, και την παροχή τέτοιων συστημάτων εκπαίδευση και κατάρτιση από τα κράτη-μέλη. Ε, ο εξυγχρονισμό αυτών των συστημάτων και η ε, ευθυγράμμισή τους με την αγορά εργασίας λαμβάνει υπόψη τους μηχανισμούς προσαρμογής ε, στις νέες τάσεις. Προκειμένου να έχουμε τις σωστές αποφάσεις για αυτά τα θέματα. Μετράμε όχι μόνο το... Από τις μελέτες που έχουμε κάνει έχουμε δει ότι η ζήτηση για υψηλού επίπεδου προσόντα αλλά και μεσαίου επίπεδου προσόντα θα είναι πολύ σημαντική τα επόμενα χρόνια. Το να δώσουμε εργαζόμενους ε, με προσόντα που προσαρμόζονται στην αγορά εργασίας είναι πολύ σημαντικό για τους νέους ανθρώπους ε, είναι πολύ καλό ε, συνολικά για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Αυτή η τάση ότι θα χρειαστούμε ε, υψηλού επίπεδου προσόντα σημαίνει ότι θα πρέπει να εστιάσουμε περισσότερο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και όχι τόσο στη δευτεροβάθμια. Παρότι και, αυτό είναι, και αυτή η πολιτική και αυτή η προσπάθεια είναι πολύ απαραίτητη. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να δώσουμε στους ανθρώπους τα προσόντα τα οποία θα είναι και γενικά αλλά και εξειδικευμένα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και για να βρουν δουλειά και για να την κρατήσουν. Ο Ποτάρης, ο Μπουτάρης, συγγνώμη, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, και μην ξεχνάτε, είπε ότι Στη Θεσσαλονίκη υπήρχαν παλιά καλές τεχνικές σχολές. Ε, μην ξεχνάτε όμως ότι στη Θεσσαλονίκη σήμερα η ανεργία των νέων έχει φτάσει στο 60%. Όλες αυτές οι σχολές σήμερα ε, έχουν εξαφανιστεί. Έχει μειωθεί η ζήτηση τέτοιων ανθρώπων από τέτοιες σχολές. Οι σχολές αυτές δεν είναι πλέον ελκυστικές. Και τα προσόντα αυτά δεν είναι ελκυστικά. Αν συνειδητοποιήσουμε ότι και τα προσόντα ε, ενός μετρίου επίπεδου θα εξακολουθήσουν να είναι σημαντικά, πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα της ε, ελκυστικότητας το, της επαγγελματικής κατάρτισης. Ε, σε ορισμένε χώρε, επίση υπάρχουν τρομερέ διαφορέ από χώρα σε χώρα στην επαγγελματική κατάρτιση. Ε, σε ορισμένε χώρε ε, το 30% των παιδιών ακολουθούν τέτοια τεχνική κατάρτιση, σε άλλε χώρε το 70%. Ε, επίση, η τεχνική κατάρτιση, η μαθητεία, ε, η εκμάθηση μιας τέχνης θεωρείται πάντα δευτεροκλασάτη απασχόληση σε σχέση με τα πτυχία πανεπιστημίων. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει προσπάθεια για να έχουμε επαγγελματική κατάρτιση υψηλής, υψηλού επίπεδου. Επίσης, να υπάρχει δυνατότητα να μεταπηδήσει κανείς από την τεχνική ε, εκπαίδευση στην ανώτατη. Οι χώρες οι οποίες έχουν επενδύσει πολύ στην, επαγγελματική, στην τεχνική και επαγγελματική κατάρτιση έχουν βγει κερδισμένε. Υπάρχουν 30 εκπαιδευτικά προγράμματα. Τα 15 αφορούσαν την ε, πανεπιστημιακή εκπαίδευση και τα υπόλοιπα υψηλού επίπεδου τεχνική κατάρτιση. Επίσης είναι σημαντικό να ενημερώνουμε τους γονείς αλλά και τους ενδιαφερόμενους ε, αν θέλουμε να βελτιώσουμε την ελκυστικότητα της επαγγελματικής κατάρτισης. Είναι σημαντικό να δίνουμε επαγγελματικό προσανατολισμό επίσης ε, στα παιδιά και στους γονείς. Ε, βεβαίως αυτό θα πρέπει να γίνεται παράλληλα με την προσαρμογή της επαγγελματικής κατάρτασης, κατάτησης και με τη συμμετοχή όλων των διαφερομένων και των εργοδοτών στη διαμόρφωση των, α, της τεχνικής εκπαίδευσης και των προσόντων που δίνει αυτή. Ε, όσοι προέρχονται από την τεχνική εκπαίδευση, ε, λόγω της κρίσης ε, δηλώνουν ότι έχουν δυσκολίες να βρουν μια δουλειά. Έχουμε στοιχεία από 142 χώρες που δηλώνουν ότι η δυσκολία το να βρούμε δουλειά πέρα από την ε, έλλειψη εμπειρίας ε, οφείλεται και στην έλλειψη κατάλληλων προσόντων. Πολλοί ενδιαφερόμενοι θεωρούν ότι η έλλειψη απασχολησιμότητάς τους οφείλεται στην, ε, στην, και στην έλλειψη ήπιων λεγόμενων προσόντων. Υπάρχουν διαφορετικές ανισότητες μεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης. Φυσικά, αλλιώς βλέπουν ε, οι καθηγητές ε, την ε, επαγγελματική κατάρτιση και αλλιώς οι εργοδότες. Το 70% των εργοδοτών θεωρούν ότι το σύστημα εκπαίδευσης και κατάρτισης φταίει για τους ε, εργαζόμενους που δεν έχουν τα απαραίτητα προσόντα. Αυτό που είπε ο Ξαβιέ στην ομιλία του για τις νέες τεχνολογίες φυσικά είναι ένα σημαντικό, μια σημαντική τάση, μια σημαντική συνιστόσα και πρέπει να τη λάβουμε υπόψη μας. Κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Είναι η πολύ σωστή μαθητεία στην αρχή της επαγγελματικής καριέρας κάποιου. Κάτι που πρέπει να αλλάξουμε και να βελτιώσουμε είναι να αυξήσουμε τον αριθμό των επιχειρήσεων που προσφέρουν τη δυνατότητα της μαθητείας. Βέβαια δεν μπορούμε να μπούμε σε πολλές λεπτομέρειες για αυτό το θέμα τώρα, αλλά πιστεύω ότι έχουμε στοιχεία ότι αν μια εταιρεία ετοιμάσει μαθητευόμενους, προσαρμόζει και την κουλτούρα για τον τρόπο μάθησης. Η επιχείρηση η ίδια, γίνεται μια, ένας οργανισμός ε, γνώσης και μάθησης. Και τα άτομα βγαίνουν μέσα στον, ε, σε έναν ανταγωνιστικό κόσμο ε, με προσόντα για να, για αντιδράσουν στις εξελίξεις αγοράς και για να είναι επιτυχής. Αυξάνεται δηλαδή η ανταγωνιστικότητά μας γενικά. Εάν οι εταιρείε γίνουν τέτοια φυτόρια γνώσης και μάθησης, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ε, τους ε, ήδη εργαζόμενους ως ε, καθηγητές τροποντινά ε, που θα διδάξουν τους νεότερους. Επίσης ε, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας το γεγονός ότι έχουμε κενά δεξιοτήτων. Αυτό το πρόβλημα, αυτά τα χάσματα μπορούν να επιληθούν με αυτή την αλληλεπίδραση των νέων με τις επιχειρήσεις. Επίσης κάποιος, πέρα από την αρχική μαθητεία που θα κάνει αμέσως μετά τις ε, σπουδές του, μπορεί να συνεχίζει να μαθαίνει μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας επίσης ε, ότι όσοι έχουν λίγα προσόντα, μεταξύ αυτών βρίσκονται και οι... Ε, από εκεί μάλλον θα προκύψουν οι μελλοντικοί άνεργοι. Όσοι έχουν χαμηλά προσόντα δεν έχουν τη δυνατότητα να προσαρμοστούν και αύριο μεθαύριο θα γίνουν οι ίδιοι άνεργοι. Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, θα ήθελα να πω εν κατακλείδη, είναι τρομακτικές. Και δεν έχουμε τους επαρκείς πόρους. Πιεζόμαστε πολύ. Αλλά κάνουμε ό,τι μπορούμε σε συνεργασία με τις άλλες υπηρεσίες, με την Κομισιόν. Προσπαθούμε να δώσουμε στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα στοιχεία, ούτως ώστε να, τις, να τα προσανατολίσουν για τα μέτρα που μπορούν να πάρουν. Σε ευχαριστώ πολύ κύριε Λετμάιε. Επίσης σας ευχαριστώ για την πολύ σημαντική αυτή παρέμβασή σας με την εισήγησή σας και για τις παρατηρήσεις που κάνατε για το έργο της υπηρεσίας της οποίας είσαστε πρόεδρος. Στη συνέχεια αμέσω θα δώσω τον λόγο στον κύριο Χουάν Μενέντες Βαλντές που είναι ο διευθυντής της Eurofound και που θα μας κάνει λόγο για ένα θέμα το οποίο αφορά την μεταμόρφωση, την αλλαγή πορείας μας, αλλαγή κατεύθυνσης προς μια ε, πιωσμένη Ευρώπη πιο ανταγωνιστική μέσω καλύτερων συνθήκων διαβίωσης και εργασίας. Χουάν Μενέντες Βαντές, έχετε τον λόγο παρακαλώ. Σε ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Όπως γνωρίζετε, Eurofound το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για την μετίωση των συνθήκων διαβίωσης και εργασίας ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσπαθούμε να δώσουμε στοιχεία για να βοηθήσουμε την ανάπτυξη των κοινωνικών θεμάτων. Το κοινωνικό πρότυπο διαδραματίζει ένα ρόλο κλειδιού με μεγάλη σημασία σε όλα τα θέματα όλα τα ζητήματα τα οποία τέθηκαν σε πιο εύρος και πώς μπορεί να διασφαλίσει το κοινωνικό της πρότυπο η Ευρωπαϊκή Ένωση και ταυτόχρονα να είναι, είναι η πιο ανταγωνιστική, μια από τις πιο ανταγωνιστικές ε, οικονομίες είναι μέρος των συζητήσεών μας. Έχουμε και το πρόγραμμα το οποίο ε, ε, βρίσκεται υπό ανάπτυξη και εξέταση και συζητούμε ακριβώς αυτά τα θέματα. Δηλαδή για μια καλύτερη επικέντρωση για στοιχεία, για καλύτερες μεταρρυθμίσεις και μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα συζήτηση, σε ποιο βαθμό η ανταγωνιστικότητα και η δικαιοσύνη, η αλληλεγγύη, η ανάπτυξη μπορούν να αποτελέσουν τμήματα και να έχουν ένα ρόλο. Ο Κρίστιαν Λετμάιερ είπε ότι έχουμε δυναμικό μας δείχνουν ότι υπάρχει κάτι το οποίο δεν είναι ε, δεδομένο για όλες τις χώρες και βλέπουμε ότι μπορούμε να παραμείνουμε στα ανώτερα επίπεδα στην ε, αξιολόγηση της ανταγωνιστικότητας και ταυτόχρονα να διασφαλίζουμε ασφαλή συστήματα και βιώσιμα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης. Και όλες αυτές, όλες αυτές οι χώρες και όλες αυτές οι πολιτικές πρέπει διαρκώς να προσαρμόζονται σε σχέση με αυτά τα πρότυπα. Και αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο που πρέπει να λαμβάνετε υπόψη. Πρέπει να προσαρμοζόμαστε στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κοινωνία μας. Για παράδειγμα, σε σχέση με την ηλικία των εργαζομένων ε, όσον αφορά την αναδιάρθρωση αγορών εργασίας για να είμαστε πιο λειτουργικοί και να μπορούμε να αντιδρούμε με πιο αποτελεσματικό τρόπο. Τα θέματα για προσαρμογές προσαρμογή κυρίως ε, και προσαρμοστικότητα και όχι εγκατάληψη του κοινωνικού προτύπου. Πρέπει να γνωρίζουμε ακριβώς τι θα αλλάξουμε, τι θα τροποποιήσουμε και πώς θα προσαρμόσουμε και θα προσαρμοστούμε. Και για να γίνει αυτό χρειάζονται γνώσεις. Πρέπει να υποπτεύουμε τις εξελίξεις και να δούμε πώς θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε αυτό το δύσκολο εγχείρημα ως πρόκληση. Και αυτός ακριβώς είναι ο ρόλος ε, της υπηρεσίας μας, του οργάνου μας. Να δώσουμε στοιχεία, γνώσεις που μπορούν να βοηθήσουν τους αρμόδιους στο πολιτικό επίπεδο να λαμβάνουν τις σωστές πολιτικές επίπεδες. Εποπτεύουμε και αναλύουμε τις εξελίξεις όσον αφορά τις συνθήκες και όρους εργασίας και απασχόλησης. Εποπτεύουμε τις τάσεις και παρατηρούμε το τι συμβαίνει σε σχέση με την αγορά εργασίας και πώς εξελίσσονται τα πράγματα σε σχέση με όλα αυτά στην Ευρώπη. Θα ήθελα να αναφέρω κάτι και αναφερόμενο στο έργο του Σαβιέ Πράτς να τονίσω κάπως τους όρους και συνθήκες απασχόλησης, working conditions. Είναι και στον τίτλο της υπηρεσίας μας, του Ιδρύματός μας. Βρισκόμαστε σε μια περίοδο κρίσης και ανεργίας. Μπορεί να πει κανείς ως λογικό επιχείρημα ότι οποιαδήποτε θέση απασχόλησης είναι σημαντική. Αληθεύει αυτό. Όμως η ποιότητα των θέσεων απασχόλησης είναι πολλές φορές ε, εξίσου σημαντικές και όχι μόνο για τα άτομα, αλλά επειδή για την κοινωνία συνολικά είναι κέρια σημασίας τα ποσοστά συμμετοχής στην αγορά εργασίας εξαρτώνται από τους, ε, την ποιότητα των συνθήκων απασχόλησης που ισχύουν στην αγορά εργασίας. Αν θέλουμε και πρέπει να εντάξουμε περισσότερους πολίτες ε, σε θέσεις απασχόλησης και να παραμείνουν σε απασχόληση, σε απασχόληση επί μακρότερα χρονικά διαστήματα, ε, διαστήματα χρειαζόμαστε επαρκείς όρους και συνθήκες για να γίνει αυτό. Να υπάρξουν επαρκή συστήματα κοινωνικής προστασίας και να υποστηριχθεί η ανάπτυξη και η ανταγωνιστικότητα. Και εδώ δεν κάνουμε λόγο μόνο για τους υπερήλικες ή ηλικιωμένους εργαζόμενους που θα εργάζονται περισσότερο και πρέπει να εργάζονται για, μεγαλύτερη χρονική διάρκεια λόγω του ότι γυράσκει ο πληθυσμός σήμερα στην Ευρώπη. Κάνουμε λόγο για τη διατήρηση ομάδων και κατηγοριών εργαζόμενων στην αγορά εργασίας. Δηλαδή ανθρώπων με διαφορετικές ανάγκες, με διαφορετικές δεξιότητες και ικανότητες ε, και με διαφορετικές ε, επιλογές, με ευθύνες όχι μόνο για παιδιά που ανατρέφουν, αλλά και για πιο ηλικιωμένους ε, συμπολίτες μας που ανήκουν στις οικογένειές τους. Αναλύουμε και προσπαθούμε να διαθέσουμε πληροφοριακά στοιχεία για το ποιες συνθήκες και όρια απασχόλησης μπορούν να δημιουργήσουν την αφορή, αηφορία στην απασχόληση. Ποιότητα λοιπόν των θέσεων απασχόλησης, που επίσης συσχετίζεται με τις πολιτικές μας. Πολιτικές σε σχέση με την περίθαλψη και την μέρημνα, κοινωνική περίθαλψη και μέρημνα. Και τα θέματα απασχολησιμότητας επίσης όσον αφορά το, τους εργαζόμενους για, την ποιότητα των θέσεων απασχόλησης πρέπει να τονίσουμε την ασφάλεια και την ε, υγεία στις θέσεις απασχόλησης στους χώρους εργασίας. Ε, είναι στοιχείο κλειδί αυτό για να, είναι, να διασφαλιστεί η αηφορία. Και ο Ξαβιέ Πράτσα και ο Κρίστιαν αναφέρθηκαν στις δεξιότητες και τις ικανότητες μέσω κατάρτισης και εκπαίδευσης. Εποπτεύουμε τους όρους και τις συνθήκες απασχόλησης από το 1990 και έχουμε και την τελευταία έκδοση το 2010 από το 1990 καλύπτουμε πάμπολες χώρες και έχουμε ε, εκπονήσει περίπλοκους ε, και κατάλληλους δείκτες αλλά και άλλα στοιχεία που είναι σημαντικά για τη διασφάλιση της ποιότητας στην απασχόληση μισθή για παράδειγμα ε, ποιότητα και όρια απασχόλησης και άλλα στοιχεία που αφορούν αυτή την πτυχή. Τα αποτελέσματα μπορούν να συνοψιστούν ως σε κάποιους τομείς καλά σε άλλους τομείς όχι τόσο καλά. Βλέπουμε ότι μία σε πέντε θέσεις απασχόλησης στην Ευρώπη <clears throat> χαρακτηρίζεται ακόμα ως χαμηλής ποιότητας, υποβαθμισμένη εργασία και πρέπει εδώ σε σχέση με τους όρους απασχόλησης να έχουμε προοπτικές να υπάρξει αλλαγή προς μια καλύτερη κατεύθυνση, προς μια αναβάθμιση και βελτίωση. Και εδώ έχουμε πολλά στοιχεία που μπορούν να είναι στοιχεία κρίσης και αξιολόγησης ε, πρώιμα ώστε να μπορέσουμε να κρίνουμε τις εξελίξεις για τα κοινωνικά συστήματα ασφάλισης και να δούμε τι μπορεί να γίνει για την αντιμετώπιση των προβλημάτων σε σχέση με τις δεξιότητες ε, που χρειαζόμαστε. Πέρα από αυτούς τους δείκτες και ενδείκτες ε, έχουμε επίσης και τα θέματα υγείας, αλλά επίσης ε, και τα θέματα πώς μπορούμε να επενδύσουμε στην ε, διοργάνωση της εργασίας, δηλαδή χρόνη εργασίας και απασχόλησης και συμφιλίωση, σύγκληση ιδιωτικής ζωής και επαγγελματικής ζωής για τους πολίτες, δεξιότητες και κατάρτιση, τονίστηκε αυτό, είναι πολύ σημαντικό θέμα για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και οι εταιρείε είναι μόνο ανταγωνιστικές αν έχουν ικανό και ε, κατάλληλα καταρτισμένο και με κίνητρα εργαζόμενο προσωπικό. Βλέποντας τις βέλτιστες πρακτικές στις εταιρείε, αυτό που κάνουμε είναι μια πρώτη ανάλυση της επισκόπησης ευρωπαϊκών εταιριών, επιτόπου, field survey, ε, φέτος. Και σε σχέση με τα όσα θα ε, έχουμε συμπεράσματα, στις 26 Δεκεμβρίου θα έχουμε παρουσίαση. Έχουμε τις πρακτικές και την τις ε, πολιτικές HR, συμμετοχή εργαζομένων, κοινωνικό διάλογο. Προσπαθούμε μέσα σε αυτό το πλαίσιο να δούμε ε, ποιου είδους win-win ε, συμφωνίες, δηλαδή εποφελείς για όλους τους εμπλεκόμενους και συμβαλόμενους μπορούν να λειτουργήσουν ώστε να υπάρχει αηφορία και να υπάρξουν κίνητρα για τους εργαζόμενους να είναι πιο παραγωγικοί. Να βοηθήσουμε λοιπόν να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα των εταιριών και της οικονομίας μας. Αληθεύει ότι οι εταιρείε είναι εκείνες που πρέπει με αυτόν τον τρόπο να μπορούν να δημιουργήσουν απασχόληση. Και η ανεργία είναι η μεγαλύτερη πιθανότητα πρόκληση που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση φυσικά. Πρέπει να δούμε τι αλλάζει στην αγορά εργασίας. Και κυρίως κάνουμε την έρευνά μας υπό την αιγίδα <clears throat> του οργάνου παρατήρησης και εποπτείας των αλλαγών και ε, παρακολουθώντας συγκεκριμένες ομάδες που την χάνουν ιδιαίτερης προσοχής ως ομάδες στόχοι. Έχουμε κάποια εξειδικευμένα εργαλεία και μέσα, βλέποντας και εξετάζοντας πώς αλλάζει στη σύνθεσή του το σώμα των εργαζομένων και έχουμε μεγάλης κλίμακας ε, ε, ε, έρευνες όπου βλέπουμε πόσα και με ποιο αποτέλεσμα δημιουργούνται θέσεις απασχόλησης ή από την άλλη πλευρά πόσα μπορούν αυτές να απολεστούν. Και δίνουμε και περισσότερα πράγματα, δίνουμε και παραδείγματα μέτρων υποστήριξης που μπορούν να βοηθήσουν τους πολιτικούς να αντιμετωπίσουν τις αλλαγές και μεταβολές αυτές και τις δομές που αναφύονται. Και έχουμε μια ολόκληρη σειρά μέσων υποστηρικτικών και μέσα από αυτά <clears throat> έχουμε και τους κοινωνικούς εταίρους που είναι οι κύριοι εμπλεκόμενοι εδώ σε αυτό το πεδίο και που έχουν ιδιαίτερη σπουδαιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι πολύ σημαντική και για την δομή την οποία υιοθετούμε. Η εταιρική σχέση για την διαβούλευση έχει τεράστια σημασία σε μια αναζήτηση παραγωγικών λύσεων ο κοινωνικός διάλογος κατοχυρώνεται και στις συνθήκες και είναι ένας πυλώνας, ένας κύριος άξονας αυτού του ευρωπαϊκού κοινωνικού προτύπου όπως το αποκαλούμε. Τελευταία μου παρατήρηση αφορά την βελτίωση των συνθήκων διαβίωσης και την κοινωνική συνοχή επίσης που βρίσκονται στον πυρήνα, στην καρδιά των ευρωπαϊκών πολιτικών και του ευρωπαϊκού κοινωνικού προτύπου. Αν θέλουμε πάλι εδώ να διασυνδέσουμε όλα αυτά με την ανταγωνιστικότητα πρέπει να δούμε τι είναι σημαντικό για τα άτομα που μπορεί να είναι διαφορετικό για τον έναν ή άλλο. Πρέπει να δούμε όμως ε, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε και εποπτεύουμε αυτά με την Ευρωπαϊκή Επισκόπηση και στοιχεία που συλλέγουμε μεταξύ αυτών τον ρόλο των ε, κρατικών υπηρεσιών δημόσιων υπηρεσιών και θεσμών που διαδραματίζουν ένα σημαντικό ρόλο για το ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο. Η αλήθεια είναι ότι κοινωνικά αυξάνονται οι ανάγκες και η ζήτηση αυτών των υπηρεσιών. Σε μια περίοδο κρίσης φυσικά αλλάζουν οι αγορές εργασίες και ενώ η ζήτηση αυξάνεται ίσως δεν υπάρχουν οι αναγκαίοι διαθέσιμοι πόροι για να ανταποκριθούμε σε αυτή την αύξηση ζήτησης. Καλούνται να αντιμετωπίσουν την πρόκληση οι κυβερνήσεις και οι πολιτικοί ώστε μέσω περιορισμένων κονδυλίων να υπάρξει αποτελεσματική δράση, ταυτοποίηση και εντοπισμό ευφυών τρόπων για να είμαστε αποτελεσματικοί. Σε ένα συνδυασμό <clears throat> ιδιωτικών και κρατικών ή δημοσίων συμπράξεων, ΣΔΙΤ, χωρίς να υποβαθμίζεται ή να υπάρχει επιδίνωση ε, όρων. Εξετάζουμε κάποια παραδείγματα στον τομέα, για παράδειγμα της περίθαλψης της μέρημνας των παιδιών από πλευράς ε, οικογενειών ε, και γονέων παρέχοντας παραδείγματα βλέποντας πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τα πράγματα με τα κονδύλια που έχουμε στη διάθεσή μας και να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Πριν από δύο εβδομάδες ε, και ολοκληρώνω έτσι είχαμε μια έκθεση για ε, ε, την εξέλιξη των, ε, της ζήτησης που υπάρχει και το δυναμικό σε ένα τομέα που υπάρχει και είναι δεδομένη η ζήτηση και αν δράσουμε σωστά με τον κατάλληλο τρόπο μπορούμε να υποστηρίξουμε και να δράσουμε αποτελεσματικά συνδυάζοντας την αντιμετώπιση κοινωνικών αναγκών και την κάλυψη κοινωνικών αναγκών δίνοντας προώθηση σε δυνατότητες τομέων να αυξήσουν την προσφορά εργασίας την δυνατότητα απασχόλησης. Θα ολοκληρώσω λέγοντας απλά ότι η δέσμευση για την κοινωνική Ευρώπη είναι ο όρος ε, ώστε η κοινωνία των πολιτών ε, να διασφαλίζει όχι μόνο μια αναβαθμισμένη ποιότητα ζωής αλλά και την προοπτική να είμαστε πιο αποτελεσματικοί σε ένα παγκοσμιοποιημένο κόσμο. Καλύτερες συνθήκες διαβίωσης και εργασίας που μπορούν να συνεισφέρουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας λοιπόν. Ευχαριστώ. Merci beaucoup. Euh, Σας ευχαριστώ πολύ. Και έτσι φτάνουμε στην Κρίστα Σέντλατσεκ. Το λέω καλά. Πρόεδρος του οργανισμού ΩΣΑ για την ασφάλεια και υγιεινή στον χώρο εργασίας. Θα μας μιλήσει ακριβώς για αυτό το θέμα, δηλαδή κατά πόσο ένας πιο ασφαλής χώρος εργασίας, όπου η ασφάλεια των εργαζομένων είναι πραγματικότητα, οδηγεί σε περισσότερη ανταγωνιστικότητα. Έχετε το λόγο 10 λεπτά, ε, μην κάνετε όπως ο προηγούμενος. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να έρθω και να σας παρουσιάσω αυτό που εγώ ως ε, πρόσωπος διευθυντής του Οργανισμού για τα Ασφάλεια και Υγιεινή στον χώρο εργασίας θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Ποια επιχειρήματα δηλαδή έχουμε για να υποστηρίξουμε ότι υπάρχει άρρηκτη σχέση ανάμεσα στην υγιεινή και την ασφάλεια όρους εργασίας και την ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν που αντιλαμβάνεστε την σχέση αυτή και αυτό φάνηκε με το ψήφισμα που εγκρίθηκε στην Ολομέλειά σας που στηρίζει την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Ασφάλεια και Υγιεινή στον χώρο εργασίας. Το... Για να ετοιμαστεί το ψήφισμα αυτό βέβαια πρωταγωνίστησε η δικιά σας επιτροπή με υποστήριξη βέβαια από όλες τις πλευρές. Τώρα για να το πω, μα, η σχέση ανάμεσα στην ανταγωνιστικότητα και στην καλή υγεία και ασφάλεια στον χώρο εργασίας στοιχειοθετείται πιστικά, απόλυτα. Οι χώρες οι οποίες έχουν πιο υψηλά επίπεδα εργατικών ατυχημάτων είναι λιγότερο ανταγωνιστικές και εκείνες που έχουν χαμηλότερο αριθμό εργατικών ατυχημάτων είναι λιγότερο ανταγωνιστικές. Και δεν μας εκπλήσει αυτό. Εκεί όπου υπάρχουν μεγάλα επίπεδα εργατικών ατυχημάτων, δεν χρησιμοποιούν όσο καλύτερα μπορούν το εργατικό δυναμικό, το εργατικό κεφάλαιο. Για να είναι παραγωγικός ε, ένας εργαζόμενος, το εργατικό μας δυναμικό, πρέπει να αισθάνεται καλά και να μην είναι στο νοσοκομείο ή αναρώνοντας το σπίτι ή και κάτι χειρότερο. Στην Ευρώπη κάθε χρόνο έχουμε 4.000 ε, ατυχήματα στο χώρο εργασίας και 2,8 εκατομμύρια εργαζόμενοι αναγκάζονται να πάρουν άδεια από τρεις μέρες και πάνω εξαιτίας κάποιου τέτοιου εργατικού ατυχήματος. Η συνέπεια είναι 83 εκατομμύρια ημέρες εργασίας που χάνονται κάθε χρόνο. Και είναι πολύ υψηλά αυτά τα επίπεδα, αλλά δεν είναι τίποτα αν συγκρίνουμε τον αριθμό των ημερών εργασίας που χάνονται εξαιτία ασθενειών που συνδέονται με το χώρο εργασίας. Κάπου 370 εκατομμύρια μέρες δηλαδή που χάνονται ετησίως χωρίς να μετράμε και εκείνους οι οποίοι ποτέ δεν θα μπορέσουν να επιστρέψουν στην εργασία τους εξαιτία των σοβαρών προβλημάτων υγείας. Οπότε για μένα το πιο σημαντικό, η πιο σημαντική εξέλιξη που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας είναι πρώτον οι αλλαγές που λαμβάνουν χώρο στο εργατικό δυναμικό και δεύτερον οι αλλαγές που λαμβάνουν χώρο στους χώρους εργασίας σήμερα. Αν δούμε πρώτα απ' όλα το εργατικό δυναμικό, όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχει μεγαλύτερη ποικιλομορφία και ότι αυξάνει ο μέσος όρος ηλικίας του εργατικού μας δυναμικού. Πράγματι, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει δημοσιεύσει έκθεση σχετικά με βάλωτες ομάδες και έχει ζητήσει να λάβει χώρα ένα μεγάλο πιλωτικό πρόγραμμα για πιο μεγάλους στην ηλικία εργαζόμενους, κάτι το οποίο εμείς εκπονούμε σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και σε συνεργασία με το Eurofound. Οι πιο σε ηλικία εργαζόμενοι είναι πιο πιθανό να έχουν ε, μεγαλύτερα προβλήματα υγείας, δεν οφείλεται αυτό μόνο στην ηλικία, αλλά και επειδή έχουν περάσει περισσότερο χρόνο στους χώρους εργασίας, άρα έχουν εκτεθεί σε μεγαλύτερους κινδύνους από τους πιο νέους. Όσον αφορά την έκθεση αυτή, τι διαπιστώνουμε. Όσο μεγαλώνει ο τριτογενής τομέας, διαπιστώνουμε περισσότερες μειοσκελετικές διαταραχές, ιδιαίτερα στην πλάτη ή ακόμα και ψυχοκοινωνικές διαταραχές, όπως το στρες. Από πλευράς ανταγωνιστικότητας είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι οι περισσότερες από τις απουσίες τους χώρους εργασίας οφείλονται σε μειοσκελετικές διαταραχές και ότι οι πιο μακρές απουσίες έχουν να κάνουν με ψυχικές ασθένειες όπως είναι η κατάθλιψη, το άγχος ή η υπερκόπωση. Αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τους στόχους της Ευρώπης 2020, να έχουμε 5% απασχόληση στις ηλικίες 20 με 64, τώρα πρέπει να δράσουμε. Να μην αφήνουμε πια τον κόσμο να εγκαταλείπει την αγορά εργασίας πριν φτάσει στην ηλικία συνταξιδότησης. Ιδιαίτερα πρέπει να επικεντρωθούμε, και το ακούσαμε και πριν αυτό, στους σημερινούς νέους εργαζόμενους, γιατί αυτοί είναι οι μεγαλύτερη ηλικία εργαζόμενοι του αύριο. Αν θέλουμε να προλάβουμε μακροχρόνια προβλήματα πρέπει να ενισχύσουμε τις προληπτικές μας προσπάθειες σε αυτήν την κατηγορία εργαζόμενων, στους νέους δηλαδή. Η οικονομική κρίση βέβαια μας δυσκολεύει τη ζωή και βλέπουμε ότι πολλές από τις νέες θέσεις απασχόλησης είναι πολύ διαφορετικές από τις παλιότερες και χαρακτηρίζονται από προσωρινές συμβάσεις, από βεβαιότητα στις ώρες εργασίας, από υψηλότερη ένταση εργασίας και άλλα μειονεκτήματα όπως για παράδειγμα δεν επιτρέπουν κατάρτιση κλπ. Αυτά τα χαρακτηριστικά λοιπόν συνδέονται και με υψηλότερα επίπεδα απουσιών που οφείλονται σε λόγους υγείας. Και επιπλέον βλέπουμε όλο και περισσότερο νέους αλλά και μετανάστες εργαζόμενους να δέχονται θέσεις απασχόλησης όπου οι προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας είναι πάρα πολύ χαμηλές. Πρόκειται για μια πίεση η οποία οφείλεται από τα υψηλά επίπεδα ανεργίας των νέων που αντιμετωπίζουμε σήμερα στην Ευρώπη. Τα ακούσαμε αυτά και πριν. Για να πετύχει η Ευρώπη 75% απασχόληση, πρέπει επίσης να αυξήσουμε και την απασχόληση των γυναικών. Πάλι και εδώ, οι πολιτικές υγιεινής και ασφάλειας έχουν να παίξουν σημαντικό ρόλο. Μένει δρόμος ακόμα να κάνουμε. Διαπιστώνουμε ότι πολλές γυναίκες έχουν μερική απασχόληση ή προσωρινή με λιγότερες δυνατότητες κατάρτισης, με χαμηλότερους μισθούς και σε ορισμένες περιπτώσεις ασχολούνται με το καθάρισμα ή με το να προσέχουν ηλικιωμένους και δεν συνοδεύεται η απασχόληση αυτή από προληπτικές υπηρεσίες, πρόληψης δηλαδή, ή από επιθεώρηση εργασίας ή από ασφαλιστική κάλυψη. Οι μικρομεσαίες τώρα επιχειρήσεις, ιδιαίτερα, ιδιαίτερα μικρές, είναι πάρα πολύ σημαντικές για την ευρωπαϊκή οικονομία. Έχουν χτυπηθεί βέβαια πολύ από την κρίση και υπάρχουν χώρες που υποφέρουν περισσότερο πολιτότητα, όπου εκεί πραγματικά τα νούμερα είναι φοβερά. Αυτό μας βάζει μπροστά σε νέες προκλήσεις. Ξέρουμε ότι οι εργαζόμενοι κινδυνεύουν περισσότερο από εργατικά ατυχήματα ή ασθένειες που έχουν να κάνουν ε, με την εργασία εφόσον εργάζονται σε πολύ μικρές επιχειρήσεις σε σχέση με πιο μεγάλες. Οι μελέτες μας τι έχουν δείξει. Έχουν δείξει πως οι μικρές επιχειρήσεις είναι λιγότερο ενημερωμένες και κάνουν λιγότερα πράγματα, δίνουν λιγότερα χρήματα για να φροντίσουν για την ασφάλεια και την υγιεινή στο χώρο εργασίας. Και είναι πιο πολύ ευάλωτες χωρίς να το γνωρίζουν και χωρίς να γνωρίζουν τις επιπτώσεις της επιχειρήσεις τους. Υπάρχουν ε, πολλές εμπειρίες πάντως στις χώρες μέλη που ο οργανισμός μας έχει φροντίσει να διαδώσει για να πείσουμε τις μικρές αυτές επιχειρήσεις ότι η επένδυσή τους στην υγεία και την ασφάλεια κάνει καλό στην επιχείρησή τους. Και αυτό είναι και το σλόγγαν που έχουμε εμείς, ότι η υγεία και ασφάλεια κάνει καλό στην επιχείρησή σας. Τώρα διαπιστώνουμε ότι πολλές φορές άνθρωποι πιστεύουν ε, πως ε, κάτι τέτοιο επιφέρει μεγάλο άχθος στην επιχείρηση, διοικητικό, οικονομικό κτλ. Αυτό ο σοσιαλισμός όμως δεν ισχύει. Τώρα που μπαίνουμε σε οικονομική ανάπτυξη, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι αυτές που θα προσφέρουν περισσότερες θέσεις απασχόλησης. Η επίπτωση λοιπόν ότι η οικονομική ανάκαμψη, δηλαδή η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα, θα μειωθεί εκτός ε, εάν παραβλέψουμε τα, τις προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας, δεν ισχύει. Και ευτυχώ αυτό έχει γίνει φανερό, διότι πέρα από το όποιο άχθος, η υγεία και η ασφάλεια έχει σαν αποτέλεσμα να ενισχύει την ανταγωνιστικότητα και ο κόσμος αρχίζει να το αντιλαμβάνεται σιγά σιγά. Πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις σήμερα και οι managers με τους οποίους ήρθαμε σε επαφή δεν είναι σε θέση να εκτιμήσουν τι ποσά δίνει η επιχείρησή τους για την ασφάλεια και την υγιεινή στο χώρο εργασίας. Δεν αποτελεί δηλαδή διακριτό μέρος της επένδυσης που κάνουν ε, και στο management. Και βέβαια δεν μας εκπλήσει γιατί είναι αλήθεια ότι ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος για τους κινδύνους στην ε, καθημερινή ζωή της επιχείρησής τους. Τώρα είτε πρόκειται για συμβουλευτικό ρόλο ή για λύσεις όπως είναι η online αξιολόγηση κινδύνου που προφέρει ο οργανισμός μας, γι' αυτό πρέπει να ενημερωθεί ο κόσμος. Αυτό το online εργαλείο αξιολόγηση κινδύνου είναι μια πρωτοβουλία που έχει αναπτυχθεί σε εθνικό επίπεδο στις κάτω χώρες συγκεκριμένες και που έχουμε μοιραστεί και με άλλες χώρες. Τέλος όμως, θέλω να σας πω ότι στα τέλη της χρονιάς αυτής και μετά από μια αναθεώρηση των μεθοδολογιών που χρησιμοποιούνται σε διάφορες χώρες, ο ΩΣΑ θα ξεκινήσει ένα πρόγραμμα για την εκτίμηση του κόστους των επιχειρήσεων σε σχέση με την ε, μη κάλυψη ψηλών προδιαγραφών υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Βάσει των ε, μελετών που είχαμε μέχρι τώρα διαπιστώνουμε ότι υπάρχει ένα ποσοστό του ΑΕΠ 3 με 4% που θα ενισχυθεί εφόσον τηρούνται οι προδιαγραφές αυτές. Άρα ενισχύεται η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα. Πάντως, νομίζω ότι αξίζει τον κόπο εδώ να πούμε ότι ενώ μέρο του κόστους, όπως είναι η μείωση στην παραγωγικότητα, η... το διοικητικό άκθος κτλ. μπορούμε να τα εκφράσουμε ποσοτικά. Υπάρχουν όμως και άλλοι παράγοντες που δεν μπορούμε να εκφράσουμε ποσοτικά, όπως είναι ο πόνος, ο θάνατος, η αναπηρία ενός φίλου, ενός συγγενούς, ενός συναδέρφου, το ότι σταματάει την καριέρα του πρόωρα, όλα αυτά πώς να τα μετρήσει κανείς ποσοτικά. Με δύο λόγια. Καταλήγω λέγοντας το εξή. Αναγνωρίζουμε ότι η ανταγωνιστικότητα είναι ακριβώς ο λόγος για τον οποίο πρέπει να διασφαλίζουμε την υγιεινή και την ασφάλεια στον χώρο εργασίας αλλά είναι και ο λόγος για τον οποίο πρέπει να τονίσουμε ότι ακριβώς η γενική ασφάλεια στον χώρο εργασίας βοηθάει τους άντρες και τις γυναίκες, νέους και μεγαλύτερους, να μείνουν στους χώρους εργασίας τους περισσότερο και όχι να τους εγκαταλείψουν πρόωρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Αυτά τα χειροκροτήματα δείχνουν πόσο πολύ είχαν απήχηση όλα αυτά που είπατε στα μέλη της Επιτροπής μας. Και τα θέματα, και όχι μόνο αυτά που είπατε, αλλά γενικά τα θέματα που συζητάνε όλοι οι ομιλητές μας. Η τελευταία ομιλήτρια σε αυτό το πάνελ προέρχεται από το Ίδρυμα, Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Κατάρτισης, η Μάρλεν Σέρμπαν που θα μας μιλήσει για τη σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις γειτονικέ χώρες ε, σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη πολιτικών καινοτόμων για το ανθρώπινο δυναμικό. Μια πολιτική που θα είναι κερδοφόρα και για μας αλλά και για τις γειτονικέ χώρες. Η διευθύντρια του Ιδρύματος αυτού ε, είναι εδώ μαζί μας. Σας ευχαριστώ όχι μόνο γιατί μου δίνετε το λόγο, αλλά και για όλες τις προσπάθειες που κάνει η Επιτροπή Απασχόλησης για να οργανώσει τη σημερινή ακρόαση. Σήμερα έχουμε τη δυνατότητα να παρουσιάσουμε στα μέλη σας και στη γραμματεία τις ανησυχίες μας και τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων μας. Τώρα θα περάσω στα αγγλικά για να σας μιλήσω για την παγκόσμια Ευρώπη. Δεν θα μιλήσω για την γραμμή του προπολογισμού από την οποία χρηματοδοτείται το Ίδρυμά μου, παρότι μιλάω εδώ στο αρμόδιο όργανο για τον προπολογισμό, θέλω να μιλήσω για την αποστολή του Ιδρυματός μου που δημιουργήθηκε για να υποστηρίξει την παγκόσμια εικόνα της Ευρώπης και το πώς θα χρησιμοποιήσει αυτή η Ευρώπη το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο ως μηχανισμό ανταγωνιστικότητας. Ε, ο Ζακ Ντελόρ αναφέρθηκε στη δεκαετία του 90 στο ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο λέγοντας ότι η οικονομική πρόοδος θα πρέπει να πηγαίνει παράλληλα με την κοινωνική πρόοδο. Και η οικονομική ανάπτυξη, επομένω θα πρέπει να παντρεύεται με την κοινωνική συνοχή. Σήμερα, μετά την κρίση, θα πρέπει να ξαναδούμε λίγο τις απόψεις που είχαμε στο παρελθόν και να αναρωτηθούμε αν αυτή η παράλληλη πορεία ανάπτυξης είναι εφικτή και αν το μοντέλο ανταγωνιστικότητάς μας ε, προσαρμοζόταν στις ανάγκες των λαών μας που είναι στην καρδιά των ε, πολιτικών κοινωνικής ε, συνοχής. Όταν μιλάμε για την παγκόσμια Ευρώπη, σήμερα στον 21ο αιώνα, πρέπει να σκεφτούμε ότι είναι μια εποχή ε, που σημαδεύεται από τις παγκόσμιες επικοινωνίες. Οι άνθρωποι, το κεφάλαιο, οι πληροφορίες, τα αγαθά, όλα ρέουν, περνάνε τα σύνορα με μεγαλύτερους ρυθμούς και η Ευρώπη δεν είναι πια μόνη της. Εάν θέλει να γίνει ανταγωνιστική ξανά και να παραμείνει ανταγωνιστική, θα πρέπει να στρέψει το βλέμμα προς τους γειτονές της. Και ο τρόπος που κοιτάζει η Ευρώπη τους ε, γείτονές της είναι ένα, ένας δίκαιος τρόπος. Γιατί δεν τους επιβάλλει τι θα κάνουν, αλλά παρουσιάζει τις δικές της πολιτικές για να σκεφτούν αν μπορούν να εμπνευστούν από αυτά που συμβαίνουν εδώ στην Ευρώπη. Θα σας εξηγήσω λοιπόν γιατί εμείς, η δική μου υπηρεσία, συνεργάζεται με τις, με υπηρεσίες και οργανισμούς που λάβατε, που ακούσατε προηγουμένως. Γιατί όλες αυτές ασχολούνται με την υγεία στην εργασία, με την κατάρτιση, με την εκπαίδευση. Ε, και το ερώτημα είναι, από τη δουλειά μας εμπνέονται οι γειτονικέ χώρες. Πιστεύω πως ναι. Επίσης ε, θα έχουμε εδώ έναν εκπρόσωπο από τη Μολδαβία, ε, ο οποίος ε, είναι αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργό Οικονομικών. Θα μιλήσει για θέματα που αφορούν την ανταγωνιστικότητα και βεβαίως σε κάποιο βαθμό η Ευρώπη μπορεί να επηρεάσει τα τεκτενόμενα στη χώρα αυτή, τη Μολδαβία. Και ο κύριος αυτός είναι ο Βαλέριου Λάζαρ. Σε αυτόν τον διασυνδεδεμένο κόσμο κυκλοφορούν τα πάντα. Άνθρωποι, αγαθά, κεφάλαια, πληροφορίες. Ε, πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ένα νέο μοντέλο ανταγωνιστικότητας. Και δεν νομίζω ότι αυτό το μοντέλο ε, έχει μια μονοκόμματη λύση για όλα και για όλους. Επίσης πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ε, τα νέα μοντέλα κινητικότητας και μετανάστευσης στη χώρα μας ποιος θα γίνει ανταγωνιστικός. Ο πολίτης, η κοινότητα, η χώρα, η Ήπειρος, ο πλανήτης, ποιος είναι ανταγωνιστικός. Και αυτές τις νέες προσκλήσεις πρέπει να τις λάβουμε υπόψη μας για να διαμορφώσουμε και να βρούμε τις ε, νέες λύσεις για την ανάπτυξη ο οργανισμός μου θα ήθελα να σας προτείνει κάποια στοιχεία τα οποία συνδέονται με τις ε, ικανότητες, με τις δεξιότητες, με τα προσόντα. Γιατί κατά την άποψή μας για να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί είναι απαραίτητη προϋπόθεση να έχουμε τα απαραίτητα προσόντα, το απαραίτητο μείγμα προσόντων δεξιοτήτων για να είμαστε απασχολήσιμοι, για να βρούμε μια δουλειά και επομένως για να συνεισφέρουμε έτσι στην ανταγωνιστικότητα. Αν θεωρήσουμε ότι οι δουλειές δημιουργούνται, ότι οι θέσεις απασχόλησης δημιουργούνται, πιστεύουμε ότι η εκπαίδευση και η κατάρτιση δεν θα πρέπει να αντιδρούν απλώς στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Πιστεύουμε ότι η εκπαίδευση και η κατάρτιση θα πρέπει να δημιουργήσουν αυτούς που διαμορφώνουν τις α, θέσεις απασχόλησης. Και θα πρέπει να είναι σε θέση, όπως είπε ο συναδελφός μου, ε, να είναι σε θέση να προβλέψει τι προσόντα χρειάζονται. Οι δουλειές που δημιουργούνται το 2010 Κάποιες από αυτές ε, είναι εντελώ καινούργιες και δεν ήταν γνωστές όταν ε, κάποια από το σημερινό εργατικό δυναμικό πήγαινε σχολείο το 2004 ας πούμε κτλ. Επομένως, μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει και οι επιχειρηματίες να είναι έτοιμα τις λύσεις είμαι επιχειρηματίας, τι σημαίνει. Ότι δημιουργώ μια επιχείρηση, αλλά και προσαρμόζομαι στις αγορές και στις προϋποθέσεις ε, του μέλλοντος ό,τι αφορά τον κόσμο της εργασίας. Εμείς λοιπόν στο εταιρειμά μου το ETF δουλεύουμε με 30 χώρες, συνεργαζόμαστε με 30 χώρες για να λάβουμε υπόψη μας τις ανάγκες που πρέπει να λάβουν αυτοί που διαμορφώνουν τις, τις πολιτικές, τις προτεραιότητες και τις λύσεις σε επίπεδο πολιτικής ε, που θα κάνουν τη διαφορά. Όταν αναφέρθηκα στην πρωτοβουλία του Ζακ Ντελόρ προηγουμένως, ήθελα, θέλω να τονίσω ότι είπα ότι η οικονομική ανάπτυξη και η κοινωνική συνοχή συνδέονται και με τη δημοκρατία. Στην Ευρώπη αυτό το θεωρούμε δεδομένο. Αλλά όταν το ETF δουλεύει στις ε, χώρες εταίρους, πάντα θεωρούμε ότι αυτό είναι από τις ε, θεμελιώδες ευρωπαϊκές αξίες. Σκεφτείτε τις πρόσφατες αναταραχές στον αραβικό κόσμο. Δεν πρέπει να σκεφτούμε ότι, να ξεχνάμε ότι η αραβική άνοιξη οφείλεται εν μέρη στην ανισότητα, στην έλλειψη προοπτικής στο γεγονός ότι η ανταγωνιστικότητα και η επιτυχία περιορίζεται για μια μικρή ομάδα ανθρώπων σε αυτές τις χώρες. Επομένως, θεωρούμε ότι το οικονομικό στοιχείο και το κοινωνικό στοιχείο όταν συμπορεύονται μπορούν να βοηθηθούν ε, όλες οι χώρες και κυρίως και οι χώρες βεβαίως εν προκειμένου της Αραβικής Άνοιξης. Επίσης υπάρχουν άλλες χώρες, οι χώρες ας πούμε που ξεκίνησαν, ξεκίνησε η δημοκρατία. Ε, δημοκρατία τι σημαίνει, συνεργασία. Ποιο λοιπόν ε, έχει τα ενία, μόνο το κράτο, Όχι. Θα πρέπει να υπάρχει διάλογος. Δεν αρκεί μόνο ο διάλογος όμως. Θα πρέπει να δώσει εξουσία στου εταίρου σου για να είναι σε θέση να συνομιλήσουν σαν ίσως προς ίσο με την κυβέρνηση. Αυτή τη δουλειά κάνουμε στο ETF. Προσπαθούμε να οικοδομήσουμε αυτό το, δυναμικό όχι μόνο για τους προσώπους των κυβερνήσεων αλλά και για τους κοινωνικούς εταίρους και να εξασφαλίσουμε ότι είναι ένας πραγματικός και αποτελεσματικός εταίρος και ότι ο διάλογος είναι πραγματικός για θέματα εκπαίδευσης και κατάρτισης. Πιστεύουμε ότι η εταιρική σχέση πρέπει να αφορά ε, τους ε, παρόχους ε, και τις επιχειρήσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης. Όπως φαίνεται από τις ευρωπαϊκές πολιτικές, οι επιχειρήσεις και ο ιδιωτικός τομέας και αυτοί πρέπει να μπουν στην εξίσωση. Αυτά ήθελα να σας πω και είμαι πραγματικά ε, ευγνώμων προς τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Μολδαβίας που δέχτηκε την πρόσκληση για να μας πει τις απόψεις του για αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ και τους τέσσερις οργανισμούς. Αυτή την ιδέα, κάθε χρόνο δηλαδή να συναντιόμαστε και ότι αυτό μας επιτρέπει έτσι να συζητάμε ένα κοινωνικό στόχο όλοι μαζί, το θεωρώ πάρα πολύ θετικό. Δεν άκουσα βέβαια όλες τις παρουσιάσεις, αλλά αυτό δείχνει πόσο σημαντική είναι αυτή η συνάντηση, ώστε να ενισχυόμαστε στην αποστολή μας. Τώρα, είναι μεγάλη τιμή για μένα να ανοίξω την συζήτηση. Θα αρχίσω από τον εξέχοντα προσκεκλημένο μας, τον κύριο Βαλεριού Λαζάρ, που είναι ο υπουργό και Υπουργό Οικονομικών της Μολδαβίας. Έχουμε δύο ερωτήσει για αυτήν την συζήτηση. Προσπαθούμε λοιπόν να αναλύσουμε τα θέματα που θίξαμε σήμερα το πρωί και θα σας διαβάσω στα αγγλικά τις ε, ερωτήσεις. Πρώτα απ' όλα διάκριση. Δέκα λεπτά θα έχει ο πρώτος μας ομιλητής και οι άλλοι θα έχουν έξι λεπτά. Τι να κάνουμε δεν βλέπω να επαναστατείτε, οπότε γίνεται αποδεκτή η πρότασή μου αυτή. Λοιπόν, ποιο είναι το θέμα. Το θέμα είναι ότι βρισκόμαστε μέσα σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία. Και έχουμε και άλλους γίγαντες απέναντί μας. Μια ισχυρή οικονομία και κοινωνική Ευρώπη είναι κάτι πιο σημαντικό από ποτέ. Πρώτη ερώτηση λοιπόν, το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο. Πώς πρέπει να εξελιχθεί για να διατηρηθεί Ποιος είναι ο ρόλος του κοινωνικού διαλόγου. Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση. Και η δεύτερη, που είναι στο εξή πλαίσιο, η οικονομική κρίση και οι δημογραφικές προκλήσεις ε, βαραίνουν πολύ στην ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα. Τα πρόσφατα χρόνια η συζήτηση έχει επικεντρωθεί στο πώς μπορεί να συνεισφέρει το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο ώστε να οδηγηθούμε σε μια σχέση win-win ανάμεσα σε επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους. Και η ερώτηση είναι η εξής. Τι νέους καινοτόμους τρόπους εργασίας και κατάρτισης μπορούν να συνεισφέρουν στην βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα. Αγαπητέ Ανεπληρωτή Πρωθυπουργέ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω ρουμάνικα, λέει ο μιλητής. Σας ευχαριστώ λοιπόν. Σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας και ευχαριστώ όλους τους συναδέρφους και από το εθνικό και... Ήθελα να ευχαριστήσω τους προλαλήσαντες και να πω ότι όλα όσα αναφέρατε είναι πολύ χρήσιμα και επίκαιρα. Σήμερα, 25 <clears throat> Σεπτεμβρίου, έχουν περάσει και ολοκληρώνονται τέσσερα χρόνια κυρίες και κύριοι από τότε που ανέλαβα το αξίωμα του Υπουργού Οικονομικών. Από τότε που το ανέλαβα και εισήχθη ε, αυτή η πρακτική, η κυβερνητική πρακτική στην οποία συμμετέχω είναι ο συνασπισμός για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση στη χώρα μας μετά από τα πολλά χρόνια κομμουνιστικής ηγεσία και διακυβέρνηση στη χώρα μας. Τέσσερα χρόνια εργαστήκαμε έντονα, αναζητήσαμε σωστές λύσεις, τις πιο ουσιώδεις και σωστές λύσεις. Γι' αυτό τονίζω για άλλη μια φορά ότι το να παρευρίσκομαι εδώ σήμερα είναι πολύ σημαντική υπόθεση για μένα και για μας. Έτσι μπορούμε να συνεισφέρουμε από πλευράς μας ε, ώστε η δημοκρατία της Μολδαβίας να αναμορφωθεί και να μετασχηματιστεί. Κάνουμε λόγο για ένα κοινωνικό πρότυπο το οποίο συνδέεται με το οικονομικό πρότυπο και γι' αυτό κάνω λόγο για το οικονομικό κοινωνικό πρότυπο στο οποίο θέλουμε, το οποίο θέλουμε να προσεγγίσουμε εμείς ως Μολδαβοί και να το αφομοιώσουμε. Όσον αφορά τις ευρωπαϊκές αξίες μπορούμε να τονίσουμε ότι οι ευρωπαϊκές αρχές και αξίες ε, είναι πολύ σημαντικές. Ε, η δημοκρατία, ένα ισχυρό οικονομικό και κοινωνικό πρότυπο που μπορεί να οδηγήσει στα ευκταία αποτελέσματα και στόχους για μας, για μας τους πολιτικούς ε, που είμαστε υπεύθυνοι για την διαμόρφωση της πολιτικής ζωής της χώρας μας και έτσι μπορούμε να συνεισφέρουμε στην αηφορία, στην ανάπτυξη της χώρας μας. Αυτό ισχύει και για άλλες χώρες, όχι μόνο για τη δημοκρατία της Μολδαβίας. 23 χρόνια από τότε που αποκτήσαμε την ανεξαρτησία μας ως χώρα, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι πρέπει να αλλάξει το πρότυπο το οποίο ακολουθούμε στη Μολδαβία η περίπτωση της δημοκρατίας της Μολδαβίας μπορεί να είναι ένα πολύ θετικό παράδειγμα πώς μπορούν τα πράγματα να αλλάξουν και να τροποποιηθούν. Είχαμε ένα κοινωνικό και οικονομικό πρότυπο κατά το παρελθόν σε μια ελληματική και κολοβή δημοκρατία. Δεν ήταν καθόλου θετικό το οικονομικό κλίμα. Δεν μπορούσαμε να προσελκύσουμε ε, επενδύσεις. Δεν μπορούσε να επιτευχθεί κάποια ανάπτυξη με αυτό το πρότυπο. Οδήγησε μόνο στην αποψήλωση του πληθυσμού μας και την μετανάστευση στο εξωτερικό. Με αυτόν τον τρόπο δεν μπορεί με κανένα τρόπο να διακυβερνηθεί μια χώρα. Και το 2009 η δημοκρατία της Μολδαβίας ουσιαστικά βρισκόταν στην πρώτη θέση. Στην πρώτη θέση όσον αφορά το ΑΕΠ και μόνο το Τατζικιστάν ήταν μετά κάτω από μας τελευταίο. Δεν είμαστε λοιπόν μια χώρα εξαγωγών, ούτε, είμαστε, ούτε είχαμε παραγωγή ανταγωνιστικών προϊόντων. Εξάγαμε ανθρώπους, ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο ισχύει ακόμα και σήμερα σε έντονο βαθμό. Ένα τρίτο των κατοίκων μας, των πολιτών μας, βρίσκονται στο εξωτερικό και εκεί εργάζονται δραστηριοποιούνται σε χώρες όπου πολλές φορές ε, τα δικαιώματά τους ε, δεν ε, είναι σεβαστά και δεν διασφαλίζονται. Γι' αυτό καταλήξαμε λοιπόν εμείς στο συμπέρασμα ότι είναι ανάγκη να αλλάξει το πρότυπο το οποίο υπάρχει στη χώρα μας και να αλλάξουμε την εξέλιξη και τα τεκτενόμενα στη χώρα μας. Να κινηθούμε προς ένα πρότυπο λειτουργούσας, λειτουργικής δημοκρατίας. Χρειαζόμαστε όρους και προϋποθέσεις για ένα πιο θετικό περίγυρο και μια πιο θετική ατμόσφαιρα για τους ε, <clears throat> επενδυτές ώστε να μην εξάγουμε ανθρώπινο δυναμικό, εργατικά χέρια αλλά να μπορέσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί. Σε αυτό εδράζεται η φιλοσοφία μας, η φιλοσοφική προσέγγιση μας ε, για την πολιτική μας ζωή. Έχουμε μέχρι το 2020 εγκρίνει ένα κοινοβουλευτικό πρόγραμμα από το κοινοβούλιο μας. Έχουμε χρησιμοποιήσει τον δικό σας χρονορίζοντα 2020 από πλευρά του Ευρωκοινοβουλίου. Επηρεαστήκαμε από τις δικές σας προσεγγίσεις στην Ευρώπη για αυτά τα θέματα και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι η σημαντικότερη προτεραιότητα από τις 7 κύριες προτεραιότητες μας είναι η πολιτική εκπαίδευση και η παιδεία. Αυτό ισχύει για εκείνε τι χώρες στι οποίες ανήκει και η δημοκρατία της Μολδαβία, όπου οι φυσικοί πόροι δεν είναι απεριόριστοι, είναι περιορισμένοι. Έχουμε δύο, ε, ισχυρά, ε, δύο ισχυρές κατηγορίες ε, δυναμικού ανθρώπινο δυναμικό και αρρώσιμες εκτάσεις, γεωργικές εκτάσεις. Έτσι λοιπόν πρέπει σε πρώτο βαθμό να επενδύσουμε στο ανθρώπινο δυναμικό μας. Αυτό είναι μεγάλη ανάγκη, η κύρια ανάγκη μας. Θα πρέπει επίσης να δούμε τι, μπορούν να γίνουν, τι μπορεί να γίνει με τις υποδομές. Επαναλαμβάνω, η σημερινή συζήτηση είναι πολύ χρήσιμη και επικοδομητική. Με αυτά τα κίνητρα και αυτές τις προτάσεις μπορούμε να προσεγγίσουμε ιδέες και προτάσεις για την ανάπτυξη της ίδιας της δικής μας χώρας. Γι' αυτό τα όσα συμβαίνουν στην Ευρώπη και το ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο είναι μια πηγή έμπνευση για μας με όλες τις δυσκολίες που περιγράψατε και συνδέονται με τη διασφάλισή του. Είμαστε ένα πολιτιστικό και πολιτισμικό πρότυπο, ένα πρότυπο κοινωνικό, πολιτιστικό και πολιτισμικό ε, το πρότυπο της Ευρώπης είναι πολύ σημαντικό για μας τα δικά σας διδάγματα και συμπεράσματα να τα λάβουμε υπόψη. Να δούμε τι έχετε συναγάγει εσείς ως συμπεράσματα για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης. Η επένδυση στους ανθρώπους, στο ανθρώπινο δυναμικό είναι το πιο αποτελεσματικό μέσο και εργαλείο. Αυτό κατανόησα από τη σημερινή συζήτηση και αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τη χώρα μας. Το θέμα της, ε, του, χρονικού, του οδικού χάρτη για την ανάπτυξη στη χώρα μας, το ανέφερα, οι επενδύσεις στο ανθρώπινο δυναμικό, η ανταγωνιστικότητα συναρτάται σε μεγάλο βαθμό με μια, από μια συνέργεια μεταξύ επενδύσεων στο ανθρώπινο δυναμικό και επενδύσεων στη βιομηχανία φυσικά. Γιατί κατά τα άλλα δεν ε, μπορούμε να προχωρήσουμε και να διαρρήξουμε τον φαύλο κύκλο στον οποίο βρισκόμαστε. Τι σημαίνουν όλα αυτά. Σημαίνουν ότι οι επιχειρήσεις στο σημερινό οικονομικό πρότυπο δεν μπορούν να προσφέρουν ανταγωνιστικούς μισθούς ε, στους Μολδαβούς. Γι' αυτό οι Μολδαβοί πάνε στο εξωτερικό. Οι ικανοί προσεργασία άνθρωποι, οι πολίτες χρειάζονται ένα θετικό περίγυρο και ικανοποιητικούς μισθούς. Το καλύτερο κοινωνικό πρότυπο για μια χώρα υφίσταται στο ότι εκείνοι οι οποίοι είναι ικανοί προσεργασία πρέπει να μπορούν να έχουν μια ανταγωνιστική θέση εργασίας η οποία θα τους προσφέρεται, στην οποία θα εργάζονται. Αυτή είναι η καλύτερη προστασία των πολιτών. Είναι ο φυσικός στόχος κάθε ανθρώπου, η φυσική του επιθυμία να έχει μια καλή θέση απασχόλησης. Είχαμε κάποια ανάπτυξη στη χώρα μας, αλλά δεν μπορέσαμε να αναπτυχθούμε όπως θα έπρεπε. Διότι ανάπτυξη και αηφορία στην ανάπτυξη δεν είναι φυσικά η εγκατάλειψη της χώρας από τους πολίτες της. Αν η οικονομία δεν μπορεί να προσφέρει ανταγωνιστικούς μισθούς, οι άνθρωποι φεύγουν, εγκαταλείπουν τη χώρα και μεταναστεύουν. Το είπα, ένα τρίτο των ενεργών Μολδαβών πήγαν στο εξωτερικό και εκεί συνεισφέρουν για τη δημιουργία πρόσθετης αξίας. Θα θέλαμε να επιστρέψουν, να μπορέσουν να επιστρέψουν αυτοί οι πολίτες πολίτες μας στη Μολδαβία για να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη της χώρας μας. Επιτρέψτε μου να επανέλθω σε αυτό κυρίε και κύριοι, αυτό το οποίο περιέγραψε η Πρόεδρος. Είναι αυτονόητο ότι υπάρχει παγκοσμιοποίηση και οι διάφορες διαδικασίες και διεργασίες παγκοσμιοποίηση πρέπει να αντιμετωπιστούν. Αυτό οδηγεί στο ότι πρέπει να είμαστε πιο ενεργοί από πλευρά κρατικών αρχών. Και από τη σημερινή συζήτηση και από την επιστημονική βιβλιογραφία μπορεί να δει κανείς ότι η ανταγωνιστικότητα είναι κάτι το οποίο από πλευρά των επιχειρήσεων πρέπει πάντα να ενισχύεται. Από την άλλη πλευρά όμως ξεχνάμε το, τους ανθρώπους. Δεν πρέπει να τους ξεχνάμε τους ανθρώπους. Να αυξάνουμε την ανταγωνιστικότητα με καλύτερη τεχνολογία και βελτιώσει σε αυτήν. Να ξεχνάμε όμως και να απεμπολούμε τους ανθρώπους. Δεν πρέπει να γίνεται αυτό. Και αυτό το οποίο ισχύει στο μικρό επίπεδο, για παράδειγμα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μικρές επιχειρήσεις, συσσωρεύεται στη συνέχεια μέχρι στο ανώτατο επίπεδο και βλέπουμε ποιες είναι οι επιπτώσεις. Γι' αυτό οι αρχές πρέπει να δραστηριοποιηθούν, η κυβέρνηση, οι κυβερνήσεις πρέπει να δραστηριοποιούνται, ώστε οι επιχειρήσεις ε, και η οικονομία να μπορέσει να αυξήσει βέβαια, να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους, να μην ξεχνάμε όμως τους ανθρώπους. Ανταγωνιστικότητα δεν σημαίνει για μας ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, η κυρία Σερβάν έθεσε ένα ερώτημα το οποίο θα ήθελα να απαντήσω. Θέλουμε να είμαστε ως χώρα ανταγωνιστικοί, όχι απλώς να έχουμε μία σε κάποιους τομείς ανταγωνιστική οικονομία. Ως χώρα να είμαστε ανταγωνιστικοί. Είναι το θέμα της επιβίωσης είναι το υπαρξιακό ερώτημα to be or not to be του Hamlet του Shakespeare. Πρέπει να δούμε, θα μπορέσουμε να επιβιώσουμε ή όχι. Αυτό εξαρτάται από την ανταγωνιστικότητά μας. Είμαστε μια μικρή χώρα με περιορισμένους φυσικούς πόρους και πρέπει να αντέξουμε στον ανταγωνισμό και να αποδειχθούμε ανταγωνιστικοί. Είναι σημαντικό λοιπόν για μας κατά τη διάρκεια των συμφωνιών και την προσέγγιση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση να καταφέρουμε να πετύχουμε να προσυπογραφεί αυτή η Συμφωνία Σύνδεσης και Συνεργασίας είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία που μας προσφέρεται, αλλά είναι και μεγάλη πρόκληση που αντιμετωπίζουμε. Διότι όπως ανέφερα, περιορίζεται η ανταγωνιστικότητά μας, είναι περιορισμένη σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Γι' αυτό αυτός ο οδικός χάρτης είναι πολύ σημαντικός για μας, για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς μας. Έτσι μπορούμε να προσαρμοστούμε εμείς ως Δημοκρατία της Μολδαβία στις απαιτήσει αυτής της Συμφωνίας Ελεύθερου Εμπορίου. Το επαναλαμβάνω, είναι ένα πολύ περίπλοκο σύνθετο θέμα η ανταγωνιστικότητα. Ξεπερνά το πλαίσιο το οικονομικό ή το κοινωνικό. Δεν μπορεί να είναι κανείς ανταγωνιστικός αν δεν είναι καινοτόμος και αν δεν ε, εξελίσσεται διαρκώς όσον αφορά την ε, ε, δημιουργική καινοτομία. Και καταλήγω και σε μία άλλη τοποθέτηση. Ισχύει το σύνθημα διαφοροποίηση ή θάνατος ή ε, αποτυχία. Τον 21ο αιώνα πρέπει όμως να το τροποποιήσουμε. Καινοτομία είναι το πιο σημαντικό. Η καινοτομία για τις επιχειρήσεις και για την ε, πολιτική παιδείας και εκπαίδευσης. Θα ήθελα να πω ότι εδώ ε, πρέπει να επενδύσουμε στο ανθρώπινο κεφάλαιο. Δεν είναι τυχαίο ή συμπτωματικό, δεν είναι συγκυρία ότι αυτό το θέσαμε ως επίκεντρο στη στρατηγική μας. Υπό τον τίτλο η συμπτωματικο δεν ειναι συγκυρια οτι αυτο το θεσαμε ως επικεντρο στη στρατηγικη μας υπο τον τιτλο πιο αποτελεσματικές, η πιο αποτελεσματική εκπαίδευση και παιδεία για την, ε, τις ανάγκες ε, της ε, ανάπτυξης και της εργασίας. Πρέπει να προσαρμοστούμε ώστε το σύστημα αυτό και εκπαίδευσης να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις και να αντιμετωπίζει τη ζήτηση. Τη ζήτηση από πλευράς της οικονομίας και της απασχόλησης. Εκεί πρέπει να θέσουμε το κέντρο βάρους και να αναπτύξουμε το έργο μας. Και τέλος θα ήθελα να πω ότι και εδώ πιστεύουμε ότι ο κοινωνικός διάλογος, πιστεύουμε και εμείς, πρέπει να προαχθεί να καλλιεργηθεί. Από κοινού με τα συνδικάτα θα θέλαμε οι εργαζόμενοι να μπορούν να εκπαιδεύονται και να καταρτίζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να επιμορφώνονται διαρκώς και να μπορούν να έχουν καλύτερες προοπτικές για ένα μεγαλύτερο μισθό. Έτσι προσεγγίζω το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Πρότυπο. Θέλω να ριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωκοινοβούλιο και τα τέσσερα όργανα για την συνεργασία. Έχουμε και από πλευρά CTF μια πολύ σημαντική υποστήριξη. Θέλουμε να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε σε όλα αυτά τα τα προγράμματα, ιδιαίτερα στο πλαίσιο της καινοτομίας, της παιδείας και της εκπαίδευσης. Ένας προλαλής σας, ένας από τους προηγούμενους στο πάνελ μίλησε για την αλληλεγγύη. Πολύ σημαντική έννοια η αλληλεγγύη. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να συμμετέχουμε σε αυτά τα σχέδια και προγράμματα, να χρησιμοποιούμε και να εκμεταλλευόμαστε την πραγματογνωμοσύνη, ώστε να μπορούμε έτσι να συνδιαμορφώσουμε το μέλλον μας, αυτό που επιθυμούν οι νέοι. Μια ευρωπαϊκή προοπτική. Ευχαριστώ. Merci beaucoup. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Αντιπρόεδρε της Κυβέρνησης για τη δέσμευσή σας αυτή και για τα λόγια σας, τα οποία βρίσκονται σε απόλυτη συμφωνία με αυτά που μας απασχολούν και μας. Αλλά μας δώσατε ένα κακό παράδειγμα. Ο κύριος Χάιντς Μπέκερ όμως θα δώσει το καλό παράδειγμα και θα τηρήσει το χρόνο του. Έξι λεπτά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Και συνάδελφοι, επιτρέψτε μου να πω, των Ευρωπαϊκών Ιδρυμάτων και Υπηρεσιών και Πρόεδρε. Πρώτα να περιγράψω αν επιτρέπετε κάποια προσωπική, ας το πω έτσι, εμπειρία σε σχέση με το Κοινοβούλιο. Ως μέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και ταυτόχρονα σαν μέλος, ως μέλος της Επιτροπής Πολιτισμού που αντιμετωπίζει καλύπτει τα θέματα παιδείας και εκπαίδευσης για την ημερήσια διάταξη. Όλα τα, αυτά καυτά θέματα για σήμερα και για το μέλλον σίγουρα για επιτυχή ε, επαγγελματική ζωή που θα βασίζεται σε αυτές τις δεξιότητες και ικανότητες ε, όπως απαιτούνται σήμερα είναι το κύριο έργο και στις δύο κοινοβουλευτικές επιτροπές. Θέλω να συνδυάσω λοιπόν και να συνδέσω τις προτάσεις που έγιναν για αυτά τα σημερινά μας θέματα και να συνδέσω αυτά τα δύο ζητήματα, ε, κυρία Πρόεδρε Μπερές, ε, τον κοινωνικό διάλογο για παράδειγμα και τις θέσεις απασχόλησης και την καινοτομία όσον αφορά καινοτόμο δράση να αναφέρω κάποια στοιχεία κλειδιά για την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού κοινωνικού προτύπου υπό τους όρους της εργασίας μας εδώ ώστε να είμαστε ανταγωνιστικοί στην Ευρώπη ώστε να διαδραματίσουμε ένα ρόλο προπομπού, ένα ρόλο πρωτοπόρου ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρώτον, να βελτιστοποιήσουμε και αν επιτρέπετε ας ξεχάσουμε εδώ όλες τις διπλωματικές διατυπώσεις και ας πάμε στο ψαχνό και ας μιλήσουμε για την ίδια την ουσία ως αξία, να βελτιστοποιήσουμε την επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση, ώστε να πετύχουμε αυτό το οποίο πρέπει να τεθεί πάνω-πάνω στην κορυφή, απασχολησιμότητα, δυνατότητα απασχόλησης. Γι' αυτό γνωρίζουμε ότι το διτό, διπλό σύστημα εκπαίδευσης και μαθητείας για τους νέους, αυτό αποκινούμε αυτά τα οποία προαναφέρθηκαν, που οδηγούν στο τρίτο επίπεδο, ανώτατο επίπεδο πανεπιστημιακής εξέλιξης τελικά ως επιστέγασμα, να αυξήσουμε τις δεξιότητες και ικανότητες των ε, ηλικιωμένων στην αγορά εργασίας, βελτιώνοντας τη διαβίου εκπαίδευση με όλες τις δυνατότητες που παρέχονται όσον αφορά ένα, μια εργαλειοθήκη με πολλά εργαλεία στην βέλτιστη ανάπτυξη και χρήση τους και από πλευράς προγραμμάτων ΣΕΝΤΕΦΟΠ για παράδειγμα σχετικά. Ας αναπτύξουμε λοιπόν το καλύτερο σύστημα παγκόσμια, σύστημα εκπαίδευσης και παιδείας. Απλό, το μόνο που χρειάζεται είναι να αποσαφίσουμε τις ανώτατες εκείνες δεξιότητες και ικανότητες που πρέπει να τύχουν της καλύτερης εκπαίδευσης με τους καλύτερους καθηγητές και δασκάλους. Θέλω να τονίσω αυτό, γιατί όλα τα άλλα πράγματα αναφέρθηκαν ή θα έχουν αναφερθεί και αυτό πρέπει να τονιστεί. Για όλα όσα ανέφερα Είμαι βέβαιος ότι χρειάζονται διάφορες και διαφορετικές δομές που πρέπει να διασφαλιστούν. Και εμείς στη δική μας Κοινοβουλευτική Επιτροπή συνειδητοποιούμε ότι πρέπει να προσαρμοστούμε σε όλα αλλά να έχουμε και μια αποτελεσματική κοινωνική εταιρική σχέση. Χωρίς μια τέτοια κοινωνική εταιρική σχέση μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών, χωρίς αυτή τη συμμαχία δεν μπορούμε να είμαστε επιτυχείς στην ε, οικοδόμηση του μέλλοντος που θέλουμε να δημιουργήσουμε, του νέου μέλλοντος. Και ας αναπτύξουμε αποτελεσματικές υπηρεσίες για την αγορά εργασίας. Όλο και μεγαλύτερη σπουδαιότητα έχουν και αποκτούν από ότι σε σχέση με τις τελευταίες δεκαετίες κατά το παρελθόν. Ας συνειδητοποιήσουμε επιτέλους επιπλέον ότι υπάρχει μια σαφέστατη παράμετρος, μια συνιστόσα που συνοδεύει αυτά τα οποία λέμε και κάνουμε. Είναι δηλαδή μια διαδικασία γύρανσης σε υγεία και αποτελεσματικότητα όσον αφορά την εργασία και την αποδοτικότητα. Αυτό είναι ένα υψηλό επίπεδο φιλοσοφικής προσέγγισης. Όλοι γνωρίζουν ότι όλα τα στατιστικά στοιχεία και συστατικά στοιχεία που χρειάζονται βρίσκονται διαθέσιμα στο τραπέζι. Δεν χρειάζεται να επινοήσουμε κάτι καινούριο. Και τις γνώσεις και τα στοιχεία τα έχουμε. Ας το συνειδητοποιήσουμε αυτό και ας δράσουμε αποτελεσματικά. Πολλά στοιχεία βρήκα στην ημερήσια διάταξη στο θεματολόγιο ημερολόγιο της ε, υπηρεσίας μας του Ιδρύματος ε, για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία. Διότι επικεντρώνονται στα κέρια στοιχεία. Και τέλος, ας πούμε, είναι και αυτό σημαντικό, ας παράξουμε κοινωνική ασφάλεια, ένα πλαίσιο κοινωνικής ασφάλειας για τους γυρεότερους, τους πιο ηλικιωμένους, τους πρεσβύτες και το λέμε αυτό διότι θέλουμε να διατηρήσουμε την ε, ικανότητά τους και το δυναμικό τους για το μέλλον. Για να γίνει αυτό χρειάζονται όλες αυτές οι μεθοδοί μεθοδολογικές ε, προσεγγίσεις και όλα αυτά τα στοιχεία αλλά από και την άλλη πλευρά ε, το θεματολόγιο για την βελτιστοποίηση αυτών των στοιχείων με τον καθορισμό σαφών προτεραιοτήτων για τον πρώτο πυλώνα των συνταξιοδοτικών συστημάτων και φυσικά πέρα από τον πρώτο πυλώνα να βελτιστοποιήσουμε και τον δεύτερο πυλώνα ώστε να είμαστε αποτελεσματικοί. Συνολικά και τα προγράμματα του Eurofound είδα ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως κατευθυντήριες γραμμές, ως προσανατολισμοί για να είμαστε αποδοτικοί. Ας τονίσω το στοιχείο της entrepreneurship, του επιχειρήν, της επιχειρηματικότητας. Αυτό δεν σημαίνει να είναι κανείς ο ίδιος ιδρυτής μιας επιχείρησης, σημαίνει μια προσέγγιση, μια έννοια, ένα ιδανικό επιχειρηματικότητας και δράσης. Και αυτό πρέπει να μας εμπνέει σε υψηλό επίπεδο. Και ολοκληρώνω κοινωνική και καινοτομία σαν ανώτατο επιστέγασμα ως ιδέα και θέλω να προσθέσω εδώ το εργαλείο, το μέσο της διαχείρισης ε, της κοινωνικής αυτής αηφορίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ που τηρήσατε και το χρόνο σας. Η Κίνγκα Γκόντς τώρα έχει το λόγο. Για έξι λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Λειτουργεί το μικρόφωνο μου, ρωτά μιλήτρια, ναι. Ωραία. Πρώτα απ' όλα. Ευχαριστώ πολύ τους τέσσερις οργανισμούς για όλα αυτά που μας είπαν. Από αυτά φαίνεται πόσο σημαντικό είναι να ακούμε τις απόψεις τους για την ασφάλεια και την υγιεινή στον χώρο εργασίας, την απασχόληση, την κατάρτιση, την επαγγελματική κατάρτιση. Όλα αυτά τα στοιχεία είναι πάρα πολύ σημαντικά. Είναι καλό να τα ακούμε αυτά τα επιχειρήματα από εσάς. Γιατί έτσι υπογραμμίζεται αυτά που σκεφτόμαστε κι εμείς. Επίσης ήταν πολύ σημαντικό για μένα να ακούσω τον Υπουργό εγώ είμαι από την Ουγγαρία. Οι, με, οι καινούργιες χώρες μέλη λίγο πολύ αντιμετωπίζουν τις ίδιες καταστάσεις. Μολδαβία, Ουγγαρία και άλλες χώρες στην περιοχή. Η συζήτηση αυτή λοιπόν θα συνεχιστεί σε αυτή την κατεύθυνση. Επίσης χάρηκα που άκουσα και τον κύριο Μπέκερ με τον οποίο χαίρομαι που συνεργάζομαι στο φάκελο αυτό για την εκπαίδευση. Προσπαθούμε έτσι να βρούμε νέους δρόμους για την εκπαίδευση που να βοηθούν στην κοινωνική ένταξη και να προετοιμάζουν καλύτερα τους νέους να είναι ευέλικτοι για να μπορέσουν να ανταποκριθούν καλύτερα στις σύγχρονες προκλήσεις και τις νέες συνθήκες εργασίας. Τη συζήτηση αυτή λοιπόν σίγουρα θα την συνεχίσουμε πέρα από την αίθουσα αυτή. Τώρα όσον αφορά το κοινωνικό μοντέλο, συνέπεια της κρίσης διαπιστώνουμε όλο και περισσότερο είναι ότι οι πολίτες όλο και περισσότερο υποφέρουν και ότι η κρίση υπονομεύει όλο και περισσότερο το, το κοινωνικό μοντέλο, γιατί πρόκειται για μια κρίση απασχόλησης, δημοσιονομική και πολιτική πολλές φορές. που με τη σειρά τους υπονομεύουν τις βασικές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεπώς, εάν θέλουμε η Ευρώπη να είναι πιο ελκυστική για τους πολίτες, τότε έχουμε ειδική ευθύνη να διατηρήσουμε το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο. Σημαίνει επίσης ότι αυτοί που χάνουν τις δουλειές τους, αυτοί οι οποίοι βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας για λίγο για πολύ, Το σύστημα κοινωνικής προστασίας πρέπει να τους προστατεύει και να τους βοηθάει να συνεχίζουν να είναι απασχολήσιμοι. Να μπορέσουν κάποια στιγμή να βρουν δουλειά. Ενώ όσο πιο πολύ χρόνο μένει κάποιος στην ανεργία, τόσο λιγότερο πιθανότητα έχει να βρει δουλειά. Χάνουν τη δυνατότητα να βρουν άλλη δουλειά. Είπατε κι εσείς ότι υπάρχουν σωματικές και ψυχικές ασθένειες που έχουν να κάνουν με την ανεργία. Η μακροχρόνια ανεργία έχει τις χειρότερες συνέπειες. Συνεπώς τα συστήματα κοινωνικής προστασίας έχουν μεγάλη σημασία ώστε οι άνθρωποι να παραμείνουν κοντά στην αγορά εργασίας, να μην απογιστρωθούν από αυτήν. Για μας είναι πολύ σημαντικό να φροντίσουμε τα εκπαιδευτικά συστήματα να προσανατολιστούν προς τις σημερινές ανάγκες, να χρησιμοποιήσουν όλο το υπάρχον δυναμικό, όλους τους νέους, για παράδειγμα. Η ιδέα του να δούμε την εκπαίδευση διαφορετικά είναι κάτι που με τραβάει. Δύο στοιχεία για μένα είναι βασικά στο εκπαιδευτικό σύστημα. Το ένα είναι τα εγκάρσια προσόντα και δεξιότητες που προετοιμάζουν τους νέους καλύτερα για να αντιμετωπίσουν τις μελλοντικές προκλήσεις της αγοράς. Να είναι δηλαδή ελαστικοί, να μπορούν να λύνουν εύκολα τα προβλήματα, να είναι δημιουργικοί, καινοτόμοι, να ξέρουν ξένες γλώσσες, να είναι αρκετά ελαστικοί για να μπορούν να προσαρμοστούν σε διαφορετικές συνθήκες εργασίας και σε διαφορετικές χώρες. Οι νέοι να μπορούν ε, να μαθαίνουν πώς να δουλεύουν ομαδικά με ανθρώπους από άλλες χώρες, άλλες νοτροπίες. Για να έχουμε ένα τέτοιο εκπαιδευτικό όμως σύστημα πρέπει να προετοιμάσουμε κατάλληλα τους δασκάλους, τους καθηγητές και αυτοί να μπορούν να έχουν επαφές με άλλες νοοτροπίες, να μαθαίνουν να προσαρμόζονται σε άλλες μεθοδολογίες ανάλογα με τις ανάγκες. Βλέπουμε σήμερα ότι όλο και περισσότερο τα παιδιά πρέπει να προσαρμόζονται στα εκπαιδευτικά συστήματα και αν δεν ανταποκρίνονται καλά, απλώς το σύστημα τους πετάει έξω. Για το 2020 έχουμε πολλούς φιλόδοξους στόχους. Για να τους πετύχουμε όμως, να μην εγκαταλείπουν το σχολείο για παράδειγμα τα παιδιά, πρέπει να αλλάξουμε και την κατάρτιση των καθηγητών και να προσαρμόσουμε τα εκπαιδευτικά συστήματα στις ανάγκες των παιδιών και όχι ανάποδα. Πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη μας όλες αυτές τις πτυχές και ο καλύτερος τρόπος για να το πετύχουμε είναι ο κοινωνικός διάλογος. Να έχουμε συνέχεια διάλογο με όλους εκείνους που έχουν να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο στο όλο αυτό σύστημα. Ελπίζοντας ότι με τον κοινωνικό διάλογο θα συμπεριλάβουμε και εκείνους οι οποίοι βρίσκονται μακριά από τους χώρους εργασίας σήμερα. Alors, Η τρίτη ευρωβουλευτής που θα μιλήσει είναι η Αντέα Μακεντάιερ. το ECR, που ήταν και η συγγήτρια για την επιχειρηματικότητα και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Ε, έχετε το λόγο για 6 λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τους οργανισμούς, ε, τους εκπροσώπους των υπηρεσιών αυτών για τις ε, συνεισφορές τους. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα τα όσα ακούσαμε και τον Υπουργό. Έχουμε διάφορα ευρωπαϊκά ε, κοινωνικά μοντέλα, το μοντέλο του Ηνωμένου Βασιλείου, το σκανδιναβικό, το βαλτικό, το γερμανικό. Το κλειδί της πρόοδου της Ευρώπης είναι η στενή συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, ο επιμερισμός των βέλτιστων πρακτικών, ο κοινό σκοπός να γίνει η Ευρώπη συνολικά πιο ανταγωνιστική ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς και η δυνατότητά μας ως Ευρώπη να, να ανταγωνιστούμε ε, στην παγκόσμια σκηνή. Διάφοροι μίλησαν για ανταγωνιστικότητα σήμερα το πρωί. Όπως σας είπε και η Πρόεδρος, είμαι εισηγήτρια της Επιτροπής μας για μια έκθεση για το πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να συνεισφέρει στην δημιουργία ενός πρόσφορου περιβάλλοντος, ούτως ώστε ε, οι επιχειρήσεις ε, και οι καινούργιες επιχειρήσεις να μπορούν να δημιουργούν θέσεις απασχόλησης. Δεν είναι οι κυβερνήσεις που δημιουργούν τις θέσεις απασχόλησης, αλλά ε, οι επιχειρήσεις και οι επιχειρηματίες που φτιάχνουν τις επιχειρήσεις δημιουργούν τις θέσεις απασχόλησης. Ξέρω ότι ε, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τα απαραίτητα προσόντα και τις δεξιώσεις. Υπάρχει ένα έλλειμμα. Παραδείγματο χάρη το προσωπικό των πληροφορικάριων. Μέχρι το 2050 θα έχουμε έλλειψη 700.000 τέτοιων ανθρώπων. Επίσης, μα λείπουν μαθηματικοί, μηχανικοί, και θα είναι δύσκολο, όλο και πιο δύσκολο να καλύψουμε τις ανάγκες, όλο και, όλο και αυξανόμενες ανάγκες των επιχειρήσεων. Αναφέρθηκε και από άλλον ομιλητή αυτό το έλλειμμα των προσόντων, των δεξιοτήτων. Χρειαζόμαστε λοιπόν πιο στενή συνεργασία μεταξύ των πανεπιστημίων ειδικά και των σχολείων βεβαίω, αλλά κυρίω των ε, πανεπιστημίων και των επιχειρήσεων. Την περασμένη εβδομάδα με μεγάλη χαρά ε, το Πανεπιστήμιο στην περιοχή μου, του Βόρειου Χάμπτερ, άνοιξε ένα γραφείο εδώ στις Βρυξέλλες και περιέγραψε τον εαυτό του στο Πανεπιστήμιο των Ευκαιριών. Γιατί ξεχωρίζει αυτό το πανεπιστήμιο, γιατί. Γιατί το 75% των φοιτητών του προέρχονται από την στενή περιοχή, δηλαδή, δηλαδή εξυπηρετούν τελικά την ίδια την περιοχή τους, την πατρίδα τους και Προσπαθεί λοιπόν το Πανεπιστήμιο αυτό να δώσει στους ανθρώπους αυτούς τέτοια προσόντα που τους χρειάζονται σε εκείνη την περιοχή ακριβώς. Ε, είμαστε στα δυτικά Μίτλαντ του Ηνωμένου Βασιλείου και έχουμε πολλές βιομηχανίες. Ε, επειδή λοιπόν αυτό το Πανεπιστήμιο λαμβάνει υπόψη α, τις ανάγκες της περιοχής, το 90% των αποφύτων βρίσκουν δουλειά. Είναι καλό το αποτέλεσμα. Βέβαια, είναι πολύ θεραπευτικό όταν βλέπετε ότι ένα πανεπιστήμιο ψάχνει και κοιτάζει να δει τις ανάγκες της ε, τοπικής βιομηχανίας και δίνει στους φοιτητές τα προσόντα που χρειάζεται αυτή η περιοχή. Εν συνεχεία θα ήθελα να μιλήσω για την επιχειρηματικότητα. Κυρία Σέρμπαν αναφέρθηκε ειδικά σε αυτό. Όταν εθαρρύνουμε τους φοιτητές, στα πανεπιστήμια πάντα, έτσι, να γίνουν επιχειρηματίες, τότε δημιουργούνται νέες ιδέες. Από αυτούς τους ανθρώπους δημιουργούνται νέες ιδέες. Ε, ένα άλλο πανεπιστήμιο στην περιοχή μου, το Άστον, που, που είναι στα περίχωρα του Μπέρμιχαμ, έχει προγράμματα όπου οι φοιτητές αναπτύσσουν ιδέες και εν συνεχεία πηγαίνουν ε, σε διάφορες μονάδες όταν αποφοιτήσουν ε, με αυτές τις ιδέες εντάσσονται σε αυτές τις ομάδες. δηλαδή γύρω από αυτούς τους φοιτητές υπάρχει υποδομή. Ε, γιατί για πάρα πολλούς ανθρώπους, μην ξεχνάτε το να ξεκινήσουν μια επιχείρηση είναι μεγάλη πρόκληση. Και το βασικό θα είναι σε όλη την Ευρώπη να βοηθήσουμε αυτού του ανθρώπου να ξεκινήσουν τις δικές τους επιχειρήσεις. Στην περασμένη εβδομάδα ακούσαμε πόσα πολλά εμπόδια υπάρχουν. Όλα τα έντυπα που πρέπει να, να, να ε, συμπληρώσει, όλα τα μέσα στα οποία πρέπει να πα ε, και πολλά μπορούν να γίνουν για να βοηθήσουμε αυτού του ανθρώπου, να ξεκινήσουν τη δική του επιχείρηση. Για τι μικρομεσαίες επιχειρήσει. Και εγώ και οι συνάδελφοί μου ατέρμονα ξανά και ξανά ζητάμε τη μείωση της γραφειοκρατίας, την απλούστευση ε, των διαδικασιών. Ο κύριος ε, Μενέντες Βαλδέσκι Κρίστα, είπαν Σέντλατσεκ, είπαν ότι μπορούμε να απλουστεύσουμε την νομοθεσία χωρίς να μειώσουμε την προστασία των εργαζομένων. Φυσικά δεν πρέπει να μειώσουμε την προστασία των εργαζομένων. Εμείς στη χώρα μου ε, έχουμε καλό, καλές επιδόσεις στην υγεία και την ασφάλεια. Αν θέλουμε να απασχολήσουμε πολλούς ανθρώπους στις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στις μικρές, ε, δεν μπορούμε συνέχεια να αναγκάζουμε το προσωπικό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων να αποκρυπτογραφούν την νομοθεσία. Και οι μικρέ επιχειρήσει και οι οικογενειακέ επιχειρήσεις θα πρέπει και θέλουν να βοηθήσουν του εργαζόμενου του να παραμείνουν υγιείς. συχνά παλεύουν να καταλάβουν την νομοθεσία. Πρέπει να του βοηθήσουμε λοιπόν, να είναι εύκολη, εύληπτη η νομοθεσία. Νομίζω θα του εξυπηρετούσαμε πάρα πολύ. Και εκεί ακριβώ οι κοινωνικοί εταίροι μπορούν να παίξουν κάποιο ρόλο. Ε, σας ευχαριστώ. σας ευχαριστούμε πολύ. Μένετε στο κοινωνικό ζήτημα, αλλά <laughs> είναι δικιά σας ε, επιλογή. Πέρασε ο χρόνος σας. Τώρα θα δώσω το λόγο στον τέταρτο. Ουι Κοντμπούχεν, Γενικός Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου μηχανικών, θα το διαβάσω στα αγγλικά, λέει η πρόεδρος, εργοδότες βιομηχανιών σχετικών με τη μεταλλουργία και την μηχανολογία. Σε ΜΕΤ είναι τα αρχικα c e C-E-E-M-E-T. Για έξι λεπτά έχετε το λόγο. Παρακαλώ. Σα ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Να σας υπενθυμίσω ότι φυσικά τα δύο κέρια θέματα είναι ο κοινωνικός διάλογος και η καινοτομία τον χώρο στις Ευχαριστώ που μας το υπενθυμίσατε για το θέμα του ε, αηφόρου κοινωνικού προτύπου και το κοινωνικό διάλογο. Ευχαριστώ για την πρόκληση, πρόσκληση ε, για να συμμετάσχουμε σε αυτό το ενδιαφέρον ε, πάνελο συζήτηση. Εκπροσωπούμε 200.000 εταιρείε που δίνουν άμεση απασχόληση σε 30 περίπου εκατομμύρια εργαζόμενου πανευρωπαϊκά. Οι περισσότεροι από τους προλαλήσαντες μίλησαν για την ανταγωνιστικότητα, τόνισαν την ανταγωνιστικότητα και το εκτιμώ ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της Μολδαβίας το ανέφερε αυτό όσον αφορά την οικονομική, το οικονομικό δυναμικό και την οικονομική ισχύ και στην κατοχήρωση του άρθρου 3 στη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αυτό το στοιχείο. Όμως αυτό βασίζεται σε μια ισορροπημένη οικονομική ανάπτυξη ως προϋπόθεση και όρο. Και όταν κάνουμε λόγο για την ε, ανταγωνιστικότητα, κάνουμε λόγο για την ανταγωνιστικότητα της ε, διακυβέρνησης, ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων ε, της οικονομίας, καθώς επίσης και για τους εργαζόμενους. Όπως είπαμε είναι μια κοινή ευθύνη και ίσως θα έχουμε συναγάγει το συμπέρασμα ότι υπάρχουν πολλά άτομα που ζητούν για αυξημένη εμπλοκή και συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, πράγμα στο οποίο θα επανέλθουμε στη συνέχεια. Χρειαζόμαστε λοιπόν την αηφορία στην ανάπτυξη, αηφορία στην αύξηση του οικονομικού μας δυναμικού και αυτό είναι η ας το πω έτσι, αποστολή στο να μπορέσουμε να πετύχουμε την αύξηση της συμμετοχής ε, ως στόχο της, ε, της πραγματικής οικονομίας των επιχειρήσεων, ώστε να υπάρξει μια συνεισφορά στην αύξηση του ΑΕΠ μέχρι το 2020, να υπάρξει μια αύξηση πάνω από το 15% μέχρι το 20% στην Ευρώπη του 2020. Χρειαζόμαστε λοιπόν αύξηση της ανταγωνιστικότητας με μια οικονομική βιομηχανική βάση ως προϋπόθεση για την αηφορία στις θέσεις απασχόλησης και την ανταγωνιστικότητά τους, για την αηφορία και των κοινωνικών συστημάτων ασφάλισης. Και εδώ επιτρέψτε μου ίσως ε, να κάνω μια σύντομη αναφορά στην έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας για την Παγκόσμια Ανάπτυξη που δημοσιεύθηκε και αναφέρει ότι για την Ευρώπη ενώ έχουμε 10% ε, κάτω από, ε, ε, του, του, συνολικού εργατικού δυναμικού παγκόσμια έχουμε 50% και παραπάνω όσον αφορά το ποσοστό παγκόσμια για την κοινωνική ασφάλιση που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να το δούμε αυτό ως συνεισφορά μαζί με τα κύρια στοιχεία συνδυασμό για την ανταγωνιστικότητα, ανταγωνιστικότητα για να αντιμετωπίσουμε την κρίση. Ναι, την κρίση αλλά και την δημογραφική γύραση, η δημογραφική κάμψη που θα είναι μια ορολογική βόμβα. Να είμαστε ανταγωνιστικοί αλλά ως επιχειρήσεις ε, πρέπει να βρισκόμαστε και είμαστε στην πρώτη γραμμή του παγκόσμιου ανταγωνισμού. Έχουμε ανταγωνιστές ε, ως Ευρωπαίοι επιχειρηματίες ε, από, όλες τις, από όλα τα σημεία του ορίζοντα ορίζοντα Πρέπει να έχουμε λοιπόν ευφυή νομοθεσία, δημιουργική νομοθεσία, συμπεριλαμβάνοντας ε, σωστές ε, μελέτες εκτιμήσεων και επιπτώσεων, ελαστικές πολιτικές ε, για την αγορά εργασίας που μπορούν να οδηγήσουν σε προσαρμογές, να έχουμε αηφόρα ανταγωνιστικά ασφαλιστικά συστήματα και υπηρεσίες, καθώς επίσης και την αντιμετώπιση αν δει κανεί για παράδειγμα το τι έγινε κατά τις τελευταίες δεκαετίες, κάλυψη των αναγκών και δεξιοτήτων που χρειαζόμαστε στην Ευρώπη για εξειδικευμένους εργάτες και εργατικό δυναμικό. Πρέπει λοιπόν να έχουμε μια συγκεκριμένη προσαρμοστικότητα και δυνατότητα προσαρμογής για να σημειωθεί ανάπτυξη από πλευράς μας. Όταν κάνουμε λόγο λοιπόν για την ανάπτυξη ως πρότυπο. Πρέπει να λάβουμε επίσης υπόψη ότι με τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2004, το Big Bang, τη μεγάλη έκρηξη της διεύρυνσης, βλέποντας την οικονομική ανάπτυξη και βαίνοντας εκ παραλίλου με τις κοινωνικές εξελίξεις και κοινωνική μετεξέλιξη αυτών των χωρών, πρέπει να πει κανείς ότι η οικονομική και κοινωνική μετεξέλιξη και ανάπτυξη δημιούργησαν ένα πολύ θετικό συνδυασμό, οικονομικό και κοινωνικό, για την σημείωση, την επίτευξη προόδου. Και όσον αφορά για τις ε, κατευθυντήριες γραμμές, ε, σίγουρα η δική μας, ε, το δικό μας όργανο είναι υπέρ του κοινωνικού διαλόγου μέσα στο πλαίσιο των επιχειρησιακών δράσεων και των βιομηχανιών μας στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Και έχουμε στο θεματολόγιο μας, στην ημερήσια διάταξη, την αντιμετώπιση των θεμάτων της, των ηλικιωμένων εργαζόμενων υπό το ναι, πρίσμα της αηφορίας και προσαρμογής και επιμόρφωσης και δεξιοτήτων λόγο για την προσαρμοσιμότητα όσον αφορά και τις συμβάσεις εργασίας. Και από πλευράς μας είδαμε με μελέτη που κάναμε ότι δεν χρησιμοποιούμε υπερβολικά αυτά τα μέσα. Είτε είναι προσωρινή απασχόληση, είτε είναι προσαρμόσιμη ελαστική απασχόληση. Συνολικά πρέπει να πούμε ότι 5% είναι η κάθε μια από αυτές τις κατηγορίες που προαναφέραμε σήμερα. Όταν γίνεται λόγος για την εκπαίδευση και παιδεία και κατάρτιση, η ΣΥΜΑΚΤ έχει δημοσιεύσει και εδώ θέλω να υπογραμμίσω απόλυτα τη σπουδαιότητα της βελτίωσης συνεργασίας μεταξύ βιομηχανίας και των παρόχων κατάρτισης και εκπαίδευσης, αλλά επίσης και συνεργασία μεταξύ βιομηχανιών και επιχειρήσεων και πανεπιστημίων σε μια συνέργεια. Όπως είπε η κυρία Μακεντάρ, υπάρχουν πολύ θετικά παραδείγματα τέτοιου είδους συμμαχιών και συνεργασιών στην Φινλανδία, για παράδειγμα, όπου από το Πανεπιστήμιο περνάνε σε επιχειρήσεις ε, και εργάζονται και ε, βρίσκουν δυνατότητα ε, περαιτέρω απασχόλησης οι νέοι. Είναι λοιπόν πολύ καλή η δουλειά που γίνεται και σε σχέση με την βιομηχανία δείχνουμε ότι είμαστε ένας αξιόπιστος εταίρος, ισχυρός εταίρος που μπορεί να συνεισφέρει και έχουμε διασφαλίσει επίπεδο απασχόλησης σε υψηλότατα επίπεδα. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Merci beaucoup. Ευχαριστούμε πολύ. Και έτσι φτάνουμε στην πρώτη τελευταία ομιλητριά μας, την Καρέλα Φίσπαχ Πίτελ, Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας των Δημοσίων Υπαλλήλων. Για έξι λεπτά έχετε το λόγο. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Λίγα δευτερόλεπτα θέλω για να πω στον κύριο Λάσλο. ότι το θέμα μας του ανταγωνισμού με φέρνει σε αυτά που ακούσαμε το πρωί για την αλληλεγγύη. Εγώ θα έχω μια διαφορετική προσέγγιση. Το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο θα το χρησιμοποιήσω εγώ σαν βάση για την εφαρμογή των ανθρώπινων δικαιωμάτων και για να πετύχουμε περισσότερη ισότητα. Αν δεχτούμε όμως αυτή την οπτική γωνία του οικονομικού ωφέλους από το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο, τότε πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και το κόστος της μη κοινωνικής Ευρώπης. Κάτι το οποίο έχει άμεση σχέση με την σημερινή κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί νέοι, ιδιαίτερα άνεργοι, που δεν έχουν καμία ευκαιρία να βρουν δουλειά και γι' αυτό και έχουμε μιλήσει για τη χαμένη δεκαετία. Εντάξει, εκπροσωπώ βέβαια τους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα και όχι μόνο, όλων των υπηρεσιών που παίζουν σημαντικό ρόλο στον κοινωτικό τομέα, είτε πρόκειται για την κοινωνική ασφάλιση, είτε πρόκειται για γραφεία βρέσεως εργασίας, εκπαίδευση. Νομίζω λοιπόν ότι πολλά μπορούμε να πούμε για το ρόλο του δημόσιου τομέα στο κοινωνικό αυτό μοντέλο. Το κύριο επιχείρημά μου πάντως είναι ότι δεν μπορούμε να δεχτούμε άλλη διάβρωση αυτού του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου. Και επειδή κάτι ρωτήσατε πριν, εγώ θα το αλλάξω λίγο, γιατί νομίζω το πλαίσιο μέσα στο οποίο θέσατε το ερώτημα, δείτε σας το λέτε ότι με την οικονομική κρίση δεν μπορούμε ίσως να αντέξουμε άλλο αυτό το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο. Ε, λοιπόν, εγώ δεν συμφωνώ ούτε και με το επιχείρημα ή με τη σχέση που κάνετε, που βάζετε ανάμεσα στη δημογραφική κατάσταση και την οικονομική κρίση. Αναμφίβολα πρόκειται για δύο σημαντικέ προκλήσεις, αλλά, αλλά δεν είναι η ίδια όψη του νομίσματος. Πρόκειται για δύο διαφορετικούς παράγοντες. Και αν ο διπλανός μου μιλάει για ορολογική βόμβα, είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε το γεγονός μιας ε, μεγαλύτερης ηλικία κοινωνίας. Κάτι άλλο που θέλω να υπογραμμίσω είναι ότι αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης και των μέτρων που έχουν ληφθεί στα πλαίσια της οικονομικής διακυβέρνησης, ο κοινωνικός διάλογος υποφέρει πολύ. Σε πολλές χώρες έχει πληγή με την λιτότητα στην Ελλάδα, στην Ισπανία, στις βαλικές χώρες, στη Ρουμανία. Αυτή η κατάσταση πραγμάτων υπονομεύει τα θεμελιώδη κοινωνικά δικαιώματα. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσης είναι απρόθυμη να έρθει να προτείνει ξεκάθαρα κοινωνικά μέτρα. Και ακόμα πιο σημαντικό είναι ότι εμεί πιέζουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρουσιάσει μια στρατηγική για την ασφάλεια και την υγεία στο χώρο εργασία. Συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπε η προηγούμενη ομιλήτρια Κρίστα Σέλτερτσεκ. Η, υγεία και η ασφάλεια είναι βασικός παράγοντας που ενισχύει την ανταγωνιστικότητα. Μη υγιείς εργαζόμενοι δεν είναι παραγωγικοί στοιχείο που είναι κλειδί για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας και των κοινωνιών μας. Πιστεύω ότι αυτή την οπτική γωνία δεν πρέπει να την παραβλέπουμε, αντίθετα. Υπάρχουν τρεις εκλαδικές συμφωνίες, συμβάσεις, τις οποίες έχουν διαπραγματευτεί ευρωπαϊκά συνδικάτα που καλύπτουν τους τομείς της υγείας και της ασφάλειας είναι την αλληλεία από τα εσωτερικά ύδατα και από τους κομμωτές. Οι εργαζόμενοι, οι εργαδότες και τα συνδικάτα έχουν συμφωνήσει πάνω σε ένα κείμενο το οποίο καλύπτει πολύ σημαντικά στοιχεία. Όλες αυτές οι συμφωνίες ζήτησαν ανεργαζόμενοι να γίνουν οδηγία. Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή όμως έχουν σταματήσει. Κάτι που βρίσκω απαράδεκτο και πιστεύω επίση ότι πρόκειται για παραβίαση των συνθήκων. Πρέπει να διορθωθεί αυτή η κατάσταση επιγόντω. Εσείς που είσαστε Επιτροπή Απασχόλησης μπορείτε να παίξετε τον σωστό ρόλο και να στηρίξετε επ' αυτού τους εργαζόμενους. Τέλος. Έχει μεγάλη σημασία και το θέμα των, ε, του εισοδήματος. Τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό. Χαίρομαι που εξακολουθούν να υπάρχουν διαβουλεύσεις για να καταπολεμηθεί η αδήλωτη εργασία. Διότι μόνο έτσι μπορούμε να έχουμε έσοδα από την κοινωνική ασφάλιση και μπορούμε να καταπολεμήσουμε και την παράνομη εργασία. Αύριο νομίζω εξετάσετε την έκθεση της Γιούκα Στάινεκ που αναφέρεται στις επιθεωρήσεις εργασίας που είναι μια στρατηγική για τις καλές συνθήκε εργασίας. Χαίρομαι για την πρωτοβουλία αυτή και ελπίζουμε ότι θα μας δοθεί ευκαιρία να συνεργαστούμε και παρατέρω μαζί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ για τις ε, συνηθίσεις ε, ε, συμφωνίες. Περιμένουμε να μας ενημερώσει βεβαίως η Κομισιόν. Πρέπει να σας πω ότι η δική μας Επιτροπή είναι πολύ κινητοποιημένη και θέλουμε να, και ξέρετε πολύ καλά ότι πιέζουμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να περάσει αυτό το θέμα από το Σώμα Επιτρόπων. Επίσης για τη δημιουργία ενός ε, σώματος επιθεωρητών και εκεί είμαστε πολύ κινητοποιημένοι. Η τελευταία μας παρέμβαση είναι από τον Μποντουάν Ρεγκού, τον ευχαριστώ που ήρθε. Είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τροποντινά, έτσι. Δεν θέλουμε να μας απαντήσει το θέμα των κομμωτών. Εκπροσωπεί το Γραφείο Συμβούλων Ευρωπαϊκής Πολιτικής τον ΠΕΠΑ και έχει μία πιο στρατηγική ματιά. Θέλω να μας μιλήσει και για τον κοινωνικό διάλογο και για την καινοτομία στον τόπο εργασίας και για την εκπαίδευση. Έξι λεφτάκι για σας, όπως όλοι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να απαντήσω τις δύο ερωτήσεις σας ε, λέγοντας τρία πράγματα. Κάποια από αυτά που θα πω δεν είναι ε, καινούργια, είναι παλιά, αλλά δημιουργούν μια θετική επίπτωση και για τις δύο μεριές. Μερικές φορές όμως πρέπει να κάνουμε κάποια παζάρια, κάποια, κάτι να δώσουμε και κάτι να πάρουμε. Και τρίτον πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και την εξέλιξη των τεχνολογιών. Κοιτάξτε λοιπόν καταρχάς την πρώτη κατηγορία. Πού κερδίζουμε όλοι οι εμπλεκόμενοι. Ε, όλοι όσοι μίλησαν α, συμφωνούν ότι η εκπαίδευση, η ασφάλεια, η υγεία, οι καλές συνθήκες εργασίας είναι σημαντικές για το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο, αλλά βοηθούν και την, το ανταγωνισμό και την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία. Και αυτές οι επιχειρήσεις είναι κατά πάσα πιθανόν να αναπτύξουν την καινοτομία αυτή. Ε, επίσης, κάποια μέτρα για την ε, οικογένεια είναι τμήμα του ευρωπαϊκού οικονομικού μοντέλου και κάποια θέματα κατά των διακρίσεων. Δεν το συζήτησαμε πολύ αυτό, αλλά τέλος πάντων. Πάντως, γύρω από τα θέματα υπάρχει γενικά ευρεία συνένεση. Αν λοιπόν ε, υπάρχει συμφωνία, τότε φυσικά οι εργαζόμενοι ενδιαφέρονται να προωθήσουν αυτά τα πράγματα, αλλά και οι επιχειρήσεις, γιατί και οι μέρη και κερδίζουν. Ξέρετε πολύ καλά ότι ορισμένε ε, επιχειρήσεις, ε, παραδείγματο χάρη στην, ε, στα ξενοδοχεία, στι βιομηχανίε, κάνουν τέτοια προσπάθεια. και δημιουργούν, ας πούμε, μαθητείες και στάζ για τους εργαζόμενούς τους πολλές επιχειρήσεις. Επίσης, για το πώ θα γίνουμε ανταγωνιστικοί. Πρέπει να είναι ανταγωνιστικέ οι αγορέ. Αν τα επιχείρησει είναι πιο θετικέ, ε, πιο καλές, θα κερδίσουμε μερίδα της αγοράς, θα βγάλουν κέρδη. Ε, η ανταγωνιστική αγορά εξασφαλίζει ότι θα έχουμε κέρδη και βεβαίως ε, υπάρχουν και τα, απαραίτητα κίνητρα για τις εταιρείε. Και τότε και ο κοινωνικός διάλογος είναι πιο απλός. Φυσικά υπάρχουν διαφορές ε, από χώρα σε χώρα. Παραδείγματος χάρη τα μέτρα υπέρ της οικογένειας δεν είναι τα ίδια σε όλες τις χώρες. Αλλά εν πάση υπάρχει ένα σύστημα κοινωνικών εταίρων που προωθεί όλα αυτά τα θέματα. Η, δεύτερη συνιστόσα ε, είναι οι περιπτώσεις όπου δεν κερδίζουν όλοι, δεν συμφωνούν όλοι και δεν κερδίζουν όλοι. Ε, το θέμα των ε, συντάξεων καταρχάς Υπάρχουν πάρα πολλέ προκλήσει, γίνονται πάρα πολλέ συζητήσει. Ε, ορισμένοι συζητάνε το όριο ταξιοδότηση. και μια άλλη συζήτηση είναι για την προστασία, την κοινωνική προστασία. Ε, υπάρχει γενικά ε, συνένεση ότι πρέπει να υπάρχει κοινωνική προστασία, αλλά ποιο θα την παράσχει αυτή την προστασία, τα κοινωνικά συστήματα, οι, οι επιχειρήσει, οι κυβερνήσει, ποιο θα την οργανώσει την προστασία. Εκεί γίνονται πάρα πολλέ συζητήσει και είναι πολύ σημαντικό ο κοινωνικό διάλογο και οι κοινωνικοί εταίροι κάπω να συμφωνήσουν. Φυσικά στην πράξη οι κυβερνήσεις συμμετέχουν σε αυτές τις ε, συζητήσεις γιατί συχνά τα συστήματα κοινωνική ασφάλιση και τα συνταξιδοτικά συστήματα χρηματοδοτούνται και από τι κυβερνήσει. Επομένω, ε, και οι κυβερνήσει αλλά και οι φορολογούμενοι πίσω από αυτέ πρέπει να συμμετάσχουν. Ε, δεν θα πω τίποτα άλλο. Θέλω να μπω στην τρίτη κατηγορία. Είναι το, η τρίτη συνιστόσα του κοινωνικού μοντέλου. Υπάρχουν νέοι καινοτόμοι τρόποι εργασίας που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν νέες ε, θετικές καταστάσεις. Αν ε, ακούτε τους ε, μελλοντολόγους, τους συμβούλους, και εγώ ήμουν παλιά σύμβουλος, ακούτε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Ε, μιλάμε για την εργασία η οποία να βασίζεται στο project, στο έργο, στο πρόγραμμα ή, εν πάση περιπτώσει, να οργανώσει διαφορετικά την ιεραρχία της δουλειάς. Οι ιεραρχικές σχέσεις να είναι αλλιές. Ε, γίνεται πολλή δουλειά για την αυτοαπασχόληση. Ε, ε, online εκπαίδευση και προσφορά εργασίας. Δεν ξέρω τι θα δουλέψει από όλα αυτά τα μοντέλα. Δεν ξέρω. Είναι το μέλλον, ακούγεται ενδιαφέρον, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δοκιμάσουμε αυτές τις ιδέες αλλά ίσως θα πρέπει να ρωτήσουμε και τους μάνατζερ που η δουλειά τους είναι να οργανώσουν όλη αυτή την ιστορία. Σε συνεργασία βέβαια με τους εργαζόμενους. Αν τους πούμε τι θα επικρατήσει από όλα αυτά, κανένα δεν ξέρει. Άλλοι θεωρούν ότι το α θα κερδίσει, άλλοι το β. Εγώ ως υπεύθυνο για τη διαμόρφωση της πολιτικής ε, θεωρώ ότι δεν μπορώ εγώ να κάνω αυτή τη δουλειά ε, και να υποκαταστήσω τις επιχειρήσεις. Εξάλλου, ε, μπορεί η απάντηση να διαφέρει από επιχείρηση σε επιχείρηση και από τομέα σε τομέα. Και ω αρμόδιο τη διαμόρφωση πολιτική, θέλω να του ακούσω του επιχειρηματίε, να δω αν μπορούν να συμφωνήσουν. Μερικέ φορέ βλέπω ότι δεν γίνονται κάποια πράγματα γιατί υπάρχουν εμπόδια. Θέλω να του ακούσω, εν για να είμαι σίγουρο για το τι μπορεί να γίνει. Αν υπάρχει μια οριζόντια λύση, θα είναι σίγουρα το να εμπιστευτούμε τον κοινωνικό διάλογο και να βάλουμε όλα αυτά τα θέματα στον κοινωνικό διάλογο. Να τα βάλουμε και να τα συζητήσουμε. Bien, alors, maintenant... Euh, Μάλιστα. Ο ρόλος της Προέδρου είναι φρικόδη, διότι πρέπει να ξεκινήσω, να δώσω την αρκτήριο λάκτισμα στη συζήτηση και έχουμε ελάχιστο χρόνο. Δώσω την προτεραιότητα στους βουλευτέ. Η κυρία Γεζοβίτσκα έχει γραφτεί στον κατάλογο. Ποιο άλλο βουλευτή θέλει να πάρει το λόγο. Σαρκάς Κοστελό, Ατουμπατού, εσύ Άλλος κανείς που θέλει το λόγο. Μη σηκώνετε όλοι το χέρι μαζί, έτσι. Λοιπόν, άλλε δύο ερωτήσει. Όχι, καλώ. Α, εσεί, ωραία, μία, εντάξει. Ένα. παρεμβαίνων απ' έξω. Οπότε έχουμε πέντε ομιλητές. Ένα λεπτό καθένας. Παρακαλώ, κύριε Γεζορέσκα πρώτα. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πιστεύω ότι αν θέλουμε να οικοδομήσουμε ένα νέο, ισχυρό, αποτελεσματικό κοινωνικό πρότυπο, πρέπει πρώτα να δούμε τη σημερινή επίκαιρη κατάσταση και να την αξιολογήσουμε. Έκανε λόγο προλόγη σας γι' αυτό τα μέτρα τα οποία πρέπει να θεωρούνται περιτά πρέπει να καταργηθούν και να εισαχθούν νέα. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε 28 νέα, 28 ε, κράτη-μέλη με διαφορές μεταξύ τους. Ταυτόχρονα όμως πρέπει να λαμβάνουμε πάντα υπόψη την αρχή της αλληλεγγύης που πρέπει να εκφράζουμε εκπλήσωμαι ότι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τόσο σπάνια ή όχι τόσο συχνά κάνουμε λόγο για την αλληλεγγύη. Θα πρέπει στην επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό όταν κάνουμε λόγο για αυτήν να δούμε ποιες είναι πρώτα οι ανάγκες της αγοράς εργασίας σχετικά. Αν δούμε το όριο ηλικίας κατά το οποίο συνταξιοδοτούνται οι εργαζόμενοι αν θέλουμε να είμαστε αποτελεσματικοί πρέπει να το επεκτείνουμε για να, είμαστε, να προσαρμοστούμε στις ανάγκες μας. Και η ενεργοποίηση των γυναικών στην αγορά εργασίας πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ως θετικό στοιχείο. Έχετε ερώτηση? Θα ήθελα, θα ήθελα να πω ότι θα έπρεπε να σκεφτούμε ότι η δημιουργία ενός νέου ευρωπαϊκού κοινωνικού προτύπου θα έπρεπε να πάρει τέτοιου είδους μόρφη, να πάρει σάρκα και οστά με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορούμε να ενεργοποιηθούμε από κράτη που ε, ε, έχουν ανάγκες να καλυφθούν, να ενεργοποιηθούμε, να καλυφθούν οι ανάγκες με τον καλύτερο τρόπο. Αλεχάνδρο Θέρκας, μετά Μπέναραμπα του, ο κύριος Αλεχάνδρο Θέρκας, ένα λεπτό παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ίσως ε, δύο δευτερόλεπτα μόνο για να ευχαριστήσω τους Γενικούς Διευθυντές των Οργάνων ε, για το έργο που επιτελούν όταν έχουμε τους εχθρούς ε, του κράτους πρόνοιας που είναι όλο και πιο ενεργό και έντονο το έργο τους και να δούμε τις ανάγκες που υπάρχουν. Καθώς η φυσική πόρη η ενεργεια είναι περιορισμένη στην Ευρώπη το μόνο δυναμικό που έχουμε στη διάθεσή μας ε, είναι το ανθρώπινο δυναμικό και να έχουμε μια κοινωνία ισόρροπη και δίκαια που θα επιτρέπει να δώσουμε καινοτόμε δράσεις ε, ώστε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις του μέλλοντος ε, και να μην ακολουθήσουμε μια λανθασμένη πορεία καταστρέφοντας και υπονομεύοντας ακριβώς τους όρους και τα στοιχεία στα οποία πρέπει να βασιζόμαστε. Ερώτησή μου, έχει μέλλον το ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο. Και πρέπει με την ερώτηση που θέλουμε να διατυπώσουμε ως εξής. Πιστεύετε ότι έχει μέλλον η Ευρώπη χωρίς αυτό το ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο. Ευχαριστώ. Κυρία Μπέναράμπα Ματού, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Κάποιος είπε ότι μια ανταγωνιστική επιχείρηση, μια επιχείρηση που κοινωνικά προσφέρει ένα καλό περιβάλλον, χέρι μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα. Δεν είναι όμω αλήθεια αυτό. Η Amazon, για παράδειγμα, που είναι μια πολύ ανταγωνιστική επιχείρηση, παρόλα αυτά οι συνθήκε εργασία που επικρατούν εκεί είναι πολύ κακέ. Για την κυρία Έντλεν Σερμπάν θέλω να πω, η οποία αναφέρθηκε στις σχέσεις με τις γείτονε χώρε και τι πρέπει να κάνουμε για αυτά τα θέματα. Χτες οργάνωσα μία διάσκεψη με έναν ε, ειδήμονα για το Μαγκρέπ και το ρόλο των χωρών Μαγκρέπ στην πολιτική γυτνίασης. Όλοι οι εμπειρογνώμονες πρέπει να ξέρετε λένε ότι Κίνα, Ηνωμένε Πολιτείε, ο άξονα αυτός βλέπουν το ρόλο της Αφρικής να ενισχύεται προς το 2030. Οπότε στις σχέσεις της με το Μαγκρέπ η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο. Είναι σημαντικό δηλαδή να έχουμε υπόψη μας ότι ο ρόλος μας για τις σχέσεις με την Αφρική πρέπει να ενισχυθεί γιατί θα μας βοηθήσει στο μέλλον. Ευχαριστώ. Μαρ Καστέλο και μετά ο δόκτωρος Μελτατζόν. Παρακαλώ κύριε Κοστέλο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θέλω και εγώ να ευχαριστήσω όλους όσοι πήραν το λόγο σήμερα εδώ, αλλά και τους οργανωτές. Δεύτερον, υπάρχει μια αντίφαση. Από τη μια λέμε ότι θέλουμε να επενδύσουμε στην εκπαίδευση, να προστατεύσουμε το κοινωνικό μοντέλο και από την άλλη μεριά χώρες όπως είναι η Ιρλανδία που αναγκάζεται να επιβάλλει μέτρα λιτότητας κάνει περικοπές στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. Και φαίνεται αυτό από τον ε, επερχόμενο προπολογισμό στην Ιρλανδία. Δεύτερον, αν θέλουμε να αλλάξουμε την εκπαίδευση, τότε πρέπει να, να αναθεωρήσουμε και την πιστοποίηση της εκμάθησης, της γνώσης. Να μην υπάρχουν πάντα δεσμευτικοί όροι είναι κάτι που μπορούμε να προσταθήσουμε από το 2015 μέχρι το 2018. Να δούμε τα μέσα εργαλείας που έχουμε για την αξιολόγηση της μάθησης. Ώστε να φροντίσουμε έτσι να έχουμε τα προσόντα τα οποία χρειαζόμαστε για το μέλλον και την κατάλληλη αξιολόγηση. Ευχαριστούμε που θέσατε και την ερώτησή σας σε ένα λεπτό. Το λόγο τώρα έχει ο καθηγητής Dr. Σμέλφα Τζον καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Σταμπρούκ της Γερμανίας. Ένα λεπτό κι εσείς. σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε αυτή την ευκαιρία. Αναφέρθηκε το ζήτημα ουσιαστικά αν είναι επικοδομητικό να προλάβουμε και αν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, σε, να επενδύσουμε σε ασφαλείς θέσεις απασχόλησης σε μια περίοδο κρίσης. Εγώ επιστημονικά είμαι αισιόδοξο, διότι τα στοιχεία είναι σαφή. Για κάθε ευρώ που επενδύουμε έχουμε επιστροφή 2 ευρώ στην αποδοτικότητα. Μπορεί να έχουμε και επιστροφή 5 ευρώ αν δούμε και τις ε, ε, δεξιότητες όσον αφορά την αντιμετώπιση των ε, ασθενειών από τον χώρο απασχόλησης. Και ακούσαμε από την κυρία Φίσμπαχ ότι οι κομμότριες εθελοντικά οι κοινωνικοί εταίροι συμφώνησαν εθελοντικά σε ανώτερα επίπεδα, αναβαθμισμένα επίπεδα βελτιώσεων και μπορούμε να δείξουμε με παραδείγματα διαφορετικών χωρών ότι είναι αποδοτικές αυτού του είδους οι δράσεις. Ο αριθμός εκείνων που έχουν προβλήματα λόγω της απασχόλησής τους σε σχέση με την υγεία, σε σχέση με τα όσα μπορούν να εξοικονομηθούν αν έχουμε τις σωστές επενδύσεις είναι πολύ σημαντικά. Ίσως μπορούμε να βρούμε και άλλους τομείς που θα ήθελαν να συμμετάσχουν σε αυτόν τον σε αυτή τη δράση. Κοινωνικοί εταίροι που θα μπορούσαν να υποφεληθούν από βελτιωμένη πρόληψη λοιπόν ως δράση. Ευχαριστώ. Μια που έχουμε τους τέσσερις οργανισμούς και τον Υπουργό βέβαια, στους οποίους θέλω να ξαναδώσω το λόγο, νομίζω ότι πρέπει να φτάσουμε στο τελευταίο έτσι μέρος της συνάντησή μας και να σας ζητήσω σε πέντε λεπτά ο καθένας να αντιδράσετε στα όσα ακούσαμε και να απαντήσετε και στις ερωτήσεις που τέθηκαν. Λοιπόν, οι τέσσερις διευθυντές των οργανώσεων και ο υπουργό θα πάρουν το λόγο. Επειδή δεν έχουμε αρκετό χρόνο, έτσι. Ρώτα λοιπόν, Κρίστα Λετμάγερ, που είναι ο διευθυντής του ΣΕΝΤΕΦΟΠ, για να αντιδράσει στις παρατηρήσεις που έγιναν και να απαντήσει στις ερωτήσεις. Πέντε λεπτά παρακαλώ. Σε ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστώ για όλες τις ερωτήσεις αυτές. Ευχαριστώ και για τη συζήτηση και για τις ε, θετικές ανταποκρίσεις και αντιδράσεις της παρουσιάσεις. Πιστεύω ότι πιο σημαντικό είναι να επανέλθουμε σε αυτό το οποίο αναφέρθηκε ε, σε λόγο που εκφωνήθηκε, σε παρέμβαση που έγινε, πρέπει να δαπανίσουμε με καλύτερο τρόπο, να χρησιμοποιούμε τα κονδύλια με πιο σωστό τρόπο στην εκπαίδευση. Μετά θα ήθελα να προσθέσω κάτι. <clears throat> Υπάρχουν συντριπτικά αποδεικτικά στοιχεία για αυτό τις ε, θετικές αυτές ε, επιδόσεις. Δεν μπορούμε να κατανοήσουμε γιατί πρέπει να συνεχίσουμε να δρούμε με τον τρόπο που ε, δράσαμε κατά τα τελευταία έτη. Βλέπουμε το τέλος, το τέλος του τούνελ, βλέπουμε φως στην άκρη της σύραγγας. Δεν λειτουργούν τα πράγματα όπως ακολουθήθηκαν. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα θεμελιώδη μέτρα που μπορεί να είναι σκληρά θα πρέπει να αποφευθούν σε αυτές τις τις χώρες που πρέπει να μεταρρυθμιστούν, αλλά όχι με τόσο ομό και σκληρό τρόπο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Στη συνέχεια ο Χουάν Μενέντες Βαλντές ε, θα λάβει τον λόγο από πλευρά σε Eurofort. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ και σύντομα Αρκετά φυσικά πράγματα, πολλά πράγματα αναφέρθηκαν από όσου συμμετέχουν στο πάνελ και σε σχέση με τον κοινωνικό διάλογο. Θα ήθελα μόνο να τονίσω κάτι και πάλι, την σπουδαιότητα του να βρούμε λύσεις για τον κοινωνικό διάλογο. Διότι παρέχεται και πρέπει να διασφαλίσετε μια σωστή ισορροπία <clears throat> σε όσους ε, ε, επιθυμούν να ακολουθήσουν αυτή την πορεία. Και για το win-win ως ε, δηλαδή λύσεις, δηλαδή εποφελείς λύσεις για όλους, στην πλευρά του win-win. Δηλαδή αν υπάρξει μια συμφωνία θα εφαρμοστεί λέει από όλους. Δεν είναι τόσο απλό. Χρειάζεται να ευαισθητοποιήσουμε. Πρέπει να δείξουμε ποιο είναι το δυναμικό αυτής της win-win κατάστασης. Να δείξουμε και να αποδείξουμε πώς πρέπει να γίνουν όλα αυτά. Και να βοηθήσουμε να υπάρξει υλοποίηση αυτών των λύσεων με τον καλύτερο τρόπο έρευνα, παραδείγματα, διάχυση στοιχείων και γνώσεων που μπορεί να είναι υποφελής για τους κοινωνικούς εταίρους ε, και για τη διαμόρφωση των πολιτικών που απαιτούνται. Και για κάποια από τα θέματα που αναφέρθηκαν από διάφορους συμμετέχοντες, ο Αλεχάνδρο Θέρκας ανέφερε ένα θέμα για το πώς ε, θα είναι το μέλλον της Ευρώπης Πώς μπορεί να έχει μέλλον η Ευρώπη χωρίς το κοινωνικό πρότυπο. Εδώ φυσικά κάνουμε λόγο για προσαρμογές, δεν κάνουμε λόγο για αμφισβήτηση αυτού του προτύπου, αλλά επίσης για το ερώτημα ποια άλλα πρότυπα ανταγωνιστικότητας θα θέλαμε ή ποιο πρότυπο ανταγωνιστικότητας θα ήταν εφικτό για την Ευρώπη που πρέπει να αναζητηθεί. Και σε σχέση με το ζήτημα της κυρίας Κοστέλο για κάποιες αντιφάσεις μπορούμε να κάνουμε λόγο και καμιά φορά με θετικές διατυπώσεις ε, φιλικές για την ανάπτυξη, φορολογικές ε, προτάσεις. Ε, πρέπει ο προϋπολογισμός να λαμβάνεται υπόψη σε σχέση με τις ανάγκες και να δούμε τα trade-offs, δηλαδή τα ωφέλη που μπορούν να απορρεύσουν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και τώρα η Κρίστα Ζέτλατσεφ. Ευχαριστώ. Θέλω να επανέλθω σε κάποια από τα θέματα που ακούστηκαν ήδη και μετά θα συμπληρώσω αυτά που είπε η Γιόν. Έχουμε στοιχεία και αρκετές μελέτες ότι οι επενδύσεις στους ανθρώπινους πόρους είναι επικερδής. Εμείς θα συνεχίσουμε να συλλέγουμε στοιχεία για να αποδεικνύουμε ότι οι επενδύσεις στην υγεία, στην εκπαίδευση, στην κατάρτιση είναι, προσ... είναι επικερδείς και προσοδοχώρες. Έχουμε στοιχεία, το τονίζω. Υπάρχουν αρκετές μελέτες, το είπε και η κυρία Πέκα, και πρέπει όλα αυτά που ξέρουμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Ένα άλλο θέμα στο οποίο θέλω να επανέλθω είναι η απλούστευση της νομοθεσίας. Φυσικά ξέρουμε ότι η κατάσταση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των μικρών επιχειρήσεων είναι δεινή, ειδικά σε εποχές οικονομικής πίεσης. Προσοχή όμως να μην ε, δημιουργήσουμε δύο ομάδες εργαζομένων, ούτε δύο ομάδες επιχειρήσεων. Συμφωνώ ότι αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να βοηθήσουμε τις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να εφαρμόσουν την νομοθεσία. Και η αξιολόγηση της νομοθεσίας θα δείξει ότι ίσως υπάρχουν και διαφορετικοί νέοι τρόποι χρησιμοποίησης νομοθεσίας. Είναι σημαντικό πάντως να βοηθήσουμε ε, για την δημιουργία εργαλείων, ειδικά για τις μικρές επιχειρήσεις, για να μην δημιουργήσουμε δύο ομάδες εργαζομένων διακριτές. Ένα άλλο θέμα που αναφέρθηκε θα ήθελα να το σχολιάσω. Υπάρχουν επίσης στοιχεία ότι ακόμα και οι κακές επιχειρήσεις με κακό ρέκορτ στην υγεία και την ασφάλεια, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα δεν θα επιβιώσουν. Έχω πολλά παραδείγματα μεγάλων επιχειρήσεων, α πούμε στη Γερμανία, που δεν επέζησαν, δεν επιβίωσαν. Οι όροι εργασίες, οι συνθήκες εργασίας ήταν τόσο άσχημες που φαινόταν για μας με γυμνό μάτι ότι δεν θα επιβιώσουν. Και τελικά ούτε οικονομικά αποδείχθηκαν βιώσιμες. Χωρίς ε, υγιές και κινητοποιημένο γεμάτο ζήλο προσωπικό δεν επιβιώνουν οι επιχειρήσεις κάτι που είπαμε όλες οι υπηρεσίες, ότι αν δεν χρησιμοποιήσουμε το κοινωνικό διάλογο, οτιδήποτε και να κάνουμε, δεν πρόκειται να τα καταφέρουμε. Δεν πρόκειται να μπορέσουμε να συνεισφέρουμε στην ευρωπαϊκή κοινωνία. Μαντλέν Σέρμπαν και συνεχεία θα δώσω το λόγο στον Υπουργό. Η Σέρμπαν. Ευχαριστώ να τονίσω πόσο σημαντικό είναι το ευρωπαϊκό μοντέλο για τις ε, γειτονικέ χώρες. Φυσικά δεν είναι τέλειο. Πόρο απέχει από την τελειότητα. Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις για το πώς πρέπει να συνεχίσουμε. Αλλά αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι τα ελάχιστα πρότυπα ε, αυτά μας βρίσκουν όλους σύμφωνους. Μιλώντας για το ευρωπαϊκό οικονομικό, κοινωνικό μοντέλο, δεν νομίζω ότι είναι θέμα έτσι, θεωρίας και ακαδημαϊκό. Το θέμα είναι η δράση και η εφαρμογή. Και εδώ μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά ανάμεσα στον, στον ορισ... σε επίπεδο πολιτικής και στην εφαρμογή της. Δεν αρκεί να δηλώνουμε ότι έχουμε ένα ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο, πρέπει να το εφαρμόζουμε κιόλα. Εάν θεωρηθούμε καλή, αυτό θα πρέπει να, να φανεί, να αποδειχθεί με βάση τα αποτελέσματά μας. Και ποιος θα αποδεικνύει αυτό, η ίδια η αγορά. Επίσης, κάποιος βουλευτής ε, ζήτησε δράση για να δούμε ε, τι, κάνει, τι κάνουν οι προσπάθειές μας. Στην Ευρώπη πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι στο μέλλον θα έχουμε ε, μία γυράσκουσα κοινωνία όπου θα χρειάζεται ε, παρόλα αυτά κάποια προσόντα. Ε, όταν συγκριθούμε με την ε, Αφρική και με το Μαγκρέμπ, η τα δημογραφικά δεδομένα είναι τελείως διαφορετικά. Στην περίπτωση της Μολδαβίας, οι μελέτες δείχνουν ότι οι μετανάστες και ειδικά οι εξειδικευμένοι δεν θεωρούν ότι είναι ο πιο ελκυστικός προορισμός η Ευρώπη. Να σκεφτούμε γιατί οι ταλαντούχοι άνθρωποι από τι γειτονικέ χώρε δεν θέλουν να έρθουν στην Ευρώπη, αλλά ψάχνουν άλλους προορισμούς. Ίσως έχουμε κάποιο εμπόδιο, πρέπει να τα κατεδαφίσουμε. Θέλουμε να φαινόμαστε ως οι μεγαλύτεροι δωρητές στον κόσμο. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να επενδύουμε περισσότερο στο εξωτερικό, στους τομείς που μας ενδιαφέρουν. Τώρα θα δώσω το λόγο στον Υπουργό και συνεχεία και στους υπόλοιπους. Έχουμε λίγο χρόνο. Κρίστα, να σα ρωτήσω κάτι. Η... Ποια είναι η απάντηση στην ερώτηση της Μπένα Αράμπα. Μπένα Αράμπα. Ας πούμε, είπατε ότι πρέπει να δούμε τις ε, ανταγωνιστικές επιχειρήσεις. Η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων εξασφαλίζεται από τις ε, συνθήκες εργασίας, ε, στον χώρο εργασίας. Υγεία, ασφάλεια και καλές συνθήκες. λέμε ότι είναι στοιχείο ανταγωνιστικότητα, αλλά υπάρχουν ε, επιχειρήσεις που είναι τόσο ανταγωνιστικές και όμως δεν έχουν αυτές τις προϋποθέσεις, δεν, είναι ούτε, δεν υπάρχει ούτε ασφάλεια, ούτε υγεία στον χώρο εργασία, ούτε είναι καλέ συνθήκες εργασίας. Πώς συμβαίνει αυτό, αφού ισχύει, λέτε ότι ισχύει κάτι τέτοιο. Ε, Παρ' όλα αυτά γνωρίζω τα σχετικά με τους όρους και προϋποθέσεις απασχόλησης σε σχέση με την Amazon. Γενικά όμως θα έλεγα ότι υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα οι επιχειρήσεις δεν θα επιβιώσουν στην αγορά αν δεν βελτιώσουν τους όρους απασχόλησης των εργαζομένων τους. Είχαμε διάφορες επιχειρήσεις στη Γερμανία και επειδή τότε εργαζόμουν στο Βερολίνο το γνωρίζω αυτό και μπορούσαμε τότε ήδη να αναγνωρίσουμε ότι οι κακοί όροι απασχόλησης σήμερα είχα σαν επακόλουθο υψηλότερα ποσοστά ατυχημάτων, μεγαλύτερες απουσίες, μακροχρόνιες απουσίες από τον χώρο εργασίας λόγω ασθένειας ή ατυχήματος και όλα αυτά δεν ήταν ανταγωνιστικά στοιχεία για μια επιχείρηση. Είναι αρνητικά και πρέπει να καταπολεμηθούν. Γενικά πρέπει να διασφαλίσουμε ότι δεν γίνεται χωρίς επενδύσεις να τα καταφέρουμε και δεν μπορούν να επιβιώσουν αυτές οι επιχειρήσεις. Δεν είχα επαφή με τους εργαζόμενους ε, ή τους εκπροσώπους αυτών των επιχειρήσεων. Όμως γενικά πρέπει και μπορούμε να το πούμε. Γενικά αυτά είναι τα συμπεράσματα της έρευνας και αυτά είναι τα τεκμήρια τα οποία η επιστήμη καταδεικνύει. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ, ίσως εσείς θα μπορούσατε να μας πείτε. Τι συμπεράσματα βγάζετε από αυτή τη συζήτηση και ποιο είναι το τελευταίο μήνυμα που θέλετε να μας περάσετε. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Σε ευχαριστώ Πρόεδρε. Πολύ προσεκτικά άκουσα σε αυτή τη συζήτηση τα όσα αναφέρθηκαν και τα παρακολούθησα εκ του σύνεγγυς. Κάποιες ερωτήσεις ε, σε σχέση για παράδειγμα με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό και Οικονομικό Πρότυπο τα οποία συνεισέφεραν στη συζήτηση και εμπλούτησαν τη συζήτηση. Είναι ένα θελκτικό ελκυστικό πρότυπο για όλα τα γειτονικά κράτη αυτό το κοινωνικό πρότυπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ο πυρήνας και ο κινητήρας ε, της επιτυχίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δυστυχώς έχω περιορισμένο χρόνο στη διάθεσή μου και δεν μπορώ να επισέλθω σε όλες τις λεπτομέρειες και σε όλα τα στοιχεία. Αλλά κάποια σημαντικότερα στοιχεία θα μπορούσα να τα τονίσω. Η αηφορία αυτού του κοινωνικού προτύπου ως πρώτο. Ιδιαίτερα η αηφορία όσον αφορά την σημερινή οικονομική συγκυρία είναι πολύ σημαντικό πράγμα διότι είναι δαπανηρό αυτό το πρότυπο, κοστίζει στις επιχειρήσεις το να, να το διατηρήσουν και να το διασφαλίσουν. Το κράτος λοιπόν πρέπει να δαπανίσει κονδύλια ώστε να διασφαλιστεί αυτό το κοινωνικό πρότυπο. Γι' αυτό είναι σημαντικό να συζητήσουμε όλα αυτά τα ζητήματα. Δεύτερον, κάποιος ρώτησε πώς θα βρούμε λέει αυτή την, αρμονική σχέση μεταξύ ανταγωνιστικότητας όσον αφορά τις επιχειρήσεις και την ανταγωνιστικότητα γενικότερα όσον αφορά την οικονομία μιας χώρας και πώς θα μπορούν να διαδράσουν οι κοινωνικοί εταίροι. Πιστεύω ότι η αηφορία του ευρωπαϊκού οικονομικού προτύπου φτάνει στα όρια του, στα όρια της σήμερα αυτή η αηφορία αν επικεντρωθούμε και δούμε μόνο τους κοινωνικούς εταίρους και βασιστούμε μόνο σε αυτούς. Αυτό όμως που επιθυμούμε εμείς να κάνουμε είναι να δημιουργηθεί απασχόληση μέσα στα πλαίσια αυτού του κοινωνικού προτύπου. Έτσι δεν είναι. Να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης. Ένα από τα αίτια της οικονομικής ε, κρίσης πρέπει να το ομολογήσουμε και να το αναγνωρίσουμε με ειλικρίνεια, ευθέως. Ασκήθηκαν πιέσεις ε, τους δημόσιους ε, προϋπολογισμούς, στα δημοσιονομικά γενικότερα, ιδιαίτερες πιέσεις. Και πρέπει να πούμε, αν δεν ε, μπορέσουμε να ανακουφίσουμε αυτή την κατάσταση και δεν θέσουμε αλλού το κέντρο βάρους και δεν δημιουργήσουμε θέσεις απασχόλησης με λιγότερο γραφειοκρατικό βάρος, με λιγότερες ρυθμίσεις και λιγότερο περίπλοκο χαρακτήρα δεν θα στεφθεί με επιτυχία το εγχείρημά μας. Χρειαζόμαστε επενδυτές που μέσα σε ένα φύλλο επιχειρησιακό πλαίσιο θα μπορέσουν να δράσουν. Ένα περίγυρο και ένα περιβάλλον θετικό ώστε να υπάρξουν κίνητρα και προϋποθέσεις ώστε να μπορέσουν να βρουν κίνητρα και να μπορέσουν να λειτουργήσουν θετικά και οι εργαζόμενοι να έχουν και κίνητρα και να μπορέσουν να είναι και πιο παραγωγικοί. Όλα αυτά που κρυσταλώθηκαν και απέρευσαν από τη συζήτηση που, που ε, διεξαγάγαμε και είναι γεγονός ότι χρειάζεται μια πιο θετική και ενεργός πολιτική από πλευρά των κυβερνήσεων. Δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση. Η εναλλακτική λύση θα ήταν να επιβαρύνονται ακόμα περισσότερο οι επιχειρήσεις, να δαπανώνται ακόμα ακόμα μεγαλύτερα, περισσότερα κονδύλια και να επιβαρύνονται ακόμα περισσότερο οι, τα δημοσιονομικά για τη διασφάλιση του κοινωνικού προτύπου. Αυτό επιβαρύνει όμως τις επιχειρήσεις και επιβαρύνει και τους πολίτες με υψηλότερη φορολογία και μεγαλύτερες εισφορές. Θα μπορούσαμε με καλύτερες επενδύσεις, βελτιωμένες επενδύσεις στην τεχνολογία και στο ανθρώπινο δυναμικό να καταφέρουμε να, να βελτιώσουμε την κατάσταση πιο αποτελεσματικά. Προσπαθούμε λοιπόν με άλλα λόγια από την πείρα άλλων χωρών και από την εμπειρία που έχουν συλλέξει να δούμε τι μπορεί να γίνει. Να δημιουργήσουμε ένα θετικό για τις επιχειρήσεις πλαίσιο ώστε να επιτύχουμε επενδύσεις στην καινοτομία και επενδύσεις στο ανθρώπινο δυναμικό που θα καταστούν εφικτές. Γιατί χωρίς επενδύσεις από τον ιδιωτικό τομέα θα βρισκόμαστε στο ίδιο σημείο, θα ε, ε, είμαστε αποτελματωμένοι στο ε, ίδιο σημείο και θα κάνουμε βήμα σημειωτών χωρίς να μπορούμε να σημειώσουμε πρόοδο. Φυσικά το κράτος πρέπει να ενεργοποιείται αλλά υπέρ των εργαζομένων και υπέρ των επιχειρήσεων. Ένα ενεργό κράτος, ε, είναι σημαντικό το επαναλαμβάνω πάντα αυτό, ενεργό κράτος υπέρ των επιχειρήσεων και των εργαζομένων. Αν θέλουμε να είναι αποτελεσματικές οι επιχειρήσεις μας τότε πρέπει να προστατεύονται οι πολίτες, να μπορούν να προστατεύονται επαρκώς ώστε να διασφαλίζονται οι όροι εκείνοι που να διασφαλίζουν ε, ασφαλείς και αηφόρες θέσεις απασχόλησης. Δεν επιτρέπεται όμως μόνο στην προστασία να επενδύει το κράτος. Πρέπει να ανακουφίζονται και οι επιχειρήσεις, να ανακουφίζονται ώστε να απελευθερώνονται κεφάλαια για την βελτίωση των όρων εργασίας και απασχόλησης των εργαζομένων. Η καινοτομία των στις επιχειρήσεις πρέπει να προαχθεί, ώστε οι άνθρωποι να τύχουν κινήτρων, να δοθούν κίνητρα στους ανθρώπους, να δημιουργήσουν μια διαφορετική νοοτροπία νοοτροπία υπέρ της εργασίας και υπέρ της παραγωγής ώστε να είναι θετικό και να μπορούν οι πολίτες να το θεωρούν ότι είναι θετικό να εργάζονται παραγωγικά. Κάπως χάθηκαν νομίζω και παραμελήθηκαν αυτές οι αξίες σε σχέση με τους πολίτες μας και πρέπει αυτά να αναζωογονηθούν και να στηριχθούν σε ένα κοινωνικό διάλογο, σε ένα πλαίσιο κοινωνικού διαλόγου. Να δουν οι κοινωνικοί εταίροι και να γνωρίζουν ποιος θα συνεισφέρει και με ποιο τρόπο σε αυτόν τον κοινωνικό διάλογο και τι θα, πετυχε... θα πετυχαίνουμε ο καθένας από εμά σε αυτόν τον κοινωνικό διάλογο. Συμμετοχή όλων με ένα πνεύμα ευθύνη και υπευθυνότητα όλων σε αυτόν τον κοινωνικό διάλογο. Αυτή είναι η σωστή πορεία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ε, παιδί μου. Θα δώσω το λόγο σε όσους βουλευτές ε, συμμετείχαν. Πρώτα στο Hans Becker για τη συνέχεια που θα δοθεί στη συζήτηση που κάναμε σήμερα το πρωί, γιατί πρόκειται για μια συνάντηση, ένα ραντεβού που είχαμε σήμερα το πρωί. Δεν είναι τυχαίο αν σήμερα το πρωί κάνουμε τη συζήτηση αυτή με τους τέσσερις οργανισμούς και με τους προσκεκλημένους μας. Παρόλο που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την επόμενη εβδομάδα, 2 Οκτωβρίου, έχει να δημοσιεύσει τη δικιά της συνεισφορά για την κοινωνική διάσταση της ΟΝΕ, η συζήτηση θα συνεχιστεί. Να μας πείτε λοιπόν τι συμπεράσματα βγάζετε και τι διδάγματα για τις μελλοντικέ μας εργασίες στα πλαίσια και τη συζήτηση που θα κάνουμε για την κοινωνική διάσταση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πρώτα γερμανικά και τώρα αγγλικά. Είναι ένα υψηλά σύνθετο και περίπλοκο ζήτημα αυτό ως θέμα για να είμαι σύντομος και για να ε, μιλήσω ειλικρινά και ευθέως. Συμβαίνει το εξής. Κατανοώ σίγουρα ότι βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου ένα ανώτατο επίπεδο θέμα, υψηλότατο επίπεδο θέμα μας απασχολεί κινείται γύρω από μας, εμάς αυτό τον περίγυρο. Η Κοινωνική Ένωση, η Κοινωνική Ευρωπαϊκή Ένωση. Ω σύμβολο το χρησιμοποιώ αυτό για όλες τις ιδιομορφείς και εξειδικευμένες προσεγγίσεις για τα διάφορα θέματα τα οποία συζητούμε εδώ σήμερα. Πώς θα έχει το μέλλον, πώς θα διαμορφωθεί το μέλλον και όπως είπα για να είμαι σύντομος, πιστεύω ότι δεν βρισκόμαστε σε μια θέση όπου αυστηρά και σοβαρά να μπορούμε να εργαστούμε για μια κοινωνική ένωση. Είμαι απόλυτα βέβαιος ότι ο τρόπος με τον οποίο εργαστήκαμε μέχρι σήμερα κατά το παρελθόν με τις δομές τις σημερινές θα πρέπει να βελτιστοποιήσουμε με τον καλύτερο τρόπο το έργο μας ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις σημερινές προκλήσεις και τις μελλοντικές προκλήσεις εξίσου. Διότι, διότι θεωρώ ότι μια η Δημοσιονομική Ένωση, ε, Φορολογική και ε, Οικονομική Ένωση. Θα πρέπει να σχεδιαστούν και να κατατιστούν εξειδικευμένα και να αναγνωριστούν στη σπουδαιότητά τους προτού κάνουμε λόγο για όλα αυτά. Κάνω λόγο για αυτήν την κοινωνική ένωση και ενότητα, διότι δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία και θέλω να είμαι σύντομος για τους στόχους των ιδρυμάτων και οργανώσεών μας και οργανισμών μας που ακούσαμε να τίθενται επί τραπέζι σήμερα και το έργο μας στην δική μας Κοινοβουλευτική Επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου είναι στη σαφή αυτή κατεύθυνση να αυξηθεί η κοινωνική αλληλεγγύη σε αυτή την κοινωνική Ευρώπη. Για αυτούς όλους τους λόγους δεν θέλω να απολέσουμε χρόνο, να μην χάσουμε χρόνο ε, και ε, ε, έργο και αποτελεσματικότητα. Είμαστε τόσο ισχυροί όταν είμαστε ενωμένοι για να συζητήσουμε τις ε, ανωτέρου επίπεδου στρατηγικές που μέχρι σήμερα δεν ε, υλοποίησαν αυτούς τους στόχους επαρκώς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Κίνγκα Κόντς τώρα. Και ποιος άλλος. Κίνγκα Κόντς πρώτα. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι αυτό που μαθαίνουμε από τη σημερινή συνάντηση είναι ότι δεν έχουμε να διαλέξουμε ανάμεσα στην κοινωνική προστασία, το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο και την ανταγωνιστικότητα. Μπορούμε κάλλιστα να έχουμε και τα δύο. Να έχουμε ανάπτυξη μέσα από επενδύσεις και εφόσον υπάρχει ανάπτυξη μπορούμε να επενδύσουμε στο κοινωνικό μας μοντέλο. Αν κληθούμε να επιλέξουμε, αυτό είναι λάθος. Νομίζω ότι αυτό είναι το μήνυμα που βγήκε από όλες τις πλευρές σήμερα. Και συμφωνώ απόλυτα και για το ότι η αλληλεγγύη είναι κάτι από το οποίο δεν πρέπει να παραιτηθούμε. Βλέπουμε όλο και λιγότερη αλληλεγγύη σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εμείς όμως πρέπει να επιμείνουμε σε αυτήν. Είναι η μόνη διέξοδος. Αυτό. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Κυρία Μακεντά. Ευχαριστώ. Ειλικρινά με εξέπληξαν τα τελευταία σχόλια του Υπουργού και συμφωνώ με τα περισσότερα όπω είπατε. ο κ. Γερουλεύσκο είπε, έκθεσε το, το ερώτημα, θέλουμε εξάρτηση για τον πλούτο ή θέλουμε ανταγωνιστικότητα, δημιουργία. Μα θέλουμε δημιουργία, από αυτήν όλοι έχουμε να αποφεληθούμε. Δεν θέλουμε να φτιάξουμε ένα κοινωνικό μοντέλο το οποίο να σας τραβάει προς τα κάτω. Όχι. Θέλουμε μια ελαφριά πινελιά. Θέλουμε να ενθαρρύνουμε τον κόσμο να επενδύσει, να αποκτήσει δεξιότητες και έτσι φτιάχνουμε μια ανταγωνιστική Ευρώπη, η οποία να μπορεί να ανταγωνιστεί τις μη ευρωπαϊκές χώρες. Όντως είμαστε στην παγκοσμιοποίηση. Οπότε ναι, χρειαζόμαστε ε, νέες σύγχρονες δεξιότητες. Δεν μπορούμε να κοιτάμε πίσω τα επαγγέλματα που κάποτε υπάρχουν. Όχι, αλλάζει η αγορά εργασίας. Ο ευρωπαϊκός τρόπος εκπόνησης πολιτικής πρέπει να ανταποκρίνεται στις σημερινές ανάγκες. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε επίσης πολύ τις ε, μελέτες αντικτύπου σε όλους τους τομείς. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Πράγματι είναι αυτή μια πολιτική διάσταση που βάζετε στη σημερινή συζήτηση. Και αντιλαμβάνομαι ότι οι ευρωβουλευτές που καταλήγουν σε συμπεράσματα το κάνουν βάσει της πολιτικής τους δέσμευσης από τη δικιά τους πολιτική οικογένεια, χωρίς να αντικατοπτρίζουν το συλλογικό μας έργο, βέβαια, ως Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Αλλά είναι λογικό σε αυτή τη συζήτηση. Τώρα από τους τρεις προσκεκλημένους ε, θέλουν όλοι φαντάζομαι να πάρουν το λόγο, οπότε για ένα-δύο λεπτά το πολύ ο καθένας παρακαλώ. φέρετε το φασίζω όλα έτσι είναι, με την ίδια σειρά. Ούβε Κόμπιχαουν, πρώτα για δύο λεπτά. Παρακαλώ. Thank Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Και πάλι για άλλη μια φορά. Συγχαίρω για την διοργάνωση αυτής της εκδήλωσης που ήταν ιδιαίτερα εμπλουτιστική και ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα σε υψηλά πολιτικά επίπεδα. Κρίμα που έφυγε ο κύριος Σέρκας, διότι θα ήθελα να υπογραμμίσω και αυτό το οποίο αναφέρθηκε και από τον συνάδελφο. Δεν είναι δική μας δουλειά ή να πει η Επιτροπή τι θα γίνει με τις επιχειρήσεις. Πρέπει να έχουμε μια νέα προσέγγιση συνολικά για τις επιχειρήσεις με κανόνες και ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Σε σχέση με τα όσα είπε η κυρία Φίσμπαχ, δεν είμαστε κατά εμείς της κοινωνικής διάστασης καθόλου. Αλλά όπως είπε η κυρία Μακίνταερ, δεν υπάρχει μονολυθική μονοδρομική προσέγγιση, μονοβαρής προσέγγιση σε σχέση με ένα πρότυπο ισοπεδωτικό και μπορώ να, να επαναλάβω αυτό το οποίο αναφέρθηκε. Αυτά τα οποία δαπανούμε στην Ευρώπη σε σχέση για παράδειγμα με τον υπόλοιπο κόσμο στα ποσοστά αυτά και όσον αφορά και το πακέτο για την απασχόληση πρέπει να δούμε και το κόστος ε, που συνεπάγονται και σε σχέση με τον κύριο Άντερς ε, να δούμε το κόστος, ε, το εργατικό, το εργασιακό κόστος και τις δαπάνες και τέλος η κρίση έδειξε ότι όταν υπάρχουν ελαστικές αγορές για την προσαρμογή μας στις ανάγκες τους και αν και όταν μπορεί να λειτουργήσει ο κοινωνικός διάλογος είμαστε ιδιαίτερα αποτελεσματικοί για την διαχείριση και αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης ερωτήσεις. Ολοκλήρωσα. Ευχαριστώ. Ε, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Σε σχέση με την Amazon, τουλάχιστον στη Γερμανία, οι εργαζόμενοι προχώρησαν σε απεργία και προσπαθούν να πετύχουν την αναγνώριση ε, μισθών που να ισχύουν στον τομέα Να ένα παράδειγμα λοιπόν σχέσεων εργοδοσίας εργαζόμενων. Ένα άλλο πράγμα που θέλω να πω είναι ότι η δικιά μου η σύλληψη της ανταγωνιστικότητας βασίζεται στην ποιότητα των προϊόντων μας, στην δυνατότητα να καινοτομήσουμε, αλλά και στην θετική διάθεση των εργαζόμενων και στην ικανότητά τους να προσαρμόζονται. Οπότε οι δυνατότητες που έχουμε για την ανταγωνιστικότητα δεν έχει να κάνει τόσο με το ανταγωνιστικότητα με οποιοδήποτε τίμημα, κοινωνικό για παράδειγμα, όχι. Τέλος, όσον αφορά τις επενδύσεις. Νομίζω ότι στην ευρωπαϊκή πολιτική πρέπει πια να καταλάβουμε ότι η λιτότητα δεν λειτουργεί. Ότι υπάρχει δυνατότητα για πολλές επενδύσεις, ανθρώπους, υπηρεσία, σε απασχόληση Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα όπου, όπως το είπε και ο κύριος Τζον, επενδύεις ένα ευρώ και τελικά παίρνεις πίσω πολύ περισσότερα. Αυτό είναι το μήνυμα που πρέπει να βγει. Πρόεδρο, σε ευχαριστούμε πολύ, Ριγκό. Και ήρθε και ο Επίτροπος και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθε. Εγώ θα φύγω πριν ολοκληρώσουμε, οπότε τον χαιρετώ εδώ. Εκείνος θα σας παρουσιάσει πώς γίνονται οι συζητήσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα απαντήσει ίσως και στις ερωτήσεις που θα ακουστούν τώρα. Δικό Ποντουάν λοιπόν, δύο λεπτά. Ευχαριστώ για την Amazon, μια που εδώ συζητήθηκε αρκετά. Είναι ενδιαφέρον, είναι μια ανταγωνιστική επιχείρηση, ναι, αλλά τι βαθμό ανταγωνιστικότητας έχει στον κλάδο της, δεν ξέρω, οι αρχές για τον ανταγωνισμό θα απαντήσουν σε αυτό. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να το κρίνει κανείς όπως και με τις επιχειρήσεις, οι αεροπορικές εταιρείες και έχω πολλές να συγκρίνω. Με την Amazon ίσως είναι λιγότερο. Πρέπει να συγκρίνει κανείς για να μπορεί να πει τελικά ποιο είναι ανταγωνιστικό και ποιο όχι. Έτσι κι αλλιώς δεν είναι όλα άσπρο ή μαύρο. Σίγουρα υπάρχει περιθώριο για κοινωνικό διάλογο, για την ε, οργάνωση των εργαζομένων και να προσπαθήσουν να λύσουν το προβλήματα όσο γίνεται καλύτερα οι τέσσερις οργανισμοί εδώ εννοείται ότι πρέπει να πούν τι πρέπει να γίνει. Να κάνουν το κήρυγμα για κάποιο τρόπο. Δώσαμε παραδείγματα εδώ, τα είπε και η κυρία Γκόντς. Θα έπρεπε επιχειρήσει να καταλάβουν ότι όταν έχουν στα διοικητικά συμβούλια και στα εκτελεστικά τους όργανα επιχειρήσεις γυναίκες, ανεβαίνει η αποτελεσματικότητά τους και η παραγωγικότητά τους για να καταργηθεί η διάκριση που γίνεται πολλές φορές σε βάρος των γυναικών. Και το τελευταίο που θέλω να πω. Εντάξει, μπορεί και εγώ να προσπάθησα να σας προκαλέσω εδώ σήμερα και μπορώ να το κάνω και ακόμα πιο πολύ, αλλά πάντως δούλευα στη Νέα Υόρκη και από εκεί με απέσπασαν στις Βρυξέλλες από όπου και έρχομαι. Στο μεταξύ έχουν επιδεινωθεί οι συνθήκες εργασίας μου τώρα που ήρθα στις Βρυξέλλες παρόλο που πρόκειται για μια κοινωνία που θεωρείται πάρα πολύ καλή στο χώρο εργασίας κτλ. Και αναρωτιόμουν γιατί, ποια είναι η διαφορά. Μα στη Νέα Υόρκη, αν δεν ήμουν ικανοποιημένο από τη δουλειά μου, πήγαινα στο αφεντικό μου και του έλεγα δεν μ' αρέσει και πήγαινα σε μια άλλη επιχείρηση. Εδώ είναι πολύ πιο δύσκολο να το κάνω αυτό. Μπορούμε να το συζητήσουμε περισσότερο, αλλά ποιο είναι το ηθικό δίδαγμα. Δεν λειτουργούμε εν κενό. Το περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργούμε έχει πολύ μεγάλη σημασία. Το κατά πόσο δηλαδή οι εργαζόμενοι έχουν την ευκαιρία να αλλάξουν, να βρουν μια άλλη δουλειά. Αυτό πρέπει να το δουλέψουμε περισσότερο εδώ στην Ευρώπη. σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ όλους τους οργανισμούς που ήρθαν Κύριε Αντιπρόεδρε της ε, Κυβέρνησης της Μολδαβίας, σας ευχαριστούμε και σας πολύ για τη δικιά σας συνεισφορά στη συζήτηση. Ευχαριστώ και όλους τους συναδέλφους βέβαια που πήραν το λόγο. Τώρα έχω να κάνω κάποιες παρατηρήσεις, οι οποίες εννοείται ότι δεν δεσμεύουν ολόκληρη την Επιτροπή μας. Εδώ η συζήτηση γίνεται ανοιχτά. Αλλά θέλω να πω ότι όσον αφορά το θέμα του κοινωνικού διαλόγου και την καινοτομία στον χώρο εργασίας, στην εκπαίδευση, δεν υπάρχει διαφωνία μεταξύ μας όσο μένουμε στα γενικά. Όταν όμως πηγαίνουμε στα συγκεκριμένα, τι σημαίνει αυτό για την εξέλιξη των συστημάτων, τότε τίθεται το ζήτημα τι μέσα θα χρησιμοποιήσουμε, τι εργαλεία. Και εκεί είναι το μεγάλο διακύδευμα. Με ξέπληξε πολύ αυτό που είπε ο Μποντουά Ριγκό πριν από λίγο. Και ο Βεκομπούρ επίσης το είπε ότι τελικά πρέπει να αφήνουμε ήσυχε τις επιχειρήσεις. Εντάξει, μπορεί να υπερβάλλω, αλλά εγώ έχω δει σε πολλούς τομείς τις επιχειρήσεις που λένε αφήστε μας ήσυχους και έτσι καθορίζουν μόνες τους τις συνθήκες κτλ. Αυτό λέγεται αυτοπιθαρχία. Και είδαμε που οδήγησε αυτό. Κύριε Ποντουάν Ριγκό, είπατε, για παράδειγμα, ότι στα διοικητικά συμβούλια όταν έχουμε περισσότερες γυναίκες τότε είναι πιο αποτελεσματικές ναι. επιχειρήσεις. Ε, ωραία, μια που μάθαμε λοιπόν ότι είναι πιο αποτελεσματικές, ε, τότε να το αποδείξουμε. Αν ο νομοθέτης μπορεί να παρέμβει για να βοηθήσει πιο πολύ προς το δρόμο της αποτελεσματικότητας και να δώσει ένα κίνητρο για να το κάνουν επιχειρήσεις, ε, δεν θα ήταν κακό. Άρα νομίζω ότι έχει τη σημασία του να παρέμβουμε. Η κυρία Μακεντάιρ τώρα που αναφέρθηκε στην ανάπτυξη, φυσικά και τη χρειαζόμαστε την ανάπτυξη, αλλά βγαίνουμε από μία περίοδο δεκαετή όπου είδαμε τι σημαίνει τρελή ανάπτυξη. Αν λοιπόν δεν διοχετεύσουμε σωστά την ανάπτυξη, αν δεν μπούμε τα κέρδη από την ανάπτυξη, η προσθέμενη αξία της ανάπτυξης θα πρέπει να χρηματοδοτούν το κοινωνικό μοντέλο, τότε η ανάπτυξη αυτή ενισχύει τους κερδοσκόπους και μόνο. Πράγμα το οποίο δεν νομίζω ότι θέλει κανένας από εμά. Κύριε Αντιπρόεδρε της Κυβέρνησης. Εξεπλάγει από πολλά που είπατε σήμερα το πρωί. Ιδιαίτερα όταν είπατε ότι η ανταγωνιστικότητα στο κάτω-κάτω πρέπει να τίθεται σε επίπεδο χώρας. Αν η ανταγωνιστικότητα είναι διακύδευμα για τη χώρα, τότε όλοι οι φορείς πρέπει να αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους και δεν μπορεί να λύνεται το ζήτημα σε επίπεδο επιχείρησης και μόνο. Είπατε επίση ότι για σας υπάρχει ένα θέμα που σοκάρει. Είπατε επιλέξει το και τα δικαιώματα των εργαζομένων σας στο εξωτερικό δεν ε, είναι εγγυημένα. Αυτή είναι μια άλλη συζήτηση που έχουμε στην Επιτροπή μας αυτή. πολύ ουσιαστικό αυτό που είπατε. Έπειτα για τον κοινωνικό διάλογο, και ελπίζω εδώ να μην προδίδω τη σκέψη σας, αλλά είπατε νομίζω ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να μάθουν τι σημαίνει κοινωνικός διάλογος. Εμείς πρέπει να το πάρουμε αυτό το δίδαγμα από αυτά που λέτε. Επίσης, εγώ θυμάμαι και τον πρόεδρο Μπαρόσο, όταν ε, παρουσίασε την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2012. Δεν το ξαναπέφετος αλλά πέρυσι στην ε, ομιλία του αυτή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Ολομέλεια, είπε ότι το θέμα του κοινωνικού μοντέλου είναι θέμα ανταγωνιστικότητας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ νομίζω ότι αυτό πρέπει να το λέμε και να το ξαναλέμε. Δεν συμφωνώ πάντα με τον πρόεδρο Μπαρόζο, αλλά από αυτού, ναι, είναι κάτι βασικό. Και για να το πετύχουμε εδώ σας δίνω την προσωπική μου άποψη που συμμερίζονται όμως πολλοί εδώ, αλλά όχι όλοι. Το θέμα του πώς γίνεται ανταγωνιστικότητα. Δεν πρέπει να τη βλέπουμε μόνο ως κόστος εργασίας. Τέλος, θέλω να ανοίξω εδώ δύο νέους ορίζοντες που σχετίζονται με αυτά που συζητήσαμε σήμερα το πρωί και που έχουν να κάνουν με την νέα κατάσταση που αντιμετωπίζουμε και θα αντιμετωπίσουμε, το από και η κυρία Συνήθως σκεφτόμαστε την κατάρτιση, την μεταφορά γνώσης που ανήκει σε μια άλλη εποχή. Από διπλή άποψη. Πρώτον, επειδή η ανεργία ήταν αλλιώς, τώρα έχουμε τεράστια ανεργία Έχουμε συστήματα κατάρτισης που τα φτιάξαμε όταν η ανεργία δεν ήταν τόσο μαζική όπως είναι τώρα. Σήμερα έχουμε να κάνουμε με μια μαζική ανεργία με φαινόμενα μεταφοράς των επιχειρήσεων σε τέτοιο βαθμό που ποτέ δεν το είχαμε ξαναδεί αυτό πριν από 10 χρόνια. Το άλλο είναι η εξέλιξη στην τεχνολογία που επιταχύνθηκε με ρυθμούς που δεν τους ξέραμε όταν είχαμε φτιάξει τα πρώτα συστήματα επιμόρφωσης. Συνεπώς, η πρόκληση που αντιμετωπίζουμε είναι πρώτον τα συστήματα κατάρτισης που προτείνουμε να ξέρουμε ότι δεν είναι μόνο για να συνοδεύουν και να βοηθούν τους εργαζόμενους που είναι στην ανεργία προς την επόμενη θέση εργασίας τους. Όχι, είναι για να αντιμετωπιστεί αυτή η μαζική ανεργία που είναι μια άλλη διαφορετική πρόκληση για τα εκπαιδευτικά μας συστήματα. Όσον αφορά τώρα τις τεχνολογικές εξελίξεις, υπάρχει αυτό που ονομάζουμε mismatch, δηλαδή που δεν ανταποκρίνονται στην αγορά εργασίας τα εκπαιδευτικά μας συστήματα. Πολλές φορές όμως ακούμε ότι αρκεί να διορθώσουμε άπαξ το εκπαιδευτικό σύστημα για να ανταποκριθεί στις σημερινές ανάγκες της αγοράς εργασίας. Αλλά δεν πρόκειται μόνο για προσαρμογή προγραμμάτων, πρόκειται για αλλαγή στη μέθοδο. Γιατί αλλιώ θα τρέχουμε πάντα από πίσω για να προλάβουμε την καινοτομία και να προσαρμόσουμε την εκπαίδευση. Άρα είναι θέμα μεθόδου και πώς θα καταρτήσουμε τους ίδιους τους εκπαιδευτές δεδομένων των τεχνολογικών εξελίξεων. Συνεπώς, την Προεδρία τη δίνω στην Edith Bauer και δίνω το λόγο στον Επίτροπο, από τον οποίο ζητώ και συγγνώμη που δεν θα μπορέσω να παραμείνω για να τον ακούσω. Θα έχει και άλλες ευκαιρίες για να μου μεταφέρει τα κύρια μηνύματά του. Κύριε Επίτροπε, έχετε το λόγο. Uh, Πρόεδρε, αγαπητοί ευρωβουλευτές, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να συγχαρώ το Κοινοβούλιο και τις agencies αυτές που διοργάνωσαν αυτό το σεμινάριο και ζητώ συγγνώμη που δεν μπόρεσα να παραστώ από την αρχή. Αυτό όμως δείχνει τη θαυμάσια δουλειά που κάνουν οι υπηρεσίες αυτές βοηθούν την Κομισιόν, της δίνουν αποδεικτικά στοιχεία για μια πλειάδα πολιτικών. Η Κομισιόν και όσοι βασίζονται στις ε, δραστηριότητες των ε, υπηρεσιών αυτών ε, χαίρονται και αυτή τη δουλειά που κάνει η ΟΣΑ, το ΣΕΝΤΕΦΟΠ, το ETF ε, κτλ. Τα τελευταία πέντε χρόνια η Ευρώπη ε, έζησε τη μεγαλύτερη οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Σε αυτή την κρίση, το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο ήταν ένα μεγάλο ατού, προστάτησε του ανθρώπου από τι συνέπειε τη ε, οικονομική αναστάτωση. Μέσω του ισχυρού κοινωνικού διαλόγου σώθηκαν πολλέ θέσει απασχόληση και δόθηκαν ευέλικτε απαντήσει μέσα το, μέσω των αυτόματων κοινωνικών σταθεροτοποιητών το εισόδημα στην πρώτη φάση της κρίσης των εργαζομένων προστατεύτηκε. Και... Όμως η κρίση μας δίδαξε κάποια πράγματα. Μας δίδαξε ότι για να δημιουργήσουμε μια πιο ευημερούσα και μια πιο ανθεκτική κοινωνία, ένα κοινωνικό-οικονομικό μοντέλο πιο ανθεκτικό. Χρειαζόμαστε περαιτέρω βελτιώσει σε επίπεδο κρατών μελών, αλλά και σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση. Προφανώ, για να μπορέσουμε να βγούμε από την κρίση, η Ευρώπη πρέπει να αλλάξει, να διορθώσει κυρίω το επιχειρηματικό τη μοντέλο. Χρειαζόμαστε ε, καλή χρηματοπιστωτική ρύθμιση, χρειαζόμαστε καλύτερη πολιτική, πολιτική και και βιομηχανική πολιτική και πρέπει να μεταρρυθμιστεί και το ελληνικό μας μοντέλο. Επίσης, πρέπει να δούμε τι πρέπει να αλλάξουμε στο κοινωνικό μοντέλο. Η Ευρώπη πρέπει να κάνει πολλά, πολύ περισσότερα και όχι λιγότερα από ό,τι έκανε. Η δέσμευσή μας στους στόχους, ε, όπως εγγράφονται στη συνθήκη, δεν πρέπει να παραμεληθούν. Υπάρχει κοινωνική πρόοδος, με μια υψηλά ανταγωνιστική αγορά, με κοινωνική, θα πρέπει να υπάρξει κοινωνική και οικονομική συνοχή, καθώς και αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών. Πλήρης απασχόληση, μαζί με την κοινωνική πρόοδο, με μια πολύ ανταγωνιστική κοινωνική οικονομία. Αυτό αναφέρεται στο άρθρο 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το άρθρο λέει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να προωθήσει την ε, κοινωνική, οικονομική και εδαφική συνοχή και την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών. Ε, δημιουργεί μια ισορροπία ανάμεσα στην, στις ατομικές ε, ευθύνες των κρατών μελών και την αλληλεγγύη με, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση μιλάει και για τις ατομικές ευθύνες αλλά και για μια επιμερισμένη αλληλεγγύη. Η αλληλεγγύη στα κράτη-μέλη μπορεί να ενισχυθεί εάν ενισχυθεί η αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών. Και αυτό δεν πρόκειται να γίνει χωρίς ε, πιο ισχυρό ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να συνεργαστούν και τα εθνικά συστήματα κοινωνική προστασίας επλήγησαν μετά, μετά τα προγράμματα λιτότητας λόγω της κρίσης του χρέους το πακέτο για τα κοινωνικά, τις κοινωνικές επενδύσεις της Κομισιόν δίνει δυνατότητα να εκμοντερνιστούν τα συστήματα κοινωνικής προστασίας, να χρησιμοποιηθούν οι πόροι πιο αποτελεσματικά, ούτω ώστε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα όπως η φτώχεια των παιδιών ή οι άστεγοι. Ε, έχουν ξεκινήσει κοινωνικές μεταρρυθμίσεις για να βελτιωθεί η ακαταλληλότητα, η βιωσιμότητα και η ασφάλεια των συνταξιωτικών συστημάτων. Η πράσινη και η λευκή βίβλωση ήταν σημαντικές για να δώσουν τα σωστά επιχειρήματα και προσανατολισμούς για αυτές τις συζητήσει και τις μεταρρυθμίσεις μέσα στα κράτη-μέλη. Η... Το πακέτο, τα διάφορα πακέτα της Κομισιόν, όπως αυτό της, για την νεότητα, βοηθάει την κινητοποίηση των οικονομικών πόρων ε, και την καταπολέμηση της ανεργίας ε, ε, βασιζόμενη στα μοντέλα εκπαίδευση και κατάρτισης και μετάβαση από το σχολείο στη δουλειά. Η εγγύηση για την νεολαία και η πρωτοβουλία για τους νέους που χρηματοδοτούνται με 6 δισεκατομμύρια ευρώ δίνουν καλά παραδείγματα για το πώς η Ένωση μπορεί να αναλάβει συλλογική δράση για να αντιμετωπίσει συλλογικά τις μεγάλες κοινωνικές προκλήσεις με βάση συγκεκριμένα κριτήρια αναφοράς. Το, η εγγύηση για τους νέους θα βοηθήσει τους νέους, θα τους εξασφαλίσει καλύτερα, θα βοηθήσει να γίνουν πιο απασχολήσιμοι μακροπρόθεσμα, να αποφύγει να χάσουν δεξιότητες, δεξιότητες ε, εστιάζοντας τις ανάγκες και προσφέροντας στους νέους την σημαντική κατάρτιση ή τη μαθητεία μπορεί να συνεισφέρει στην καταπολέμηση της φτώχειας της Ευρώπης. Πιστεύω ότι αυτές οι πρωτοβουλίες θα βοηθήσουν την οικονομική ανάπτυξη και άμεσα, αλλά και θα βοηθήσουν ε, προς ε, την ε, μακροπρόθεσμη ανοικοδόμηση του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου. Άλλα τμήματα των προσπαθειών ανοικοδόμησης είναι από κάτω, έρχονται από κάτω προς τα πάνω και Φυσικά χρειάζεται και το κατάλληλο περιβάλλον. Φερρυπίν. Η κοινωνική οικονομία που σημαίνει ε, τις ασφαλιστικές εταιρείες, ε, τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, ε, τα διάφορα μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, ε, τις κοινωνικές επιχειρήσεις, ε, δίνει πολλές υπηρεσίες σε όλη την Ευρώπη και βεβαίως δημιουργεί και εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης. Το, τις δυνατότητες του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, ένα άλλο οικονομικό εργαλείο, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί καλύτερα από τα κράτη-μέλη, ούτω ώστε να αναπτύξουν περισσότερε κοινωνικέ επιχειρήσει και μια ευρύτερη κοινωνική οικονομία. Μια διάσκεψη που έγινε τον Ιανουάριο στο Στρασβούργο, ή μάλλον που θα γίνει στο Στρασβούργο, θα βοηθήσει πολλού ενδιαφερόμενου να συζητήσουν ε, κάτω από την ίδια στέγη. Και πιστεύω ότι η περιγραφή του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Μοντέλου θα είναι πλήρη αν δεν μιλήσουμε για την σημασία του κοινωνικού διαλόγου. Πρέπει να ενισχύσουμε την εμπλοκή των κοινωνικών εταίρων στη συζήτηση που γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τι πολιτικές και στη λήψη των αποφάσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, υποστήριξε τον ε, κοινωνικό διάλογο στα κράτη-μέλη μέσω της οικονομικής ε, βοήθεια για οικοδόμηση δυναμικού προ αυτήν την κατεύθυνση μεταξύ άλλων. οι διαβουλεύσεις με του κοινωνικού εταίρου σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορούν να γίνουν πιο αποτελεσματικέ. Ο στόχο θα ήταν να έχουμε διαφανεί και αξιόπιστες ε, διαδικασίες διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Είναι σημαντική η περαιτέρω εξέλιξη του κοινωνικού διαλόγου. Ειδικά ε, σε ορισμένε χώρε πρέπει να ξαναχτιστεί ο κοινωνικό διάλογο. Κυρίε και κύριοι, θα ήθελα να τονίσω τρει τομεί πολιτική όπου η δραστηριότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση του επόμενου μήνε θα είναι κρίσιμη, κρίσιμε, ούτω ώστε να υλοποιήσουμε τις κοινωνικέ μας δεσμεύσει. Καταρχάς να κάνουμε πιο πολλά για να εξασφαλίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Αγορά Εργασία δίνει καλές ευκαιρίε στου πολίτε μα Και έχουμε την ε, υψηλή ανεργία. Υπάρχουν δύο εκατομμύρια όμω ε, θέσει απασχόλησης που δεν έχουν ε, καλυφθεί. Α πούμε δεν έχουμε αρκετού προφορικάριους, αρκετού μηχανικού, αρκετού επαγγελματίε υγεία, καθώς και αρκετούς χρηματιστές και λογιστέ. Φυσικά πάντα θα υπάρχουν ε, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή και νέε θέσει απασχόληση, αλλά μπορούμε αυτή την ανισορροπία με την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού να την καλύψουμε και σε τοπικό και σε περιφερειακό και σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να βελτιώσει και να ε, εξυγχρονίσει τι δυνατότητε ε, του Ευρωπαϊκού Δικτύου Γιούρε που δίνει υπηρεσίε απασχόληση, ούτω ώστε να μα δίνει σε πραγματικό χρόνο μια εικόνα για, τις, ε, για το που βρίσκονται και νέες θέσεις απασχόλησης. Ε, το γύρος θα γίνει με, τις, ε, με τη μεταρρύθμιση που προτείνουμε πιο αποτελεσματικό και θα δώσει δυνατότητα στα κράτη-μέλη να δίνουν υπηρεσίες πιο ευέλικτες ανάλογα με τις ε, βασικές ανάγκες της αγοράς εργασίας. Μια καλά λειτουργούσα εύρυθμη ε, αγορά εργασίας μπορεί να βελτιώσει την παραγωγικότητα και τις οικονομικές επιδόσεις, εξασφαλίζοντας ότι ο κόσμος κινείται γρήγορα και βρίσκει την επόμενη δουλειά, αν χρειαστεί, από την εκπαίδευση στη δουλειά πολύ πιο γρήγορα και από την ανεργία στη δουλειά πάλι πιο γρήγορα. Αλλά πρέπει να κάνουμε πολύ περισσότερα για να βελτιώσουμε την, ε, τις επιδόσεις του δημοσίου τομέα και την, την αποτελεσματικότητα των πολιτικών απασχόλησης. Αυτή η περίοδος είναι πολύ σημαντική, θέλω να το τονίσω αυτό. Είναι μια περίοδος όπου θα αποφασιστούν πάρα πολλά για το μέλλον των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε επίπεδο ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και η χρήση τους μέσα στα κράτη-μέλη ε, στις συζητήσεις για το πολιτές νομικό πλαίσιο θα πρέπει να εξασφαλίσουμε το μέλλον και την ε, επαρκή χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου αλλά και της Ευρωπαϊκής ε, Πρωτοβουλίας για την ε, νεολαία το... καθώς και το ευρωπαϊκό Ταμείου για τους πιο και διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία. Αυτά είναι σημαντικοί πόροι για να βελτιώσουμε τη λειτουργία της ε, ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας, να ενισχύσουμε το ανθρώπινο δυναμικό και να κρατήσουμε την κοινωνική συνοχή. Αν ε, εφαρμόσουμε τις σωστές ε, κοινωνικές πολιτικές, σημαίνει ότι επενδύουμε στο ανθρώπινο κεφάλαιο και στην κοινωνική συνοχή. Αυτές είναι προϋποθέσεις για την ανταγωνιστικότητα και την οικονομική ανάπτυξη στην παγκόσμια αγορά του 21ου αιώνα. Και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο παίζει ένα σημαντικό ρόλο κυρίε και κύριοι, μια εύρυθμη αγορά εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση σημαίνει δίκαιε συνθήκες εργασίας, προστασία βεβαίω και ασφαλεία και υγεία στο χώρο εργασίας. Αυτό είναι άλλο στοιχείο του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Μοντέλου φυσικά και σημαντικό μέλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα. Καλή υγεία και ασφάλεια στην ε, δουλειά σήμερα ε, καταπολεμά την, ε, τον αποκλεισμό, προωθεί την επανένταξη στην αγορά εργασία, στην απασχολησιμότητα και μειώνει την πρόορη ταξιδότηση. Σε αυτή την οικονομική κρίση, το να βελτιώσουμε την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία θα συνεισφέρει αποτελεσματικά στην, στους στόχους της Ευρώπης 2020. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Ασφάλεια και την Υγεία στον χώρο εργασίας μας έπεισε ότι η αποτελεσματική διαχείριση αυτών των στοιχείων ε, είναι και οικονομικό επιχείρημα, είναι οικονομικό κίνητρο για την επιχείρηση. Ένα ασφαλέ ε, πλαίσιο δουλειά, όπου κινητοποιούνται και οι εργαζόμενοι και οι εργοδότε, όπου παράγουν και εργάζονται πιο αποτελεσματικά, φυσικά προωθεί και την ανταγωνιστικότητα τη Ευρώπη. Βοηθάει σε αυτήν. Ε, πέρα από την ασφάλεια και την υγεία, θα πρέπει να εγγύψουμε και σε άλλε πρωτοβουλίε για να βελτιώσουμε ένα πλαίσιο ποιότητας πρώτα απ' όλα για την κατάρτιση των νέων κυρίως, αλλά και ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την αδήλωτη εργασία είναι δύο πολύ σημαντικά εργαλεία. Κυρίες και κύριοι, σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα η Ευρωζώνη αντιμετωπίζουν μια οικονομική κρίση, κοινωνική κρίση και κρίση απασχόλησης. Η κατάσταση βέβαια διαφέρει από χώρα σε χώρα και έτσι η πόλωση ενισχύεται μεταξύ των κοινωνιών. Οι τάσεις αυτές έρχονται σε αντίφαση με τον στόχο μας για πλήρη απασχόληση που με την κοινωνική πρόοδο, το είπα ήδη, είναι από τους στόχους που αναφέρονται στις ίδιες τις συνθήκες. Δεν είναι μόνο στόχοι πρέπει να βρίσκονται και στην καρδιά της εκπόνησης οικονομικής πολιτικής και του σχεδιασμού της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Το ίδιο άρθρο στη συνθήκη λέει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προωθεί την οικονομική, την κοινωνική και την εδαφική συνοχή και αλληλεγγύη. Αυτό σημαίνει ότι από όλες τις κοινωνικές ομάδες και όχι μόνο η ελίτ πρέπει να χαίρουν τη αρρωγής αυτής και να υποστηρίζονται από τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι οικονομίες των χωρών μελών είναι αλληλεξαρτούμενες ημέν από τις ΔΕ. Σε μερικές χώρες η κατάσταση είναι ιδιαίτερα σοβαρή, ιδιαίτερα μέσα στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Η η Νομισματική Ένωση δεν κατάφερε να αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα. Δεν κατάφερε να αντιληφθεί τις πραγματικές οικονομικές εξελίξεις και τα ζητήματα όπως είναι η ένδια, οι ανισότητες, η ανεργία που είναι πολύ βασικά στοιχεία μέσα σε μια οικονομική ένωση. Από το ξέσπασμα της κρίσης διαπιστώνουμε μεγαλύτερο ρήγμα μεταξύ των χωρών που βρίσκονται στο βορρά στο κέντρο της Ευρώπης και εκείνων που βρίσκονται στο νότο της Ευρώπης. Στις πρώτες χώρες αγωνίζονται να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της κρίσης, στην άλλη κατηγορία όμως στο νότο η ανεργία αυξάνεται φόβερα, όπως επίσης και η ένδια. Η πόλωση αυτή είναι ιδιαίτερα αισθητή μέσα στην Ευρωζώνη όπου δεν μπορεί να υπάρξει υποτίμηση νομίσματος πια. Πώς λοιπόν να ανακτηθεί η ανταγωνιστικότητα με εσωτερική υποτίμηση ή με τη μετανάστευση γιατί πολλοί κόσμος φεύγει από τις χώρες του. Οι αρνητικές συνέπειες όλων αυτών στο ανθρώπινο δυναμικό και την κοινωνική συνοχή είναι μεγάλος και από την άλλη μεριά υπάρχει και ο κίνδυνος για λαϊκισμό, για αύξηση των ε, ακραίων θέσεων. Όλα αυτά είναι απόρρια της κρίσης και επιδεινώνονται όσο κρατάει η κρίση περισσότερο. Χρειάζεται λοιπόν ένα δημοσιονομικό σύμφωνο για να βγούμε από αυτή την κατάσταση. Οι ανισορροπίες πλήττουν την Ευρωπαϊκή Είναι λοιπόν τα θέματα τα οποία θα αντιμετωπιστούν με την ανακοίνωσή μας για την κοινωνική δήλωση, για την κοινωνική συνοχή, συγγνώμη, που θα κάνουμε την επόμενη εβδομάδα. Η ο, ναι, φυσικά και είναι κάτι πολύ σημαντικό, αλλά πρέπει να φροντίσουμε να υπάρχει οπωσδήποτε κοινωνική συνοχή και ευημερία για τους ανθρώπους η λειτουργία της ΟΝΕ δεν θα πρέπει να έρχεται σε αντίφαση με τους κοινωνικούς στόχους των κρατών μελών. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Thank Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ε, εισήγησή σας, την παρέμβασή σας, για το καλό μήνυμα ότι πολύ σύντομα θα έχουμε αυτή την πρόταση επιτραπέζης και θα μπορέσουμε να συζητήσουμε την κοινωνική διάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης πλέον. Έχω απλά τώρα το έργο να κλείσω, να ολοκληρώσω την εκδήλωσή μας, ε, το σεμινάριό μας, με πολλές ευχαριστίες προς τον κύριο Επίτροπο προς τον αναπληρωτή Πρωθυπουργό και Υπουργό Οικονομικών της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, ε, κύριο Λάζαρ, θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τους διευθυντές των οργάνων και ε, ιδρυμάτων, τον κύριο Λέτμαερ, τον κύριο Μενέντες Βαντές ε, Σέντλατσέκ και την κυρία Σερβάν, Σερμπάν, Σερμπάν και τα μέλη του πάνελ που συμμετείχαν. Τέλος εξίσου σημαντικό, θα ήθελα να προσθέσω και εγώ μια θετική αγγελία, προαναγγελία ότι έχουμε μια μικρή δεξίωση εδώ μπροστά στην αίθουσα που σας περιμένει να συμμετάσχετε. Ευχαριστώ πολύ. Λίγη συνεδρίασή μας. Ευχαριστώ.